Καλησπέρα και καλώς ήρθατε. Θα ξεκινήσουμε με τα διαδικαστικά στην αρχή. Πρώτα απ' όλα έχετε μπροστά σας την ημερήσια διάταξη. Αν δεν υπάρχουν άλλες προτάσεις, μπορούμε να εγκρίνουμε την ημερήσια διάταξη. Σύμφωνοι. Ωραία, ευχαριστώ. Στη συνέχεια έχουμε ανακοινώσεις της Πρόεδρου και έχω κάποια καλά νέα να σας πω. Ήταν μια μεγάλη απόφαση αυτή που πήρε η Επιτροπή για τα βραβεία Νόμπελ που έδωσε τα βραβεία Νόμπελ σε τρεις γυναίκες οι οποίες δουλεύουν κάτω από πολύ δύσκολες συνθήκες είτε σε χώρους όπου υπάρχουν συγκρούσεις η Έλεν Τζονσέλεν πρώτα απ' όλα, η Έλκα Μπομποβέ επίσης από τη Λιβερία και η κυρία κακάρμαν επίσης. Για την Λιβερία πρέπει να σας πω ότι είναι η μόνη γυναίκα που είναι επικεφαλής ε, Αφρικανικού κράτους. Γυναίκα. Το ότι πήρανε λοιπόν το βραβείο αυτό γυναίκες και από την κοινωνία των πολιτών που οργάνωσαν τόσο καλά τις διαμαρτυρίες που ανάγκασαν ακόμα και τον Τέιλορ να εγκαταλείψει την εξουσία είναι εξωσημείωτο. Μου θυμίζει αυτό επίσης ότι εμείς στην ε, Υποπετροπή μας για τα ανθρώπινα δικαιώματα δύο φορές ασχοληθήκαμε με την Λιβερία και με την ε, Δημοκρατία του Κονγκό, το Κιβού και ασχοληθήκαμε με την τραγική κατάσταση που επικρατεί εκεί και που έχει να αντιμετωπίσει εκεί η κοινωνία των πολιτών στην ε, Λιβερία. Ε, περίπου 70% του θηλυκού πληθυσμού έχει βρεθεί θύμα βιωτήτων, σεξουαλικών βιωτήτων. Και η Ταπακούλ από την Ιεμένη, που είναι η τρίτη, είναι η γυναίκα η οποία οργάνωσε τις μουσουλμάνες γυναίκες δραστηριοποιήθηκε στα ανθρώπινα δικαιώματα και δημιούργησε μια οργάνωση η οποία ονομάζεται Γυναίκες Δημοσιογράφοι Χωρίς Αλυσίδες. Από τον Ιανουάριο που μας πέρασε κινητοποιεί την κοινωνία των πολιτών με διαμαρτυρίες. Ελπίζουμε ειλικρινά ότι το βραβείο αυτό θα τις βοηθήσει να συνεχίσουν το έργο τους. Τώρα όσον αφορά το Αζερμπαϊτζάν. Μου είπαν ότι ο Όμπουτσμαν από το Αζερβαϊτζάν έχει ήδη έρθει. Σας ενημερώνω λοιπόν λιγάκι τώρα ότι τον Μάιο είχαμε ένα ψήφισμα για το Αζερβαϊτζάν και ο πρόεδρος Μπούζεκ επισκέφθηκε την χώρα. Εμείς πάντα υπογραμμίζαμε την ανάγκη να διασφαλίζονται βασικές ελευθερίες οι οποίες απελούνται συνεχώς στο Αζερβαϊτζάν. Δυστυχώς το είπαμε εμείς αυτό, αλλά η κατάσταση κάθε άλλο παρά έχει βελτιωθεί. Επτά ε, πολιτικοί από την αντιπολίτευση εστάλησαν ε, στις φυλακές μετά από μια ειρηνική διαμαρτυρία που έκαναν τον Απρίλιο. Άρα τώρα είναι 14 αυτοί οι οποίοι που για πολιτικούς λόγους βρίσκονται στην φυλακή. Εμείς στηρίζουμε την έκκληση της ε, Λέιντις Άστον και του Γενικού Γραμματέα του Συμβουλίου της Ευρώπης που καταδικάζουν την καταστολή αυτή. Για την ε, Κίνα τώρα. Εδώ θέλω να επιστήσω την προσοχή σας και πάλι στην ε, κατάσταση που επικρατεί όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα του Γκάο Τζισέγκ, ο οποίος είναι αγνούμενος από τον Απρίλιο του 2010. Εμείς στείλαμε διάφορες επιστολές στον πρόεδρο Πούτσεκ που και αυτός με τη σειρά του έθεσε το θέμα στις συνομιλίες που είχε με τον Κινέζο πρέσβη. Δεν έχουν συμβεί όμως και πολλά από τότε. Το Σεπτέμβριο ακούσαμε ε, μια έκθεση από την γυναίκα του, την Χι, η οποία ε, μίλησε μετά από μια συνάντηση στα Ηνωμένα Έθνη και ανέφερε ε, βασανιστήρια κατά του συζύγου της. Όταν θα έχουμε την επόμενη συζήτησή μας στις 5 Δεκεμβρίου για την Κίνα, τότε θα μάθουμε περισσότερα νέα για το τι συμβαίνει με αυτόν στην ακρόασή μας τότε. Και μια που πρόκειται για έναν αγνοούμενο, θέλουμε να σημειώσουμε εδώ ότι η κινέζικη κυβέρνηση συζητάει μήπως ε, νομιμοποιηθεί κάπως ε, η διαδικασία αυτή που έχει σαν αποτέλεσμα η αστυνομία να μπορεί να φυλακίσει σε ένα μυστικό χώρο και χωρίς καμία ανάκριση κάποιον που θεωρεί ύποπτο. Εμείς αυτό πρέπει να το συζητήσουμε το Δεκέμβριο. Έρχομαι τώρα στην Ουκρανία. Στις 11 Οκτωβρίου το δικαστήριο αποφάσισε να καταδικάσει την τέος πρωθυπουργό Τζούλια Τιμοσέγκο σε επταετή φυλάκιση. Ο πρόεδρος Μπούτσεκ έκανε δήλωση με την οποία εξέφρασε την ανησυχία του ε, για την ε, κατάληξη αυτή, για την ετοιμιγορία αυτή που ε, ίσως έχει πολιτικά κίνητρα. Πριν από λίγο συναντήθηκα με κάποιους από την κοινωνία των πολιτών από την Ουκρανία που μίλησαν για την Τιμοσέκο και είπαν ότι πρέπει να ε, κοιτάξουμε και αυτή την περίπτωση αλλά και τις σχέσεις της Ουκρανίας και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει από τη Ρωσία. Αίγυπτος τώρα. Εδώ συνεχίζεται και αυξάνει η βία μεταξύ ε, της χριστιανικής μειονότητας ε, και των άλλων Αιγυπτίων. Στο Κάιρο είχαμε δύο γεγονότα στις 9 Οκτωβρίου. Ο πρόεδρος ε, Πούτσεκ έκανε μια, ένα ανακοινωθέν ε, τύπου και εμείς στην σύνοδο την επόμενη εβδομάδα στο Στρασβούργο θα το συζητήσουμε αυτό το θέμα. Θα υπάρξει ψήφισμα γι' αυτό. Την Ισία τώρα. Εδώ νομίζω ότι πολλοί από εσά θα πάτε στην την Ισία για να είσαστε παρατηρητές στις εκλογές που θα λάβουν χώρα την Κυριακή. Υπάρχει μια μεγάλη ομάδα παρατηρητών υπό τον κύριο Αλμπερτίνη. Προετοιμάζοντα την αποστολή αυτή, σκεφτήκαμε ότι καλό θα ήταν να είχαμε μια συνάντηση με την ΑΦΕΤ στις 10 Νοεμβρίου, έτσι ώστε να μάθουμε περισσότερα για τις εκλογές. Με τον πρόεδρο Μπούσεκ επίσης συμφωνήσαμε ότι στις 10 Νοεμβρίου θα έρθει στη συνεδρίασή μας για να μας μιλήσει για το τι έχει γίνει όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα κατά τη διάρκεια της Προεδρίας του. Οπότε αυτό το θέμα θα το προσθέσουμε στην ημερήσια διάταξη τότε. Σας υπενθυμίζω επίσης ότι στις 23 Νοεμβρίου και μετά από την πρωτοβουλία του Πρόεδρου Μπούζεκ θα υπάρξει μια τεράστια διάσκεψη εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με πολλά βραβεία Ζαχάροφ και άλλους ε, ανθρώπους που ασχολούνται με τα ανθρώπινα δικαιώματα ή που έχουν τιμηθεί με βραβεία για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Στο Μποζάρ θα γίνει εκεί μια άλλη εκδήλωση. Σας το λέω να το σημειώσετε. Έρχομαι τώρα στο Ιράν. Το Συμβούλιο αποφάσισε την προηγούμενη εβδομάδα για νέες κυρώσεις. Τώρα υπάρχουν 29 Ιρανοί τον οποίο θέλουν να απαγορεύσουν τις θεωρήσεις και να παγώσουν τα περιουσιακά του στοιχεία. Υπάρχει επίσης και η περίπτωση του Γιαγιτακάνη, ο οποίος καταδικάστηκε και προβλέπεται γι' αυτόν η θανατική ποινή. Εμείς γράψαμε στις Ιρανικές αρχές για να σταματήσει αυτή η διαδικασία και ζητούμε και από την ε, Βαρόνη Άστον να κάνει μια δήλωση. Πράγμα το οποίο έκανε. Σύρια. Το Συμβούλιο εδώ ε, χαίρεται για τις προσπάθειες της πολιτικής αντιπολίτευσης στη Συρία και του Εθνικού Συμβουλίου της Συρίας προκειμένου να ε, προωθήσει χωρίς βία δημοκρατικές αξίες. Βέβαια δεν αναγνωρίζεται ακόμα επίσημα το Συμβούλιο αυτό. Δεν υπάρχουν επιπλέον κυρώσεις. Πάντως θα μπορούσαν να ληφθούν νέες κυρώσεις από το Συμβούλιο μέσα στις επόμενες ημέρες ίσως. Όλοι παρακολουθούμε από κοντά τις εξελίξεις εκεί. Λίβανος. Η διακοινοβουλευτική αντιπροσωπεία Ευρωπαϊκή Ένωση Λίβανος στις 12 Οκτωβρίου είχαν διαβουλεύσεις. Προσκάλεσαν και την πρόεδρο της Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για να συζητήσουν την κατάσταση εκεί με διάφορους βουλευτές. Για μένα ήταν πολύ ενδιαφέρον να ακούσω ότι εκείνοι θέτουν πολύ περισσότερα θέματα από αυτά που θέτουμε εμείς. Για παράδειγμα λένε ότι χρειάζονται τη στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να τους βοηθήσει να ξεπεράσει το πρόβλημα των φυλακών όπου έχουν πολύ περισσότερο κόσμο από όσων αντέχουν και ότι τίθεται θέμα επίσης παραβίασης ανθρωπίνων δικαιωμάτων και στα νοικοκυριά στη χώρα. Έπειτα το θέμα των Παλαιστινίων προσφύγων και αυτό είναι κάτι το οποίο μας έθεσαν. Υπάρχει μια καθυστέρηση επίσης όσον αφορά την νομοθεσία για τη βία σε βάρος των γυναικών και επίσης και το θέμα των βομβών διασποράς και αυτό το θέμα μας έθεσαν. Είναι και αυτό ένα ζήτημα το οποίο δημιουργεί πολύ πόνο. Είπαν επίσης ότι έχουν πρόβλημα με την παιδική εργασία και ότι χρειάζονται περισσότερες επιθεωρήσεις από τη διεθνή κοινότητα για να αντιμετωπίσουν το ζήτημα. Εμείς από την πλευρά μας ε, θέσαμε το θέμα της όχλησης των υποστηρικτών ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Λίβανο και το θέμα της στήρησης και του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων γενικώ. Τέλος, θέλω να σας ενημερώσω για το ότι έχω τον Πιλάρ Νοριέγκα από το Μεξικό που είναι δικηγόρος που υποστηρίζει και τον Τίγνα και κάποιον άλλον υποστηρικτή ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ο οποίος ο πρώτος πριν από 10 χρόνια, στις 19 Οκτωβρίου του ε, διώχθηκε. Η, η δικηγόρος έχει ερευνήσει πάρα πολλές περιπτώσεις δολοφονιών, αγροτών, αλλά και αγροτών που έχουν ε, οικολογικές ε, καλλιέργειες. Υποστήριξε λοιπόν και το άτομο εκείνο το οποίο βρήκε το θάνατο πριν από 10 χρόνια, όπως είπαμε. Είπαν ότι πρόκειτο για αυτοκτονία και είπαν επίσης ότι η πολιτική της δουλειά ήταν ε, καρπός ε, μιας παρανοϊκής σκέψης. Τότε είχαμε κάνει κάποια εκστρατεία υπέρ της. Η δικηγόρος της λοιπόν ήρθε και λέει ότι θα ζητήσουν μια ανεξάρτητη έρευνα και ότι πήγαν στο Διαμερικανικό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Είναι πολύ χρήσιμο να μιλήσουμε μαζί της και ελπίζω να τα καταφέρει, να ερευνηθεί περισσότερο η περίπτωση. Αυτές ήταν οι ανακοινώσεις που είχα να σας κάνω. Τώρα, περνάμε στο επόμενο θέμα της ημερήσιας διάταξης που είναι η ακρόαση που έχουμε για τα ανθρώπινα δικαιώματα στην Τουρκία εν ώψη της έκθεσης πρόοδου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Υποθέτω ότι έχουμε εδώ όλους τους εμπειρογνώμονες. Ναι. Σας βλέπω. Καλώς ήρθατε. Η έκθεση προόδου, η αιτήσια για το 2011-12, όσον αφορά την Τουρκία, είναι γενικά θετική. Αναγνωρίζει την πρόοδο που έχει επιτευχθεί όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα και ε, επαναλαμβάνει ότι η διαδικασία αυτή είναι ο καλύτερος τρόπος για την προσέγγιση μας με την Τουρκία. Επίσης, όταν ο Επίτροπος Φίλε παρουσίασε το θέμα αυτό, εξέφρασε την πρόθεσή του να δώσει νέα όθηση στον διάλογο Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας προκειμένου να καταπολεμήσει την μεγάλη απογοήτευση που επικρατεί επειδή καθυστερεί η πρόοδο στι διαπραγματεύσει. Εδώ στην Υποβιτροπή μα αυτή πάντα επικεντρωνόμασταν ιδιαίτερα στην κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Κοιτάμε δηλαδή και τα θετικά, αλλά τι περισσότερε φορέ κοιτάμε τι είναι αυτό το οποίο καθ' άλλο παρά ικανοποιητικό είναι σε μια χώρα. Εδώ λοιπόν υπάρχουν διάφοροι τομεί που δημιουργούν ανησυχία. Η ελευθερία έκφραση, για παράδειγμα, γιατί όπως λέει και στην έκθεση πρόοδου, ενώ έχει υπάρξει σημαντική πρόοδος κατά τα τελευταία 10 χρόνια, παρόλα αυτά πρέπει να γίνουν σημαντικές προσπάθειες για να διασφαλιστούν τα θεμελιώδη δικαιώματα στην πράξη και ιδιαίτερα η ελευθερία έκφρασης. Το νομικό πλαίσιο δεν διασφαλίζει ακόμα επαρκώς την ελευθερία έκφρασης. Πολλές περιπτώσεις υπάρχουν κατά δημοσιογράφων και ο αριθμός των δημοσιογράφων που εξακολουθούν να κρατούνται είναι άλλη μια πηγή ανησυχίας μας. Είναι δηλαδή δημοσιογράφοι οι οποίοι έχουν κάπως πιο επικριτική άποψη για διάφορα θέματα που μπορεί να έχουν να κάνουν με το περιβάλλον, με προγράμματα που γίνονται και από τα οποία πλήττεται το περιβάλλον, ε, αυτοί διώκονται. Επίσης εκφράζει και ανησυχία για τις πολλές περιπτώσεις που είναι σε βάρος μεταφραστών και εκδοτών οι οποίοι μεταφράζουν και εκδίδουν βιβλία τα οποία αλλού κυκλοφορούν ελεύθερα. Μια άλλη πηγή ανησυχία μα είναι ότι σύμφωνα με, την, με τον Επίτροπο για Ανθρώπινα Δικαιωμάτα, τον κύριο Χάμερβερ του Συμβουλίου τη Ευρώπη, τα πρόσφατα χρόνια ε, υπήρξαν από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων πολλέ αρνητικέ αποφάσει σε βάρο τη Τουρκία. Και το θυμάμαι και εγώ ήταν αξιοσημείωτο μερικές φορές η απάντηση που παίρναμε από τις τουρκικές αρχές που λέγανε ότι ναι δέχονται την απόφαση, την ετοιμιγορία και λένε κάθε φορά ότι ναι πρέπει όντως να φροντίσουν να κάνουν κάτι. Τώρα η εξελίξη όσον αφορά τους Κούρδους και ιδιαίτερα οι επιπτώσεις τους πάνω στον ε, πληθυσμό και στο βόρειο Ιράκ ε, ιδιαίτερα είναι κάτι το οποίο μας δημιουργεί ανησυχία. Κάποιοι είπαν από τους ευρωβουλευτές μας ότι σε αυτήν την ακρόαση πρέπει να ακούσουμε και τους εμπειρογνώμονές μας να μας μιλούν για την κατάσταση των Κούρδων εκεί. Όπως επίσης και την κατάσταση των ε, Σύρων προσφύγων. Πάνω από 7.500 πρόσφυγες Σύροι βρίσκονται τώρα στην νοτιοανατολική Τουρκία. Είναι εξωσημείωτο, έχει ανοιχτά σύνορα, έχει καλές ε, σχέσεις με τους γείτονές της, αλλά όταν ε, ερχόντουσαν οι πρόσφυγες από το Ιράν για παράδειγμα, ε, άλλες γείτονες χώρες δεν θέλανε να τους υποδεχτούν. Πρέπει λοιπόν να δούμε τώρα τι συμβαίνει στην Τουρκία. Νομίζω ότι δεν έχουν νόμους που να ανταποκρίνονται σε αυτές τις περιπτώσεις προσφύγων, να αποφεύγονται βασανισμοί κλπ. Αυτή η ανταλλαγή απόψεων που θα έχουμε μεταξύ μα είναι μια ευκαιρία για να συζητήσουμε την τρέχουσα κατάσταση όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα στην Τουρκία, στα πλαίσια μάλιστα τη διεύρυνση. Έχουμε πολύ καλούς εμπειρογνώμονες εδώ μαζί μας. Έχουμε την Αλεξάνδρα Κασγκράνχε, που είναι διευθυντή για την Κροατία, την Τέσσερα Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία τη Μακεδονία, την Τουρκία και την ε, Ισλανδία από την Γενική Διεύθυνση διευρυνση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Έχουμε επίση την Ελένη Φλόρτρο που είναι πρόεδρο τη Αντιπροσωπεία μα για τι σχέσει Ευρωπαϊκή Ένωση Τουρκία και έχουμε και την Έμα Σίνκλερ Βέμπ, που είναι από το Human Rights Watch. Έχουμε επίση την κυρία Σέμπνεμ Κορούρου Φιντσάντσι, που είναι μέλος του Συμβουλίου του Διεθνούς ε, Κέντρου Αποκατάστασης Αποβασανισμούς και πρόεδρος ε, του Ιδρύματος Τροπίνων Δικαιωμάτων της Τουρκίας. Έχουμε καλέσει επίσης και τους μασογράφους χωρίς σύνορα, αλλά δεν μπόρεσε να έρθει. Θέλουμε να συζητήσουμε για την ελευθερία τύπου. Λοιπόν, θα δώσω το λόγο ευθύ αμέσω στην Αλεξάνδρα Κασγκράνχε, και μου υποθύμησαν ότι πρέπει να επικεντρωθούμε στα κύρια σημεία μας και ότι έχετε στη διάθεσή σας πέντε λεπτά ο καθένας. Παρακαλώ. Θα προσπαθήσουμε να το κάνουμε αυτό. Να ξεκινήσω λοιπόν ε, πολύ γρήγορα και να σας πω αξιότιμα μέλη στα καθημάς. Τον περασμένο μήνα σας έδωσα μία βασική εικόνα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Τουρκία και φτάσαμε, εξετάζαμε το διάστημα το 1998 μέχρι το 2010. Αυτή τη φορά δεν θα είμαι τόσο αναλυτική, θα είμαι πιο επικεντρωμένη στις βασικές πρόσφατες εξελίξεις που είχαμε φέτος. Ε, βλέπετε τι διαπιστώσεις είχαμε ε, στην έκθεση προόδου που ε, δημοσιεύθηκε μόλις τώρα. Είχαμε θετικές εξελίξεις και να επικεντρωθούμε σε αυτές καταρχάς. Θα ξεκινήσω με τις εξελίξεις σε συνταγματικό επίπεδο. Το η κυβέρνηση ξεκίνησε την εφαρμογή του πακέτου τροποποίησης του συντάγματος το 2010 στη διάρκεια του προηγούμενου έτους. Είχαμε συγκεκριμένες διατάξεις για τα δικαστικά ζητήματα, τη δημιουργία ενός διαμεσολαβητή, την δυνατότητα να υπάρχουν ε, ε, θετικές διακρίσεις υπέρ των γυναικών. Και από όλα αυτά θεωρούμε ότι το πιο βασικό ήταν η, τρο ποποίηση της μεταρρύθμισης του δικαστικού συστήματος. Αυτή η μεταρρύθμιση με την εφαρμογή και την έγκριση της εφαρμογής της νομοθεσίας για την αλλαγή της σύστασης του δικαστηρίου και του συνταγματικού δικαστηρίου μας δίνει ένα πλαίσιο το οποίο δεν υπήρχε στο παρελθόν που μας δίνει τη δυνατότητα για ανεξαρτησία και μεροληψία του δικαστικού συστήματος και αυτό φυσικά συνάδει και με τα ευρωπαϊκά πρότυπα. Αυτές ε, οι αλλαγές αναθεωρήθηκαν από την Αρμόδια Επιτροπή και θεωρήθηκαν ότι είναι συνεπείς με το ευρωπαϊκό δίκαιο. Υπάρχει όμως ανάγκη για ένα νέο σύνταγμα πολιτικής φύσεως για να αντικαταστρήσει το στρατιωτικό σύνταγμα του 1982. Είχαμε δημοψήφισμα ε, το 2010 και εκλογές το 2011 και φυσικά είναι απαραίτητες οι αλλαγές από εκεί και πέρα και προσπαθούμε να δημιουργήσουμε συνένεση και γίνονται συζητήσεις ε, για το Σύνταγμα. Η κυβέρνηση, η κοινωνία των πολιτών ε, έχουν υιοθετήσει αυτό το νέο πρόγραμμα για το Σύνταγμα και ξεκινάει η διαδικασία πλέον. Ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου ε, μίλησε με συνταγματικούς νομικούς ε, για τη σύνταξη του νέου συντάγματος, ε, έδωσε και την έγκριση για την έναρξη ενός δημοσίου ιστότοπου στον οποίο οι πολίτες θα μπορούν να συνεισφέρουν ε, τις απόψεις τους για το νέο σύνταγμα και ζήτησε σε κάθε ένα από τα τέσσερα κόμματα στο Κοινοβούλιο να διορίσουν τρία μέλη για την Συνταγματική Επιτροπή, τη Συντακτική Επιτροπή. Όσον αφορά τώρα τη, ε, το στρατό και τις ένοπλες δυνάμεις, είχαμε κάποιες θετικές εξελίξεις. υπήρχε πολιτικός έλεγχος ο οποίος ενισχύθηκε για τις ε, στρατιωτικές και αμυντικές δαπάνες και έγινε αλλαγή από το στρατιωτικό δικαστήριο, το στρατοδικείο έγινε πλέον πολιτικό δικαστήριο. Επίσης η Τουρκία ε, προσχώρησε στη σύμβαση κατά των βασανισμών, κάτι το οποίο θεωρούμε πολύ θετική εξέλιξη. Όσον αφορά τώρα την ανεξιθρησκεία, η απόφαση να περάσουμε ε, και να επιστρέψουν ε, στην ακίνητη υπηρεσία η οποία κατασχέθηκε στο παρελθόν ε, ήταν πολύ σημαντική και εγκρίθηκε τον Οκτώβριο του 2011. Πέρα από αυτές τις πολύ συγκεκριμένε θετικές εξελίξεις, η πρόοδος όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα και την προστασία των ανηλίκων ήταν πολύ περιορισμένη πέρσι. Πρέπει να γίνουν πολύ περισσότερα, ιδίω για τα θέματα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και εδώ έχουμε και τα αρνητικά στοιχεία που έχουμε στην έκθεση Πρόεδρου που αντικατοπτρίζουν και την κατάσταση της χώρας. Η έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και η διάσκεψη έδωσε ιδιαίτερη σημασία στα ανθρώπινα δικαιώματα σε όλη την ε, Τουρκία και θεωρείται ότι το νομικό πλαίσιο δεν ε, αντικατοπτρίζει τα ευρωπαϊκά πρότυπα, δεν ε, συνάδουν τα όσα γίνονται στα ανθρώπινα δικαιώματα με την ομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Είναι πολύ ανοιχτές οι δυνατότητες ερμηνείας από το δικαστικό σώμα και θα πρέπει να γίνουν αλλαγές για τον αντιτρομοκρατικό νόμο και το ποινικό δίκαιο εν γέννη. Υπάρχουν πάρα πολλές ε, υποθέσεις ε, κατά δημοσιογράφων, συγγραφέων ε, και ανθρώπους οι οποίοι εκφράζουν ελεύθερα την απόψή τους και αυτό φυσικά έχει δημιουργήσει μεγάλες ανησυχίες και για την κατάσταση της ελευθερίας των μέσων μαζικής ενημέρωσης και φυσικά υπάρχουν και απαγορεύσεις για αρκετές ιστοτόπους ε, που δημιουργούν ε, ανησυχίες, απαγορεύσεις και λογοκρισία. Η κατάσταση τώρα στην νοτιοανατολική Τουρκία ε, είναι πολύ σοβαρή. Έχουμε παραβιάσει ανθρωπίνων δικαιωμάτων και συνδέονται και με τρομοκρατικές δραστηριότητες. Θα πρέπει η χώρα να συνεχίσει τα θαραλέα βήματα που πήρε στο παρελθόν και τα θέματα προστασίας ανθρώπων που προασπίζονται τα ανθρώπινα δικαιώματα μα δημιουργούν πολύ σημαντικέ ανησυχίε. Τώρα, για τα δικαιώματα των γυναιτών και την ισότητα των φύλων, δεν έχει ακόμα εφαρμοστεί νομοθεσία ε, σε όλη τη χώρα. η συμμετοχή στην πολιτική ε, κάποιων γυναικών ε, ανέβηκε φέτος. Από το 9 πήγαμε στο 14% στις τελευταίες εκλογές και είχαμε λοιπόν μία μικρή αύξηση στη συμμετοχή των γυναικών στην πολιτική. Από το 9% πήγαμε στο 14%. Αλλά θα πρέπει να υπάρξουν πραγματικές αλλαγές στην παιδεία, ε, τα θέματα των καταναγκαστικών γάμων που είναι σημαντικά εσωτερικά προβλήματα. Επίσης, να σας πω ότι σε γενικές γραμμές η Τουρκία θα πρέπει να συμμορφωθεί πλήρως με τα πολιτικά κριτήρια εν γέννη και τα θεμελιώδη δικαιώματα του ανθρώπου είναι απλώς και μόνο ένα τμήμα αυτών των δικαιωμάτων. Μας ενδιαφέρει το κράτος δικαίου και ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. I like Ολοκληρώνοντας να κάνω μία παρατήρηση για να υπενθυμίσω σε όλους ότι η έκθεση ε, στο κεφάλαιο 13 για τα θεμελιώδη δικαιώματα ε, υπάρχει εδώ και τέσσερα χρόνια αυτή η screening report και φυσικά θα πρέπει να ελέγχουμε τις, την πρόοδο της χώρας ανεξάρτητα από το κατά πόσον και πότε θα ενταχθεί η Τουρκία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θεωρούμε ότι είναι υψίστη σημασία για να γίνει πρόοδος ε, στα θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Τουρκία. Σας ευχαριστώ. Ίσως στην διάρκεια της συζητήσεως μπορείτε να απαντήσετε σε σχόλια και ερωτήσεις που ίσως σας γίνουν. Όσα δεν προλάβατε να πείτε τώρα θα τα πείτε μετά. Ακολουθεί η Ελέν Φλότχ, επικεφαλής της Αντιπροσωπείας για τις σχέσεις με τη Μεγάλη Τουρκική Εθνοσυνέλευση. Σε λίγο πρέπει να φύγω γιατί έχουμε άλλη ψηφοφορία στην ε, Επιτροπή Θεμελιωδών Ελευθεριών για μια γνωμοδότηση και δεν μπορώ να φύγω. Δική μου γνωμοδότηση κιόλας να προβάλλω κάποια επιχειρήματα πιο πολιτικά ας πούμε ώστε να μην ε, υπησέλθω στα όσα θα πούν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή άλλες οργανώσεις για τις προσδοκίες που υπάρχουν σχετικά με τη βελτίωση των ανθρώπινων δικαιωμάτων και της δημοκρατίας. Θυμίζω ότι από πέρσι όπου η Υποεπιτροπή είχε οργανώσει τη σχετική, το σχετικό γεγονό. Νίκησε το ΑΚΠ με μεγάλη διαφορά στις εκλογές με, ψήφου με ψήφους από όλα τα κοινωνικά στρώματα. Το κυρίαρχο κόμμα λοιπόν έχει την απόλυτη πλειοψηφία έστω και αν αν και η πλειοψηφία αυτή μέσα στην Μεγάλη Γενική Εθνοσυνέλευση δεν του επιτρέπει να προχωρήσει σε μεγάλες μεταρρυθμίσεις όπως τις συνταγματικές διότι δεν πέρασε το όριο των 330 εδρών που απαιτούνται. Είναι πολύ αποφασιστική η ατζέντα των ε, πολιτικών μεταρρυθμίσεων στην Τουρκία και εξαρτάται πολύ από την ποιότητα του πολιτικού διαλόγου και την συνένεση που θα μπορέσει να ε, προκύψει από το διάλογο αυτό. Από την άποψη αυτή λοιπόν η εκπόνηση του σχεδίου του νέου συντάγματος ε, με μέσα από μια συντακτική επιτροπή στην οποία θα συμμετέχουν με τρεις εκπροσώπους το κάθε ένα από τα πολιτικά κόμματα. Θα δούμε εάν μόνο οι κοινοβουλευτικές ομάδες ή και κόμματα που δεν μπόρεσαν να ή που πέρασαν το κατόφλι του 1% εν πάση περιπτώσει η Επιτροπή αυτή υποτίθεται ανοιχτή, οι ακροάσεις της δηλαδή είναι ανοιχτές στους ειδικού και στην ε, κοινωνία των πολιτών έτσι σε μια διαδικασία που επιδιώκει την συνένεση που σήμερα είναι απαραίτητη διότι η πόλωση μέσα στην ε, κοινωνία είναι ένα πολύ σημαντικό εμπόδιο για το βάθεμα των δημοκρατικών αλλαγών και βέβαια και για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Βέβαια, οι επιπτώσεις της θέσεως ισχύ του νέου αυτού συντάγματος θα είναι πάρα πολύ σημαντικές και για τη συνέχεια των μεταρρυθμίσεων σε θέματα ανθρώπινων δικαιωμάτων και ιδίως για το κουρδικό. Έχουμε την αίσθηση σήμερα ότι πρόκειται μάλλον για την στρατιωτική ατζέντα η οποία αρχίζει και κυριαρχεί και οι επιθέσεις κατά του ΠΚΚ είναι αυτές που δίνουν τον ρυθμό λίγο πολύ με τον οποίο μπορεί κανείς να μετρήσει την πρόοδο ή θα έλεγα την οπισθοχώρηση της υπόθεσης αυτής. Μέσα στο νέο σύνταγμα, σε ό,τι αφορά την, ε, τον ορισμό της ηθαγένειας, την αποκέντρωση, την ενίσχυση των τοπικών διοικήσεων, των εγγυήσεων, ε, των διαφόρων ελευθεριών, της ανεξαρτησίας της δικαιοσύνης κλπ. Αυτά θα πρέπει να τεθούν μέσα στα πλαίσια της εκπόνησης του νέου συντάγματος, γιατί θα έχουν κέρια σημασία για την κατάσταση και στο νοτιοανατολικό μέρος της χώρας και για το κουρδικό θέμα που θα μπει μέσα σε αυτά τα πλαίσια και που γνωρίζουν όλοι ότι πρέπει να γίνει έτσι. Ε, μπουν δηλαδή στις διαστάσεις τα θέματα αυτά και τις πολιτιστικές, οικονομικές, κοινωνικές έστω και αν εξακολουθεί να δίνεται ακόμα προτεραιότητα σήμερα περισσότερο στα θέματα ασφάλειας. Βέβαια, ο έλεγχος από τις πολιτικές αρχές όπως εξήγησε πριν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι κρίσιμος. Δεν μπορεί κανείς να φανταστεί μια δημοκρατική αποκεντρωμένη Τουρκία μέσα στα πλαίσια ενός συγκεντρωμένου, συγκεντρωτικού μάλλον στρατού που υπαγορεύει, που επιτάσσει στην κοινωνία ε, τις ε, του. Πρέπει να τονιστεί λοιπόν ότι η μισή στρατηγή είναι στις φυλακές διότι είναι ύποπτη ότι προετοίμαζαν πραξικόπημα σε βάρος της κυβέρνησης και για τους στρατηγούς και για τους δημοσιογράφους. Το λυπηρό είναι ότι πολλές από τις δίκες ακόμη δεν έχουν γίνει. Και οι προφυλακίσεις αυτές γίνονται με τρόπο καταχρηστικό. Και νομίζω ότι οι αρχές έχουν συνέστηση των απαραίτητων μεταρρυθμίσεων πρέπει να γίνουν στις δικαστικές διαδικασίες. Δηλαδή όλες αυτές οι επιπτώσεις των μεταρρυθμίσεων που έχουν εγκριθεί από το Σεπτέμβριο πρέπει επιτέλους να μπουν σε ισχύ, να εφαρμοστούν για να ξεπεραστούν τα όσα μπορούν να θέσουν σε κίνδυνο την ίδια την διαδικασία ή τις διαδικασίες δηλαδή ε, σε βάρος των στρατηγών. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι βέβαια τη θέση ρόλο πρωτοπορίας έχουμε αποστείλει Για αυτό το θέμα έχει, υπάρχει και αντιπροσωπεία ειδική ad hoc για να πάει να παρακολουθήσει τις δίκες και ταυτόχρονα να θέσει τις, τα θέματα των απαραίτητων μεταρρυθμίσεων και των άρθρων του ποινικού κώδικα αλλά και του αντιτρομοκρατικού νόμου που έχει απολύτως καταστρεφ, καταστρεπτικές συνέπειες και στους οπαδούς των κομμάτων αλλά και στους δημοσιογράφους διότι αρκεί να μεταφέρει κανείς μια είδηση για μια διαδήλωση για υπέρ των Κούρδων για να βρεθεί στη φυλακή. Πρόκειται για το άθρο 6 του αντιτρομοκρατικού νόμου. Πρέπει επιτέλου να μεταρρυθμιστεί σε βάθο ή η κατάσταση των γυναικών. Το θετικό είναι ότι τώρα η βία σε βαρο των γυναικών αρχίζει και συζητείται δημοσία. Μέχρι πριν από λίγα χρόνια ήταν πραγματικά ταμπού. Εάν μια εφημερίδα τολμούσε, καμία εφημερίδα τολμούσε μάλλον να το θέσει το θέμα, τώρα το κάνουν και πρωτοσέλιδο, επομένω έχει καθαρά ορατότητα το θέμα, αλλά δεν είναι απλώς θέμα ορατότητας, είναι και ο διαρκής χαρακτήρας του προβλήματος της βίας σε βάρος των γυναικών που πρέπει να ε, καταδειχτεί ε, ξεκάθαρα, γιατί η άσκηση βία κατά των γυναικών είναι γενικευμένη. Επίσης, η Ευρωπαϊκή Ένωση κάπως ήδη βάζει τρικλοποδιές στα πόδια στον εαυτό της, διότι δεν χρησιμοποιεί τα πιο σημαντικά εργαλεία, δηλαδή τις διαπραγματεύσεις για τα συγκεκριμένα κεφάλαια, τα δύο κεφάλαια 23 και 24 που είναι ακριβώς ε, δικαιοσύνη και εσωτερικές ε, υποθέσεις έχουν υποστεί κυρώσεις και δεν ανοίγονται. Για το θέμα αυτό τώρα των διαπραγματεύσεων, διότι τώρα έχουμε μπει σε δύο με τρία κεφάλαια που μένουν ακόμη να ανοιχτούν, εγώ τονίζω επίσης την δέσμευση του Επιτρόπου Φιούλε που τονίζει ότι είναι ανάγκη να ανοίξει μια θετική ατζέντα με τις τουρκικές αρχές για να προχωρήσουν σε συνεργασία ώστε στην δοθήσα στιγμή, δηλαδή πότε, όταν θα έχουν αρθεί ορισμένα πολιτικά κολλήματα, να είναι έτοιμοι να μπορέσουν να προχωρήσουν ταχύτερα. Επομένω, η δέσμευση αυτή τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπέρ των ε, διαπραγματεύσεων ή ας πούμε καλύτερα της προπαρασκευής των διαπραγματεύσεων μου φαίνεται πάρα πολύ σημαντική μέσα στο, πολιτικό, ε, στο παρόν πολιτικό πλαίσιο. Δυστυχώς είμαι υποχρεωμένη να αποχωρήσω και ε, θα μου πούν μετά το τι θα συζητήσετε. Ευχαριστούμε πολύ, Ελένη Φλότρο. Και τώρα ερχόμαστε στο Human Rights Watch. I want Έμα Σίνκλερ Βέμπα από το Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Ευχαριστώ πολύ. Ευχόμαστε στα θέματα του δικαστικού τομέα, των ε, δίκαιων δικών και την ελευθερία έκφρασης. Φυσικά και με άλλα πράγματα ασχολούμαστε, αλλά εδώ πέρα θα επικεντρωθώ σε αυτά τα κυριότερα. Το άλλο που μας ενδιαφέρει είναι το θέμα των στρατιωτικών ε, και πώς αυτοί εμπλέκονται στην πολιτική ζωή. Πώς θα προχωρήσουν τώρα στις μεταρρυθμίσεις η Τουρκία. Ελπίζουμε ότι όλες οι πλευρές και η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Τουρκία δηλαδή θα χρησιμοποιήσουν επικοδομητικά τα συμπεράσματα της έκθεσης και θα ξεκινήσουν βήμα-βήμα να δουν πώς μπορεί να προχωρήσει η μεταρρύθμιση του δικαστικού τομέα ώστε να διασφαλιστούν οι δίκαιες δίκες και η ελευθερία έκφρασης. Η έκθεση πρόοδου, δηλαδή, προσφέρει κάποιον τρόπο για να αξιολογηθεί η κατάσταση και για να δούμε τι ακριβώς πρέπει να αλλάξει στον ποινικό κώδικα, για παράδειγμα ο αντιτρομοκρατικός νόμος, προβλήματα που έχουν να κάνουν με τις δίκες δίκες, με τις ιδιαίτερα μακροχρόνιες προφυλακίσεις, θέματα ανακρίσεων, θέματα Ε, που δυσκολεύουν τους ανθρώπους να υποστηρίξουν τους αυτούς τους γιατί το σύστημα δεν τους το επιτρέπει αυτό. Και είναι κάτι το οποίο έχει να κάνει με εκατοντάδες και με χιλιάδες ακόμα ανθρώπους σήμερα. Για να είναι χρήσιμη λοιπόν αυτή η έκθεση πρόοδου ε, πρέπει να την ε, δούνε όλα τα θεσμικά όργανα και η δικιά σας Υποπιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Έχουμε πάντως σημειώσει ότι πολλές χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης σήμερα υπονομεύουν τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να επηρεάσουν τα πράγματα στην Τουρκία. Είναι σαν να τους έχει πάρει η Τουρκία όμοιρους κατά κάποιο τρόπο. Ενώ θέλουν να βοηθήσουν την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Τουρκία. Από την άλλη μεριά, από την πλευρά της Τουρκίας δηλαδή, η Τουρκία επικεντρώνεται πολύ περισσότερο στη δυναμική της πολιτική, αλλά δεν επικεντρώνεται επαρκώς στις εσωτερικές μεταρρυθμίσεις. Είναι θεωρητικό βέβαια να πούμε ότι η Τουρκία έχει ε, Υπουργείο για τα ευρωπαϊκά ζητήματα, οπότε θέλει να υπάρξουν τέτοιες μεταρρυθμίσεις στο εσωτερικό. Κάτι άλλο ανθαρρυντικό είναι το τι γίνεται στο Υπουργείο Δικαιοσύνη, ότι και εκεί υπάρχει μια υπηρεσία η οποία εξετάζει την εφαρμογή των ευρωπαϊκών ε, αποφάσεων, του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου δηλαδή, στην ε, τουρκική πραγματικότητα. Αυτό παντού στην Τουρκία και όσον αφορά την ελευθερία έκφραση και όσον αφορά τις καταχρήσεις που γίνονται πολλές φορές από την αστυνομία, και άλλα θέματα που έχουν να κάνουν με δίκες δίκες, με τις μακροχρόνιες προφυλακίσεις κλπ. κλπ. Πράγματα δηλαδή τα οποία ε, έχει αποφασίσει το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, αλλά η Τουρκία δεν τα εφαρμόζει. Έτσι λοιπόν, αυτό ακριβώς είναι που πρέπει να αλλάξει μέσω από μια αποτελεσματική διαδικασία που θα τροποποιήσει το Σύνταγμα και όπου θα συμμετέχει η ολόκληρη κοινωνία των πολιτών. Βέβαια, προς το παρόν η απειλή για τη διαδικασία αυτή είναι ε, το τι γίνεται με το Κουρδικό Κόμμα για την Ειρήνη και την Ελευθερία που έχει εκλεγμένους, 36 ε, βουλευτές έχουν εκλεγεί, 36 άτομα. Όμως δεν ε, επιτρέπεται και τώρα τα πράγματα βρίσκονται εκτός ελέγχου. Γιατί οι εκατοντάδες έχουν ε, κρατηθεί, βρίσκονται σε προφυλάκηση στις φυλακές και από την Ένωση Κουρδιστάν που υπάρχουν ε, ισχυρισμοί ότι είναι η βασική δομή του ΠΚΚ. Έτσι λοιπόν κατηγορούνται πάρα πολλοί αξιωματούχοι ότι είναι μέλη των οργανώσεων αυτών, του ΠΚΚ για παράδειγμα που θεωρείται ε, τρομοκρατική οργάνωση. Κάτι το οποίο, όπως καταλαβαίνετε, δυσκολεύει πάρα πολύ να, συμμετέχει το, να συμμετέχουν οι άνθρωποι αυτοί που έχουν εκλεγεί στις συζητήσεις για τις μεταρρυθμίσεις. Η κατάσταση και η ατμόσφαιρα είναι αρνητική με διάφορες επιθέσεις που λαμβάνουν χώρα. Θέλω όμως εδώ να πάω λίγο πιο πίσω όσον αφορά το κόμμα αυτό, το PDP των Κούρδων και στο πρόβλημα των ε, νόμων και του νόμου του αντιτρομοκρατικού. Υπάρχει ορισμός της τρομοκρατίας που είναι ιδιαίτερα ευρύς. Έτσι άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν κάνει κάτι το οποίο θα μπορούσε κανείς να ονομάσει τρομοκρατική ενέργεια ή κάποια παράβαση αυτού του τύπου ε, παρόλα αυτά διώκονται. Γι' αυτό και η κυβέρνηση τουρκική θα πρέπει να αλλάξει τον νόμο για να είναι πιο συγκεκριμένος και να μην υπάρχει ένα τέτοιο σύστημα δικαστηρίων που να καταλήγει σε διακρίσεις σε βάρος ορισμένων. Έπειτα υπάρχουν ε, οι αστυνομικές αρχές, ο τρόπος που δρούν. πολλοί ε, αναγκάζονται να περνάνε από δίκες, από διώξεις, χωρίς να υπάρχει συγκεκριμένη επιχειρηματολογία για το αδίκημα για το οποίο διώκονται. Πολύ σύντομα να σας πω ακόμα ότι η έκθεση πρόοδου αναφέρει δύο νόμους και τα άρθρα 6 και 7 του αντιτρομοκρατικού νόμου όπως επίση και το 120 και 314 που αναφέρεται στα μέλη τρομοκρατικών οργανώσεων. Αυτοί οι νόμοι, λέει η έκθεση, πρέπει να τροποποιηθούν. Τέλος για τις γυναίκες και όσον αφορά το νόμο για την προστασία της οικογένειας δεν εφαρμόζεται ικανοποιητικά και δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Οι οδηγίες ε, δεν υπάρχουν για το πώς η αστυνομία πρέπει να προστατεύει τις γυναίκες και την οικογένεια πρέπει να αναθεωρηθεί η νομοθεσία αυτή και εμεί θα παρακολουθούμε από κοντά τις προσπάθειες που θα γίνουν προ αυτή την κατεύθυνση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε την Emma Sinclair Web. Ε, πολύ καλές λεπτομέρειες που μας δώσετε και για το κουρδικό. Η κυρία Σέπν Κόρον Φιρτσάμψη στη συνέχεια. Φιντσάμψη. Ε, σας ευχαριστώ που μου δίνετε τη δυνατότητα να σας πούμε την άποψή μας για την πρόοδο της Τουρκίας. Σας ευχαριστούμε και για την έκθεση πρόοδου, η οποία αναγνωρίζει τις βασικές ε, προβληματικές πτυχές και φυσικά αναφέρει και ποια ε, σημεία χρειάζονται νέες αναθεωρήσεις. Εκτιμούμε τις ε, γενικές μεταρρυθμίσεις στα ανθρώπινα δικαιώματα και τα όσα γίνονται κυρίως για την αναθεώρηση της νομοθεσίας, αλλά φυσικά και την ε, κύρωση του προαιρετικού ε, πρωτοκόλου. Αλλά θα πρέπει να σας πούμε ότι έχουμε κάποια ανησυχία για τους αρχικούς προληπτικούς μηχανισμούς επειδή είναι ανεπαρκής ε, η συνεργασία με την κοινωνία των πολιτών, δεν γνωρίζουμε κατά πόσον είναι ανεξάρτητη αυτή οι μηχανισμοί πρόληψης. Στο τελευταίο σχέδιο κειμένου ε, για αυτό το μηχανισμό πρόληψης ε, μας δημιουργούνται σημαντικές ανησυχίες. Έχουμε και κάποιες ανησυχίες για τον τρόπο με τον οποίο η ανακοίνωση ε, μηδενικής ανοχής για τους βασανισμούς δεν έχει υλοποιηθεί τα τελευταία τέσσερα χρόνια. Έχουμε πολλά περιστατικά βασανισμών και η έλλειψη νομοθεσίας επί του θέματος είναι ο βασικός λόγος για τον οποίο συνεχίζονται οι βασανισμοί. Να σας δώσω κάποια στοιχεία. Είχαμε 363 αιτήσει το 2010 και τους τελευταίους 9 μήνες του 2011 έχουμε 419 αιτήσει. Κατανοείτε λοιπόν ότι δεν έχουμε βέβαια και όλες τις αιτήσει, γιατί δεν έχουν κάνει αίτηση όλα τα θύματα βασανισμών για αποκατάσταση. Βάσει των στοιχείων που έχουμε, οι ισχυρισμοί βασανισμών είναι 717 στους τελευταίους ε, 21 ε, μήνες και εξακολουθούν να γίνονται βασανισμοί και σε τρόπου, χώρους ανεπίσημης κράτησης, ακόμα και σε αστυνομικά οχήματα ε, στους δρόμους ή εκτός από ε, στην, στον πράβλιο χώρο αστυνομικών τμήματων. Θεωρούμε ότι είναι δυσανάλογη χρήση βίας διότι υπάρχει εσκεμμένη χρήση βίας, ιδίως σε διαδηλώσεις, και θα ήθελα να σας υπενθυμίσω και τις πρόσφατες ε, εκδηλώσεις που είχαμε, όπου δολοφονήθηκε ένας δάσκαλος λόγω υπερβολικής χρήσης ε, αερίου, pepper και πολλές φορές χρησιμοποιούνται επί τούτου ε, τα αέρια πάνω στο σώμα ενώ θα έπρεπε να χρησιμοποιούνται και να εκτοξεύονται με διαφορετικό τρόπο. Υπάρχουν πολλές περιπτώσεις ανθρώπων που δολοφονήθηκαν ε, μέσω αυτών των σπρέι. Μία πιο πρόσφατη περίπτωση είναι ένας ακτιβιστής για την ειρήνη, ο οποίος δολοφονήθηκε πρόσφατα ε, στα σύνορα. Να σας αναφέρω επίσης και κάποια στατιστικά στοιχεία που προέκυψαν από μία πρόσφατη έρευνά μας. Είχαμε 25.000 ε, περιπτώσεις σε ένα χρόνο ε, εξέτασης ε, κατά τη διάρκεια της κράτησης, είτε προ είτε μετά της κράτησης. Και σε αυτές τις ιατρικές εξετάσεις διαπιστώθηκαν τραυματισμοί 1.248 ατόμων ε, εντός αστυνομικών οχημάτων. Ε, αυτός είναι σημαντικός αριθμός, διότι είναι το, 50, το 5% των ανθρώπων που ε, συνελήφθησαν που βρίσκονται τραυματισμένοι θεωρούμε ότι δεν υπάρχουν αποτελεσματικές ανεξάρτητες έρευνες σε κατηγορίες κατά βασανισμών. Οι αστυνομικοί οι οποίοι ε, κρίνονται ένιωχοι για κακομεταχείριση ε, την χάνουν στη συνέχεια ποινών οι οποίες είναι αμελητές σε σχέση με αυτό που έχουν διαπράξει. Ε, πολλές φορές η έρευνα γίνεται βάση του άρθρου 256 που σημαίνει ε, ότι έχουμε υπερβολική χρήση βίας ενώ κανονικά θα έπρεπε να χρησιμοποιούνται τα άρθρα 94 και 95, ε, τα οποία έχουν άμεση σχέση με τους βασανισμούς. Ανεξάρτητα ιατρικά αρχεία βασανισμών δεν υπάρχουν ακόμα και δεν θεωρούνται αποδεικτικά στοιχεία και οι εισαγγελικέ αρχές δέχονται μόνο εκθέσεις από επίσημα ιατρικά ε, ε, κέντρα στην Τουρκία. Μας ικανοποιεί ιδιαίτερα το γεγονός ότι είχαμε εκπαίδευση 450 ε, ανθρώπων, αστυνομικών, δικαστικών ε, και ανθρώπων που ασχολούνται με το χώρο. Συμμετείχαμε σε αυτή την εκπαίδευση και κατάρτιση, αλλά δυστυχώς δεν υπήρξε παρακολούθηση του θέματος, διότι το Υπουργείο Δικαιοσύνης έχει ενστάσεις ε, σε αυτές τις εκθέσεις παρακολούθησης και τις εκθέσεις για τις αποφάσεις που λαμβάνονται σε αυτές τις περιπτώσεις. Εάν είναι να γίνεται λοιπόν εκπαίδευση του ε, αστυνομικού ε, σώματος και του δικαστικού σώματος, ε, θα πρέπει στη συνέχεια να υπάρχει και μια παρακολούθηση και θα πρέπει να προωθηθεί το ζήτημα αυτό στην Τουρκία, ώστε να διαπιστώσουμε ότι όντως έχουν υλοποιηθεί αλλαγές. Υπάρχουν και σοβαρά προβλήματα ε, για ανταπαντήσει σε μηνύσεις ή κατηγορίες για να εκφοβιστούν τα άτομα τα οποία έχουν καταθέσει αγωγές. Χρησιμοποιούνται εν είδη για αυτούς τους ανθρώπους. Το άρθρο 265 για παράδειγμα, βία ή απειλές ε, κατά ε, δημοσίου λειτουργού ε, ή αστυνομικού χρησιμοποιείται πολύ συχνά. Χρησιμοποιείται και το άρθρο που αφορά την αστυνομία και την κακή της φήμη και φυσικά ε, έχουμε βιώσει και από πρώτο χέρι αυτή την ε, μεταχείριση. Ε, έγινε μια εκδήλωση στην οποία μοιράσαμε κάποια φυλάδια, στα οποία φυλάδια απεικονίζονταν θύματα βασανισμών. Και τώρα εμείς είμαστε υπόδικοι διότι δυσφημίσαμε την αστυνομία. αυτά λοιπόν ήθελα να σας παρουσιάσω. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Ευχαριστούμε. Είναι καλό να ξέρουμε ότι υπάρχουν τέτοιες οργανώσεις σαν τη δικιά σας που συνεχίζει τη δουλειά της και ότι καταπολεμάτε τους βασανισμούς είτε είναι οργανωμένοι και συστηματικοί είτε όχι. Είναι πολύ καλό να συνεχίσετε τη δουλειά σας για να αποφεύγουμε τέτοια συμβάντα. Τώρα, ακούσαμε όλους τους ομιλητές μας και έχω εδώ κατάλογο που μιλητώνει. Η κυρία Κόπα είναι πρώτα. Παρακαλώ κυρία Κόπα. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ όλους για τις τόσο ενδιαφέρουσες παρουσιάσεις σας, οι οποίες μας δίνουν μια πολύ καλή εικόνα της κατάστασης ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Τουρκία. Εγώ θα επικεντρωθώ στην κατάσταση των γυναικών στη χώρα. Την προηγούμενη εβδομάδα δημοσιεύτηκαν ε, φωτογραφίες σε εφημερίδα μια γυναίκα που την είχε δει ο άντρας της στο πρώτο σέλιδο, έτσι δημιούργησε αίσθηση και έγινε μεγάλη συζήτηση. Κάποιοι θεώρησαν ότι οι εκδότες θέλουν να εκμεταλλευτούν για οικονομικούς λόγους το γεγονός αυτό, άλλοι πάλι είπαν ότι ήταν για να προβληθεί περισσότερο ένα φαινόμενο το οποίο είναι πολύ συνηθισμένο στην Τουρκία. Στις 12 Οκτωβρίου τώρα καταδικάστηκε ο εκδότη της εφημερίδας αυτής γιατί έκανε μη υπεύθυνη δημοσιογραφία και του ζήτησαν να παραιτηθεί. Εγώ έχω μπερδευτεί εδώ για το θέμα. Η οικογένεια και κάποιες οργανώσεις γυναικών ε, αντέδρασαν ε, σε βάρος της εφημερίδας. Θέλω λοιπόν να σας ρωτήσω, πώς έχει κατάσταση στην Τουρκία όσον αφορά την ενδοοικογενειακή βία. Εμένα με εκπλήσουν στατιστικές που διαβάζω, γιατί από ό,τι φαίνεται πέντε γυναίκες την ημέρα χάνουν τη ζωή τους από κάτι τέτοιο και πάνω από 40% των γυναικών κάποια στιγμή είναι θύματα βίας ε, από τους άντρες τους ή συγγενείς τους. Και δεν είναι πολλές αυτές που καταγγέλουν ε, τέτοια γεγονότα. Η κατάσταση λοιπόν, από ό,τι φαίνεται, έχει τεράστιες διαστάσεις. Είναι μια από τις μεγαλύτερες προκλήσεις που αντιμετωπίζει σήμερα η Τουρκία. Για μένα λοιπόν το θέμα είναι πώς μπορούμε να βοηθήσουμε. Ξέρουμε ότι για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα από την Τουρκία δεν είναι εύκολο θεσμικά γιατί υπάρχουν μόνο 7 ε, καταφύγια, 7 χώρια όπου μπορούν να πάνε οι γυναίκες που είναι θύματα ενδοικογενειακής βίας και έπειτα οι τοπικές αρχές ενθαρρύνουν τις γυναίκες να λύνουν τέτοιου είδους προβλήματα μέσα στην οικογένεια. Άρα, τι χρειάζεται. Καλύτερη ενημέρωση των γυναικών. Επίσης, καλύτερη κατάρτιση των αξιωματούχων, έτσι ώστε να ξέρουν πώς να αντιμετωπίζουν τέτοιες περιπτώσεις και πώς να βοηθούν τα θύματα. Ο Υπουργό Σαχίν προσπαθεί να ε, πάρει κάποια μέτρα ε, περισσότερο όμως έχουν να κάνουν με το πώς θα ελέγχεται η κατάσταση παρά το πώς θα προλαμβάνετε και θα αντιμετωπίζετε η ενδοικογενειακή βία. Θέλω να ξέρω λοιπόν η δικιά σας ε, η αξιολόγηση της νομοθεσίας για την προστασία των γυναικών και των μελών των οικογενειών από την ενδοικογενειακή βία πώς έχει κατά τη γνώμη σας. Σε ποιον απευθύνεται την ερώτησή σας, γενικά σε όλους μάλιστα. Η κυρία Παπαδοπούλου τώρα. Ευχαριστώ πολύ. Θα προσπαθήσω κι εγώ να είμαι σύντομη, γιατί πρέπει να πάω στη Λίμπε κι εγώ για να ψηφίσω. Ζητώ συγγνώμη γι' αυτό. Θα κάνω την ερώτησή μου και μετά κάποιος θα μου μεταφέρει την απάντηση. Συμφωνώ με όλα όσα ακούσαμε από τους ομιλητές και ιδιαίτερα από το γεγονό ότι το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων όσον αφορά την περίπτωση Κύπρος εναντίον Τουρκίας είπε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρόθεσε το θέμα των αγνοούμενων από την Κύπρο. Όπως επίσης και τα δικαιώματα των ε, ε, Κυπρίων οι οποίοι αναγκάστηκαν να φύγουν από τα σπίτια τους 40 ε, χρόνια μετά από την κατοχή. Θέλω λοιπόν σχόλια από τους ομιλητές για αυτά τα θέματα, δηλαδή για τους αγνοούμενους στην Κύπρο, για τα δικαιώματα των ανθρώπων που μετατοπίστηκαν και επιπλέον στην έκθεση Πρόδου αναφέρεται ότι η Τουρκία παραβιάζει τα δικαιώματα των μειονοτήτων μέσα στην Τουρκία. Λέει ότι δεν έχει υπογράψει το, τη σύμβαση πλαίσιο του Συμβουλίου, ε, του Ευρωπαϊκού του Συμβουλίου της Ευρώπης. Οπότε ρωτάω, στην χώρα μου που υπάρχει κατοχή, πώς θα προστατευτούν οι τουρκικές μειονότητες. Δεν είναι ηρωνικό η Τουρκία να μην προστατεύει και να μην υπογράφει τη σύμβαση αυτή για την προστασία των δικών της μειονοτήτων μέσα στην ίδια της τη χώρα, την Τουρκία. Και τι κάνει, ζητάει δύο κράτη στην Κύπρο για να προστατεύσουν εκεί την μειονότητα έπειτα το Συμβούλιο της Ευρώπης ζήτησε να υπάρξει ένα καταφύγιο, ένας χώρος δηλαδή και κάθε 7.700 ανθρώπους που να μπορούν ε, άνθρωποι οι οποίοι κινδυνεύουν από επιθέσεις να μπορούν να πάνε εκεί και να προστατευτούν οι γυναίκες ας πούμε. Ακούσαμε πριν πόσο περιορισμένος είναι ο αριθμός των χώρων αυτών. Είναι δυνατόν να υπάρχουν τόσο λίγοι τέτοιοι χώροι που μπορούν να προσφεύγουν οι γυναίκες που υποφέρουν από ενδικογενειακή βία σε μια χώρα με τόσο κόσμο. Ευχαριστώ. Συγγνώμη, αλλά τώρα πρέπει να φύγω να πω. στη Λίμπη. Την απάντησή σας θα μου τη μεταφέρει κάποιος. Η Πρόεδρος. Βεβαίως η σημερινή συζήτηση μεταδίδεται και από το διαδίκτυο και θα τα βρείτε αυτά και στο διαδίκτυο. Ευχαριστώ πολύ. Όλοι ακούμε φοβερά πράγματα από την ε, Τουρκία και το κόμμα μου, το ΠΒΒ Φιλελεύθερη, επίσης ακούμε πάρα πολλά και επιθυμούμε από το ΠΒΒ, το κόμμα της Ολλανδίας, ε, ακούμε φοβερά πράγματα όσον αφορά την Τουρκία και την θέση της στην Ευρώπη. Η κατάσταση όμως δεν είναι ικανοποιητική και ζητάω από τους συναδέλφους να ξυπνήσουν. Η Τουρκία ουσιαστικά τι κάνει. Κατέχει την Τουρκία, την, συγγνώμη, την Κύπρο, είναι δύναμη κατοχή στην Κύπρο. Αυτό πρέπει να το συνειδητοποιήσουμε όλοι. Και όχι να αφήνουμε την Τουρκία να, την Τουρκία να προχωράει. Όχι, πρέπει να τη σταματήσουμε. Να σταματήσουμε τι διαπραγματεύσει, να σταματήσουμε να δίνουμε χρήματα από του Ευρωπαίου φορολογούμενου στην Τουρκία. Η Τουρκία να βγει και από το ΝΑΤΟ και αυτό καλό θα μου φαινότανε. Νομίζω λοιπόν ότι οι συνάδελφοι πρέπει να το συνειδητοποιήσουν αυτό. Κανένας δεν σηκώνεται να τα πει όλα αυτά. Η Ευρώπη είναι ένας τίγρης χωρίς δόντια. Λοιπόν, ζητάω από τους συναδέλφους, κάντε επιτέλους κάτι. Πιέστε την Τουρκία. Ε, μέσω του εμπορίου. Με κυρώσεις, εμπορικές κυρώσεις. Τίποτα όμω δεν κάνουμε από όλα αυτά. Λοιπόν, ζητώ από του συναδέρφους επίση από την Επιτροπή να είναι πιο αυστηρή απέναντι στην Τουρκία. Ευχαριστώ. Thank Σας ευχαριστώ. Η κυρία Βεργιά. Το να μιλεί κανείς για την κατάσταση στην Τουρκία είναι συχνά δύσκολο. Υπάρχουν πολλές προκαταλήψεις σχετικά με τον με τον τρόπο που γίνεται η συζήτηση για την κατάσταση στην χώρα αυτή. Εγώ προσπαθώ να προβώ σε αντικειμενική ανάλυση της καταστάσεως. Δεν θα ήθελα άλλωστε να επαναληφθούν κάποια ασφάλματα του παρελθόντος όπου προτιμήθηκαν τα καθαρά νομικά κείμενα τα οποία έκρυβαν λίγο την πραγματικότητα Πολλοί συνδικαλιστές, δημοσιογράφοι και γενικότερα οι αντιφρονούντες στην κυβέρνηση, όσοι τολμούν να επικρίνουν τις δίθεν μεταρρυθμίσεις που εφαρμόζονται, διώκονται και δικαστικά αλλά και γενικά ε, υφίσταται ε, καταστολή Τα όσα έχουν συμβεί από τον Ιούνιο απέναντι στην κουρδική αντιπολίτευση εντελώς απαράδεκτα. Εάν η αριθμοί που έχω στη διάθεσή μου είναι ορθοί, βρισκόμαστε στις 1000 με 1300 συλλήψεις εκλεγμένων εκπροσώπων των Κούρδων. Συλλήψεις οι οποίες συνεχίζονται και ε, ε, εκτελούνται ακόμη και τώρα. Ήδη τον μήνα Ιούλιο η Τουρκία επενέβη στρατιωτικά στην κουρδική ζώνη του Ιράκ. Έτσι βρέθηκαν σε διασταυρώμενα πυρά οι Κούρδοι. Του Ιράκ, του Ιράκ, διορθώνω, ε, είχε πει Ιράν κατά λάθος κυρία Βεργέ. Ε, βρέθηκαν λοιπόν ανάμεσα σε διασταυρώμενα πυρά των Ιρανών και των Τούρκων οι Κούρδοι. Δεν ακούσαμε ουδεμία απολύτως καταδίκη αυτής ε, τουρκικής επέμβασης η οποία είχε ως θύματα αμάχους και παιδιά. Εγώ το βρίσκω αυτό απολύτως απαράδεκτο. Το ίδιο απαράδεκτο, αφόρητο μεν, αφόρητο μάλιστα, μου φαίνεται να βλέπω υπουργού ορισμένων χωρών μελών μας να μεταβαίνουν στην Τουρκία για να επενούν την τουρκική κυβέρνηση, να επενούν τη μεταναστευτική πολιτική και στο όνομα ενό αγώνα κατά τη τρομοκρατία ξαναστέλνουν στην Τουρκία ορισμένους ε, Κούρδους οι οποίοι κανονικά θα έχεραν προστασίας εδώ σε ευρωπαϊκό έδαφος. Θα ήθελα λοιπόν να τεθεί το θέμα αυτό της προστασίας της κουρδικής μειονότητα και ε, να επιληφθεί περισσότερο του θέματος αυτού η παρούσα υποεπιτροπή. Διότι ωραία είναι να μιλούμε για θέματα ανθρώπινων δικαιωμάτων, αλλά κάποια στιγμή θα πρέπει να συνάγουμε και τα απαραίτητα συμπεράσματα και να τα εφαρμόζουμε στην πράξη. Μία φράση ακόμη για το θέμα των γυναικών, γιατί τη συνάδελφό μου μίλησε πριν. Διότι πράγματι υπάρχει ένα σοβαρό θέμα για τις γυναίκες. Προσπαθούμε, όπως είπα, να εξετάσουμε τα γεγονότα αντικειμενικά, διότι ακούω όλο και περισσότερα για έναν καλπάζοντα εξισλαμισμό στην Τουρκία και το ΑΚΑΠΕ φαίνεται να, είναι, να παίζει ηγετικό ρόλο σε αυτό. Ευχαριστώ. Thank you very um, κυρία Σάκε. Θα συμφωνήσω και εγώ ότι η διαδικασία εντάξει είναι το καλύτερο εργαλείο και πορεία για την προσέγγιση της Τουρκίας. Χαίρομαι που ο Επίτροπος Φίλε τόνισε στην έκθεση πρόοδου φέτος ιδιαίτερα την ελευθεροτυπία και το κράτος δικαίου. Ήδη όμως οι ε, βουλευτές που μίλησαν προηγουμένως το τόνισαν πόσο σημαντικό αυτό είναι αυτό Επίσης όταν είναι τόσο ταχείες οι μεταρρυθμίσεις είναι σωστό να εξετάζεται εάν η εφαρμογή του νόμου είναι ίσως διαφορετική από το γράμμα του. Συχνά χρειάζεται πολλής χρόνος μέχρι ότου κάποιος βελτιωμένος νόμος να καταλήξει να εφαρμόζεται ε, μέχρι και από τον αστυνομικό ε, που κυκλοφορεί στον δρόμο και πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί γι' αυτό. Το ίδιο πρέπει να δώσουμε ιδιαίτερη σημασία για την ελευθερία του τύπου και τους δημοσιογράφους, ένα θέμα που με απασχολεί εδώ και πολύ καιρό και που θεωρώ ότι είναι, είναι πάρα πολύ σημαντικό και για την Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και για άλλες χώρες. Μεμφθήκαμε την Τουρκία για την έλλειψη ελευθερίας του τύπου και βγήκε η κυβέρνησή τους και είπε ότι οι δημοσιογράφοι δεν φυλακίζονται επειδή ασκούν το δικαίωμά τους της ελεύθερης δημοσιογραφίας, αλλά διότι υποτίθεται ότι είναι μέλη τρομοκρατικών οργανώσεων. Σε ό,τι με αφορά, εγώ θεωρώ ότι αυτό πρέπει ακόμη να αποδειχθεί. Δεν έχει αποδειχθεί. Και όποιο και αν είναι ο λόγο τη σύλληψη τέτοιου μεγάλου αριθμού δημοσιογράφων, πραγματικά παγώνει και τον ίδιο τον τύπο, αλλά και την ευρύτερη κοινωνία και την κοινωνία των πολιτών, για παράδειγμα, καθώ και των πανεπιστημιακό κόσμο. Σε ό,τι αφορά τώρα την υποκλοπή τηλεφώνων, και αυτό ένα θέμα το οποίο πρέπει να μας ε, απασχολήσει, άνθρωποι επίσης οι οποίοι έχουν ε, βρεθεί στη φυλακή και εξακολουθούν να κρατούνται στη φυλακή χωρίς να τους έχουν επαγγελθεί κατηγορίες. Βρίσκω ότι είναι ιδιαίτερα προβληματικό. Εάν δούμε ότι γίνεται κάποια κατάχρηση αντιτρομοκρατικών νόμων, αυτό θα πρέπει να είναι ένα θέμα που θα πρέπει να μας απασχολήσει πάρα πολύ με τον ευρύτερο δυνατό τρόπο απέναντι στην ε, Τουρκία. Ελπίζω γενικότερα η έκθεση προοδού που θα επεξεργαστούμε και στην Επιτροπή Εξωτερικών θα, δώσει ιδιαίτερο, θα ρίξει ιδιαίτερο φως στην γενικότερη εφαρμογή και στην ενίσχυση του νόμου, του κράτους δικαίου την ε, βελτίωση απονομή δικαιοσύνη, τον διαχωρισμό των εξουσιών, διότι η Τουρκία από οικονομική πλευρά κάνει μεγάλη πρόοδο. Εμφανίζεται ω ισχυρότερη δύναμη στην περιοχή τη και νομίζω ότι πρέπει να υπάρξει περισσότερος χώρος για μια κριτική συζήτηση, διότι μπορεί εμείς να έχουμε τι ιδέε μα από την ευρωπαϊκή πλευρά, αλλά θα ήταν πολύ καλύτερα να μπορέσει να γίνει συζήτηση κριτική ε, ε, μέσα στην ίδια την Τουρκία, ιδίω για τι απαιτούμενε συνταγματικέ μεταρρυθμίσει και εκεί η κοινωνία των πολιτών να μπορέσει να, μπορέσει να παίξει τον ρόλο τη. Σε ό,τι αφορά του ε, πρόσφυγε, είναι πολύ σημαντικό. Είναι πολύ σημαντικός ο ρόλος που παίζει η Τουρκία για την υποδοχή προσφύγων από το Ιράν αλλά και από τη Συρία και από αλλού. Ο ύπατος αρμοστής ε, του, για τους ε, πρόσφυγες είναι η οργάνωση αυτή η οποία φροντίζει τους πρόσφυγες αυτούς και τον μισό από τον προϋπολογισμό του υπατορμοστήτων χορηγεί η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ίσως λοιπόν η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να φροντίσει ώστε να υπάρξει καλύτερο συντονισμός και ενδεχομένως και να υπάρξει και ειδική ενίσχυση των τουρκικών αρχών διότι ίσως υπάρχουν και προβλήματα ικανότητας υποδοχής τόσων πολλών ανθρώπων οι οποίοι ε, καταφεύγουν στην Τουρκία διότι κινδυνεύουν από βασανιστήρια ή και από τον θάνατο στις άμεσα γειτονικές χώρες. Πρέπει να εξεταστεί και η ασφάλεια των προσφύγων. Βρίσκουν τα στην Τουρκία, αλλά βλέπουμε επίσης ότι επειδή τα σύνορα προς το Ιράν είναι ανοιχτά επί ένα τρίμηνο και προς την Συρία και υπάρχει ελεύθερη μετακίνηση και είναι και μικρές οι αποστάσεις υπάρχουν και περιπτώσεις ανθρώπων οι οποίοι υφίστανται παρενοχλήσεις μέσα στην Τουρκία όταν πρόσφυγε από το Ιράν ή από τη Συρία. Επίσης ένας υψηλό αξιωματούχος του, του Συριακού στρατού ο οποίος διέφυγε από την Συρία και με κάποιο τρόπο τον απήγαγαν και τον μετέφεραν ξανά στη Συρία και εκεί υπέστη βασανιστήρια. Αυτά λοιπόν είναι περιπτώσεις οι οποίες πρέπει να εξεταστούν και ίσως να είναι απαραίτητο να υποστηρίξουμε την Τουρκία ώστε να αποκτήσει μεγαλύτερη δυνατότητα να διασφαλίζει τα πρόσωπα αυτά. Ε, Λόχ Μπίλερ. Θα δώσω το λόγο τώρα στις τρεις... Α, με συγχωρείτε. Φρίντα, με συγχωρείτε. Φρίντα Μπρέπολς. Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θα είμαι σύντομη. Θα μιλήσω πολύ σύντομα για τα ανθρώπινα δικαιώματα στα πλαίσια της εκθέσεως πρόοδου. Έχω μια συγκεκριμένη ερώτηση προς την εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Διότι η κυρία Σίνκλερ εξήγησε με λεπτομέρεια την κατάσταση των Κούρδων και επί του παρόντος αλλά και τα πρόσφατα χρόνια. Πώς εξελίχθηκε λοιπόν τα τελευταία χρόνια η κατάσταση των Κούρδων και είπε ακόμη η κυρία Σίνκλε Βέμπ ότι καθένας ο οποίος συμμετέχει σε φιλοκουρδικό κόμμα φυλακίζεται, ιδιώκεται. Τα πρόσωπα λοιπόν αυτά βλέπουν να τους στερούν τα δικαιώματά τους. Γι' αυτό είναι σημαντικό να τροποποιηθεί ο νόμος περί ε, κομμάτων, αλλά και ο αντιτρομοκρατικός νόμος. Διαπιστώνω όμως ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάθε χρόνο το απαιτεί αυτό στην έκθεση πρόοδου της ξανά και ξανά και όμως δεν συμβαίνει τίποτα. Γίνεται απολύτως τίποτα. Και διαπιστώνω επίσης ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναγνωρίζει ότι είναι απαραίτητο να υπάρξει πολιτικός διάλογος με τους Κουρδούς που πρέπει να οργανωθεί σωστά και όπου πρέπει να συμμετέχουν όλες οι πλευρές. Διαπιστώνουμε κάθε χρόνο ότι η στάση απέναντι στους Κούρδους κληραίνει και το βλέπουμε και στην έκθεση ότι αναφέρεται πως λείπει η πολιτική βούληση προκειμένου το κουρδικό να προχωρήσει. Και ο καθένας στην Ευρώπη σε υψηλό επίπεδο πιστεύει ότι η λύση θα υπάρξει μόνο εφόσον ξεκινήσει διάλογος. Γι' αυτό θέλω να ρωτήσω λοιπόν την Επιτροπή. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σκοπεύει να κάνει κάτι ώστε να προχωρήσει η κατάσταση και να λυθεί το ζήτημα το κουρδικό γενικά, αντί να αρχίσουμε πάλι από την αρχή να μιλάμε για την ομοθεσία, την προσαρμογή της, την ε, βελτίωση, τη χρήση της γλώσσας. Νομίζω ότι δεν μπορούμε να προχωρήσουμε αλλιώς αν δεν ξεκινήσει διάλογος. Thank you very Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Μπρέπολς. Έχουμε λοιπόν τώρα τις ερωτήσεις βέβαια και δηλώσεις. Το τμήμα των ερωτήσεων που αναφέρεται κυρίως στην κατάσταση των Κούρδων, την βία κατά των γυναικών, και την ελευθερία του τύπου. Βλέπω ότι η κυρία Παπαδοπούλου επανήλθε. Το θέμα λοιπόν των μειονοτήτων επίσης και των αγνωμένων της Κύπρου. Νομίζω ότι η δική σας δήλωση, κύριε Μάρκιν, ήταν περισσότερο δήλωση ε, κομματική. Δεν ήταν τόσο πολύ ερώτηση Προ του εμπειρογνώμονε. Ε, Εσεί θεωρείτε ότι δεν πρέπει να συνεχιστούν οι διαπραγματεύσει, αλλά υπάρχουν διαφορετικέ απόψει. Αυτό ήταν λίγο πολύ ε, δήλωση του κόμματό σα, αλλά νομίζω ότι δεν, δεν την συμμερίζεται η πλειοψηφία ε, των παρευρισκομένων. Τώρα από το Τουρκικό Ίδρυμα Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Αλλά παρακαλώ να είστε σύντομοι στις απαντήσεις σας. Επιθυμώ να απαντήσω για το θέμα της κατάστασης των γυναικών που είναι και η ειδικότητά μου διότι είμαι ιατροδικαστής και ασχολούμαι με την ε, ε οικιακή βία. Είναι σημαντικές οι, ε, οι μεταρρυθμίσεις για, ε, που προβλέπονται τουλάχιστον. Υπάρχουν αυτά τα καταφύγια αλλά δεν υπάρχει επαρκής προστασία διότι μπορούν εύκολα να διεισδύσουν άλλα στοιχεία στα καταφύγια και μπορούν και εκεί να βιάσουν τις γυναίκες ή να τις βγάλουν έξω και να τις σκοτώσουν. Ιδιαίτερα λοιπόν προβληματική είναι η εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων. Βέβαια δεν είναι εύκολα τα πράγματα αυτά, διότι έχουν γίνει τόσες πολλές μεταρρυθμίσεις και σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα, ώστε για να εφαρμοστούν πρέπει να διατηρεί κανείς διαρκώς την σωστή οπτική και προοπτική. Θα χρειαστεί χρόνο. Τώρα για τον εξισλαμισμό. Δεν έχει σχέση με τα δικαιώματα των γυναικών στην Τουρκία. Αντιθέτως, υπήρχε διάκριση σε βάρος των μουσουλμάνων γυναικών που φορούσαν τις μαντήλες. Τώρα μπορούν να έχουν τα ε, εκπαιδευτικά τους δικαιώματα, για παράδειγμα. Αντιθέτως όμως, βελτιώνονται το σε Εκείνη η μόνη βελτίωση που, η κυρία μάλλον βελτίωση που μπορώ να σα επισημάνω, τα δικαιώματα των γυναικών. Για την ελευθερία της έκφρασης το πρόβλημα είναι όντως σοβαρό. 63 δημοσιογράφοι βρίσκονται τώρα στις φυλακές. Και παρόλο που οι αρχές ισχυρίζονται ότι δεν τους έχουν βάλει στη φυλακή επειδή εξέφρασαν απόψεις, Παρ' όλα αυτά αυτός είναι ο λόγος. Μπήκαν δηλαδή στη φυλακή διότι εξέδωσαν προσωρινά βιβλία. Νομίζω ότι θα αρκεστώ σε αυτά και αν με επιτρέπετε να επιστρέψω το λόγο στις συναδέλφους μου. Για, το θέμα της ε, ενδοοικογενειακής βίας θα ήθελα να πω και εγώ κάποια πράγματα. Όπως σας έλεγα, υπάρχει συνεχής δέσμευση από τον νέο Υπουργό Οικογένειας και Κοινωνικών Πολιτικών. Είναι η Υπουργός ε, η αρμόδια για να αλλάξει και το νόμο για την προστασία του οικογενειακού βίου και να υπάρχουν εντάλματα προστασίας για γυναίκες οι οποίες είναι θύματα οικογενειακής βίας και θέλουν να περιλαμβάνει και ένα ευρύτερο τμήμα του πληθυσμού. Προ το παρόν υπάρχουν πάρα πολλοί περιορισμοί στο νόμο αυτό τη προστασία τη οικογένεια. Ε, προστατεύει μόνο κόσμο ε, που είναι νομίμως ε, ή παντρεμένοι άνθρωποι που έχουν συνάψει πολιτικό γάμο. Ανθρώπου που συμβιώνουν ή που δεν συμβιώνουν με τον σύντροφό του ή έχουν παντρευτεί με θρησκευτικό γάμο δεν προστατεύονται από την νομοθεσία αυτή. Υπάρχουν πάρα πολλέ ομάδε που δραστηριοποιούνται ενεργά για το θέμα αυτό και συναντήθηκαν πρόσφατα και με την Υπουργό. Θα ήταν πολύ σημαντικό λοιπόν να παρακολουθήσουμε τη διαδικασία, να δούμε τη σχετική πρόοδο και να δούμε και πώς θα εφαρμοστεί. Αυτή τη στιγμή αλλάξει ο νόμος. Ε, εάν αλλάξει να δούμε και πώς θα εφαρμόζεται και αν θα είναι και πιο αποτελεσματικός. Δεν έχω δει το σχέδιο κειμόνου που αναφέρεται για την προστασία των γυναικών και της οικογένειας ε, κατά της βίας. Αναφέρθηκε στον τύπο πρόσφατα την περασμένη εβδομάδα, αλλά ακόμα δεν έχουμε δει το σχέδιο κειμένου, επομένως δεν μπορώ να σας πω τίποτα γι' αυτό αλλά νομίζω ότι αυτή της μορφής ε, η νομοθεσία είναι αυτό που θα θέλαμε να υλοποιηθεί στο μέλλον. Όσον αφορά το γεγονός ότι η Τουρκία δεν ε, ε, τηρεί τα διεθνή πρότυπα και δεν υπογράφει διεθνεί συμβάσεις όπως το πλαίσιο για τις εθνικές μειονότητες, εμείς ως Human Rights Watch έχουμε εκφράσει ανησυχίες για το γεγονός ότι η Τουρκία ακόμα δεν ε, εφαρμόζει διεθνείς συμβάσεις για την προστασία των μειονοτήτων και χρησιμοποιεί ε, έναν παλιό ορισμό των μειονοτήτων από τη συνθήκη της Λοζάνης. Είναι κάτι λοιπόν το οποίο είναι γνωστό, έχει ε, αναφερθεί επανειλημμένως και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις εκθέσεις προόδου της εδώ και αρκετά χρόνια. Να δώσω το λόγο στους συναδέλφους τώρα. Ευχαριστώ πολύ. Τα είπαμε όλα, αλλά δεν τα είπαμε και όλα. Συμφωνούμε, αναφέρατε κάποια στοιχεία τα οποία δεν είναι καθόλου αποτελεσματικά για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Τους τα έχουμε επισημάνει και στην έκθεση πρόοδου και συμφωνούμε απόλυτα γι' αυτό. Έχουν γίνει ή δεν έχουν γίνει αλλαγές στην Τουρκία. Νομίζω ότι είναι προφανές ότι έχουν γίνει αλλαγές σε θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ε, αν διαβάζετε και τις εκθέσεις πρόοδου που κάνουμε κάθε χρόνο, γίνεται συγκριτική μελέτη και διαπιστώνεται ότι υπάρχει πρόοδος. Η πρόοδος όμως δεν είναι επαρκής. Το κατά πόσον κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αυτό που πρέπει, εμείς έχουμε κάνει όλο και περισσότερα, προσπαθούμε να επισημάνουμε ποιοι είναι οι προβληματικοί τομέ και η αξιολόγηση ομολόγων που ε, εμπειρογνώμονες από τα κράτη-μέλη πηγαίνουν στην Τουρκία και μελετούν την ομοθεσία εις και βλέπουν πού συγκεκριμένα κάποιος νόμος δημιουργεί προβλήματα γίνεται ολοένα και περισσότερο. Ε, Και επειδή ακριβώς γίνεται αυτό, μπορούμε να σας πούμε ότι το τάδε άρθρο παραβιάζει τα ανθρώπινα δικαιώματα. Έτσι έχει γίνει έλεγχος όλων των άρθρων του αντιτρομοκρατικού νόμου που παραβιάζουν ανθρώπινα δικαιώματα. Όλα αυτά τα έχουν εντοπίσει οι ομολογοί μας και αυτός ο αγώνας δεν θα πρέπει να σταματήσει. Μόνο έτσι μπορεί να γίνει και μόνο με αυτόν τον τρόπο ε, γίνονται αλλαγέ. Είναι πρόθυμοι να κάνουν αλλαγέ στην Τουρκία, αλλά αν δεν πιέζαμε εμεί, δεν θα ήταν η κατάσταση ε, όπω είναι τώρα. Είναι καλύτερη σίγουρα από ό,τι ήταν. Βεβαίω, πόρο απέχουμε από το σημείο που θα θέλαμε να φτάσουμε, αλλά έχουν γίνει αρκετά. Δεν θα πρέπει λοιπόν να σταματήσουμε. Είναι καιρό να συνεχίσουμε και εδώ θα ήθελα να γίνω και λίγο πιο συγκεκριμένη. Για την κατάσταση στην νοτιοανατολική πλευρά τη χώρα επιδεινώνεται, το έχουμε διαπιστώσει, μα ανησυχεί ιδιαίτερα αυτό που συμβαίνει και λέμε στις τουρκικές αρχές ότι δεν μπορούν να έχουν μόνο μία στρατογική για τον Νότο, ε, που να επικεντρώνεται μόνο στην καταπολέμηση της τρομοκρατίας. Θα πρέπει να υπάρχει μια συνολική στρατογική για την νοτιολογική πλευρά της χώρας που θα περιλαμβάνει και τα κοινωνικο-οικονομικά δικαιώματα και τα δικαιώματα των μειονοτήτων και το σεβασμό της γλώσσας και της κουλτούρας ε, του λαού εκεί και να υπάρχει και ένα κατάλληλο ε, νομοθετικό πλαίσιο κατά της τρομοκρατίας. Χρειάζεται λοιπόν μια συγκεκριμένη στρατηγική για την νοτιοανατολική πλευρά της χώρας και η Τουρκία θα πρέπει να το κάνει αυτό, αλλιώς δεν θα έχουμε αποτελέσματα. Για την κατάσταση των γυναικών, σαφώς η κατάσταση βελτιώνεται, αλλά με βήματα χελώνας. Ε, αυτά που αναφέρετε είναι προγράμματα προενταξιακής βοήθειας, ε, πληρώνονται με κονδύλια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, έχουμε αρκετά προγράμματα δεν επαρκούν σε καμία περίπτωση, αλλά είναι μια διαδικασία η οποία δεν έχει ολοκληρωθεί, είναι στην αρχή της. Ε, γίνονται κάποιες πρόοδοι, αλλά ακόμα θα πρέπει να είμαστε εμείς παρόντες για να αλλάξει η νομοθεσία στον τομέα των γυναικών. Δεν έχουμε δει και εμείς τον νόμο, μόλις βγήκε το σχέδιο κειμένου και δεν το έχουμε εξετάσει και θα πρέπει να δούμε τα θέματα εφαρμογής, ε, και τα συνοδευτικά μέτρα. Και τα συνοδευτικά μέτρα είναι αυτά τα οποία θα κάνουμε με την κοινωνία των πολιτών, με μη κυβερνητικέ οργανώσει και με την κυβέρνηση, ώστε να αλλάξουν οι νοοτροπίε. Διότι δεν μιλάμε απλώ και μόνον για αλλαγή και νομοθεσία. διότι αν απλώ άλλαζε ο νόμο, θα ήταν εύκολα τα πράγματα. Εδώ θα πρέπει να αλλάξει η νοοτροπία των συγκεκριμένων λαών. Όσον αφορά τα θέματα των μειονοτήτων, και εδώ όπως σα είπα πόρο απέχουμε από αυτό που επιθυμούμε, ε, δεν υπάρχει νομοθεσία που να διασφαλίζει τα δικαιώματα των μειονοτήτων. Κάποια στιγμή πρέπει να υπάρξει, αλλά ακόμα δεν έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο. Όσον αφορά τώρα την ελευθερία έκφρασης, εκεί είμαστε πολύ σαφείς. Έχουμε εντοπίσει ποια άρθρα πρέπει να αλλάξουν, έχουμε βρει τον ποινικό κώδικα και λέμε ότι είναι τα συγκεκριμένα άρθρα, στον αντιτρομοκρατικό νόμο το, είδο, το ίδιο και στο νόμο για την ελευθεροτυπία το ίδιο. Επίσης, ε, θέλουμε να εφαρμοστούν πολύ καλά οι νόμοι από το δικαστικό το σώμα. Θέλουμε λοιπόν ε, να σταματήσει αυτός ο φαύλος κύκλος όπου ε, ενισχύει ο ένας τον άλλον ε, λόγω νοοτροπίας. Τον τελευταίο μήνα λάβαμε στις Βρυξέλλες και όχι μόνο στις Βρυξέλλες αλλά και στο Λουξεμβούργο και στο Στρασβούργο το Ανώτατο Συμβούλιο Δικαστών και Εισαγγελέων μας επισκέφθηκε και το Συνταγματικό Δικαστήριο και όλοι αυτοί οι άνθρωποι συμμετείχαν και είναι πολύ σημαντικές αυτές οι ανταλλαγές που γίνονται. Βλέπουν ποιες είναι οι ευρωπαϊκές προδιαγραφές και τα πρότυπά μας και ε, ε, πρέπει να τα εφαρμόσουν στη συνέχεια. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα συνεχίσει να κάνει τις αξιολογήσεις ε, και τις εκθέσεις της, συνεχίζει ο διάλογος ε, στα θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων, υποστηρίζουμε μη κυβερνητικές οργανώσεις και την κοινωνία των πολιτών, χρηματοδοτούμε συνεχώς προγράμματα στον τομέα αυτό και δεν θα σταματήσουμε. Και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα ήθελε πραγματικά να μπορέσει ε, να συνεργαστεί στον τομέα του κεφαλαίου 23 ε, ε, το οποίο πρέπει να συζητηθεί με την ε, Τουρκία διότι χρειαζόμαστε κατάλληλο διαπραγματευτικό πλαίσιο για να επιτύχουμε αποτελέσματα. Και κάτι τελευταίο για τους αγνεωμένους να σας παραπέμψω στην έκθεση προόδου. Αυτά είναι τα τελευταία στοιχεία που έχουμε και λέγεται εκεί σαφώς ότι αυτές οι περιπτώσεις εκκρεμούν. Αλλά τις παρακολουθούμε κάθε χρόνο. Ευχαριστώ πολύ all Σας ευχαριστώ όλες και όλους για τις ε, απαντήσεις, πληροφορίες και κρίσεις που εκφράσατε. Δεν θα μπορούσα να προβώ σε σύνοψη, αλλά νομίζω ότι ίσως χρειαστεί να περιμένουμε να δούμε σε λίγους μήνες ή σε ένα έτος πώς θα λειτουργήσει ε, ο νόμος για την πρόληψη των βασανιστήριων. Ίσως χρειάζεται να κάνουμε περισσότερα για την παρακολούθηση των επιμέρους υποθέσεων της ε, ελευθερίας έκφρασης, γιατί υπάρχουν πολλές δίκες που ε, συνεχίζονται. Εκεί που άκουσα ότι δεν υπάρχουν θετικές εξελίξεις είναι η υπόθεση της κουρδικής μειονότητας καθώς και των μελών των κουρδικών κομμάτων. Εκεί χρειάζεται περισσότερη προσοχή εκ μέρους μας σε όλες μας τις συστάσεις, όλες μάλλον οι συστάσεις και όσα είπαμε σήμερα, θα διαβιβαστούν στην Επιτροπή Εξωτερικών και θα δώσουμε ιδιαίτερο βάρος, ε, και, ναι, θα ρίξουμε ιδιαίτερο φως και στην κατάσταση στο Βόρειο Ιράκ σε άλλη ε, συνάντησή μας ε, αργότερα φέτος. Σας ευχαριστώ λοιπόν. Ε, θα προχωρήσουμε τώρα στο επόμενο θέμα μας που είναι ανταλλαγή απόψεων με διαμεσολαβητές από χώρες της ανατολικής γειτονίας και θα ε, δώσουμε ιδιαίτερο βάρος στην συνεργασία. Αναμένω με μεγάλο ενδιαφέρον την ανταλλαγή απόψεων. Ο συνάδελφός μου, Τσίπ, που κύριος Αντρέι Γζιμπ θα αναλάβει τώρα τα ενία της διευθύνσεως ε, της ε, συζητήσεως αυτής. Thank you very much, Madam President. Okay. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Θα συνεχίσω στα πολωνικά. Θα ήθελα να καλωσορίσω θερμά τους προσκεκλημένους μας για το τμήμα αυτό της ε, συνεδρίασης ε, της Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Καταρχάς θα ήθελα να καλωσορίσω θερμά τους διαμεσολαβητές από τις χώρες της Ανατολικής Συνεργασίας και θα ήθελα να καλωσορίσω καταρχάς τις κυρίες. Εδώ στην αίθουσα είναι η κυρία Ελμύρα Σουλεϊμάνοβα, Ομπουτσμαν για τα ανθρώπινα δικαιώματα του Αζερβαϊτζάν. Ε, ήταν προηγουμένως στην αίθουσα, τώρα δεν τη βλέπω. Κατόπιν έχουμε την κυρία Τατιάνα Κονσάρια, ε, αντι διαμεσολαβητής, αναπληρωτής διαμεσολαβητής, ε, ζητώ συγγνώμη αν προφέρω λάθος το όνομά σας. Ε, καλωσορίζω επίσης και την ε, κυρία Ιρένα Λίποβιτς, ε, Επίτροπο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων της Πολωνίας και μία ε, των, ε, εκ των συνεργατών που υλοποίησε αυτό που θα συζητήσουμε σήμερα και επίσης έχουμε και τον ε, εκπρόσωπο της Αρμενίας, τον κύριο ε, Αντρεάισαν και έχουμε και εκπρόσωπο της Μολδαβίας, τον κύριο Ανατόλη Μουντεάνου. Καλωθορίζω επίσης και τον κύριο Ντομινίκ Μποντί, ο οποίος είναι εισαγγελέα στη Γαλλία. Πρόκειται για μια γαλλοπολωνική πρωτοβουλία, την οποία θα συζητήσουμε σήμερα και θα αποτελέσει αντικείμενο συζήτηση σήμερα. Τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι μέρη σε εθνικό επίπεδο, αλλά το Ινστιτούτο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και οι διαμεσολαβητές διαδραματίζουν ουσιαστικό ρόλο. Με το έργο τους συνεισφέρουν σημαντικά στον έλεγχο, στην ε, έρευνα, στην πρόληψη, στις εκστρατείες ευαισθητοποίησης και εδώ έχω κατά νου όλες τις πρωτοβουλίες οι οποίες ξεκινούν ε, για να ε, ξεκινήσει μια νομοθετική διαδικασία σε κάθε χώρα. Ο ρόλος λοιπόν των διαμεσολαβητών είναι η προάσπιση του κράτους δικαίου και η μέρημνα για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Θα πρέπει λοιπόν να ενισχύσουμε το ρόλο των διαμεσολαβητών, αλλά αυτό φυσικά ε, εξαρτάται από πολλούς παράγοντες ε, και από την πρακτική σας και από την εμπειρία σας, ε, το γνωρίζετε πολύ καλύτερα από εμάς. Και ένα σημαντικό στοιχείο είναι να υπάρχει επαρκής πολιτική υποστήριξη. Θα πρέπει να διασφαλίζεται η ανεξαρτησία, η αποτελεσματικότητα. Είναι καλό να υπάρχει μια ισχυρή εντολή και μια καλή συνεργασία όταν είναι αρκετά τα γραφεία τα οποία ασχολούνται με την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και πράγματι πολλές φορές διαπιστώνουμε ότι είναι αρκετοί οργανισμοί που ασχολούνται με το θέμα αυτό. Η διεθνής λοιπόν συνεργασία μπορεί να αποτελέσει σημαντικό εργαλείο για να ενισχύσουμε τα Εθνικά Ιδρύματα Προστασίας ε, των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Το 2009 ο Πολωνός διαμεσολαβητής και ο Γάλλος διαμεσολαβητής ξεκίνησαν ένα πρόγραμμα συνεργασίας μεταξύ των διαμεσολαβητών των χωρών της ανατολικής ε, εταιρικής σχέσης το οποίο πρόγραμμα θα ε, ολοκληρωθεί το 2013. ξεκίνησε το 2009. Ο διαμεσολαβητής το 2009 ήταν ο κύριος Κοχανάουσκι, ο οποίος ε, είναι ένας εκ των θυμάτων της καταστροφής του Σμόλενσκ. Η συνεργασία λοιπόν μεταξύ των διαφόρων ε, ιδρυμάτων των διαφόρων χωρών θέλει να ενισχύσει το ρόλο των γραφείων των διαμεσολαβητών και τον ε, ρόλο των μη κυβερνητικών οργανώσεων ενισχύοντας το κράτος δικαίου. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν να λάβουμε υπόψη και τις πρακτικές πτυχές ε, και ε, για το έργο των διαμεσολαβητών, λαμβάνοντας υπόψη και τα όσα κάνει ο Πολωνός διαμεσολαβητής. Η κυρία Λίποβιτς ε, ανέλαβε τα ημεία, οργανώνονται λοιπόν σεμινάρια, ε, εκστρατείες ενημέρωσης, ανταλλαγές βέλτιστων πρακτικών από ε, το δίκτυο των διαμεσολαβητών και το πρόγραμμα αυτό δεν θέλει να διδάξει τίποτα σε κανέναν. Πρόκειται για ένα πρόγραμμα το οποίο είναι υπέρ της ανταλλαγής πληροφοριών διότι και εμεί στην Πολωνία χρειάστηκε να επιλύσουμε προβλήματα ε, στα θέματα αυτά κατά την ευρωπαϊκή μας πορεία. Τα τελευταία στοιχεία που έχουμε ε, από την έκθεση της κυρίας Δεκάιζερ αναφέρουν τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία και η κυρία Δεκάιζερ αναγνωρίζει ότι ε, είναι πολύ σημαντική και επισημαίνεται επίσης και το πόσο σημαντικός είναι ο συντονισμός σε ευρωπαϊκό επίπεδο για τις δραστηριότητες αυτές. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν να ε, είναι στη διάθεση και των υπολείπων οι καλές πρακτικές. Η σημερινή συζήτηση θα μας επιτρέψει να κάνουμε έναν απολογισμό των ε, τελευταίων δύο ετών, αλλά και να συζητήσουμε και τις ε, μελλοντικές προοπτικές συντονισμού. Καλό είναι να έχουμε και κάποιες συστάσεις για την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης από πλευράς Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προκειμένου να επαληθεύσουμε αν αυτή η συνεργασία ήταν ε, ε, αποδοτική μέχρι τούδε, να δούμε πώς μπορούμε να ενισχύσουμε αυτή τη συνεργασία και πώς μπορούμε να την επεκτείνουμε και σε άλλες χώρες και σε άλλα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα. Με ποιο τρόπο μπορεί να ενισχύσει αυτή τη συνεργασία η Ευρωπαϊκή Ένωση και από πλευράς χρηματοδότησης ε, μα ενδιαφέρει η απάντηση. Ξέρουμε ότι η ανατολική εταιρική σχέση έχει ε, χρηματοδότηση συγκεκριμένη στην Ευρωπαϊκή Ένωση και αυτό μας ενδιαφέρει. Ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων είναι ένα ζήτημα το οποίο αντιμετωπίστηκε προσφάτως, ε, έγινε και μια σχετική έρευνα από ε, έναν εκπρόσωπο της τσεχικής δημοκρατίας και τα αποτελέσματα παρουσιάστηκαν πρόσφατα σε μια συνεδρίαση της υποεπιτροπής μας. Η υποεπιτροπή ζήτησε επίσης και μια μελέτη για το συγκεκριμένο ζήτημα και η μελέτη αυτή διανεμήθηκε, θα παρουσιαστεί από τον καθηγητή Κέντζα, τον οποίο καλωσορίζω επίσης και να σας πω ότι ο καθηγητής ε, διδάσκει ε, στο Πανεπιστήμιο του Πόσναν και στην Πολωνία από τότε που ξεκίνησαν οι ελογές ε, διαστερεοποιήθηκε ιδιαίτερα. Έχει συνεργαστεί και με ε, διεθνείς οργανισμούς, εργάστηκε και στη Γενέβη και ασχολήθηκε και με τα ανθρώπινα δικαιώματα στα Ηνωμένα Έθνη. Έχει λοιπόν ε, ακαδημαϊκή δραστηριότητα και πείρα ε, σημαντική που θα μπορέσει να συνεισφέρει σημαντικά στη σημερινή συζήτηση και τα όσα συνεισέφερε στην εκπόνηση της έκθεσης ήταν ιδιαίτερα σημαντικά. Πριν δώσω λοιπόν τον λόγο στον καθηγητή, θα ήθελα να επενθυμίσω ότι σήμερα στη συγκεκριμένη συνεδρίαση είναι παρόντες και εκπρόσωποι της Επιτροπής Αναφερών. Έχουμε και επίτροπο του Ευρωπαίου Διαμεσολαβικό, διαμεσολαβητή, τον κύριο Όλιβερ Φερχέιντελ, τον οποίο καλωσορίζω. Και δίνω το λόγο στον καθηγητή. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ πολύ για τα θερμά σας λόγια και επιτρέψτε μου να συνεχίσω στα αγγλικά για να σας παρουσιάσω την έκθεσή μου. Κύριε Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αξιότιμοι, αξιότιμοι εκπρόσωποι Ιδρυμάτων για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, κυρίες και κύριοι. Καταρχάς θα ήθελα να ευχαριστήσω το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που με επέλεξε για να ετοιμάσω μία μελέτη για τη συνεργασία των ε, ε, γραφείων των διαμεσολαβητών ε, των χωρών της Ανατολικής Συνεργασίας. Με τιμά η πρόσκληση και επειδή μας πιέζει ο χρόνος, θα ήθελα να περιορίσω την παρέμβασή μου στην παρουσίαση ε, του βασικού προγράμματος, του προσανατολισμού της μελέτης και από εκεί και πέρα να σταθώ στα συμπεράσματα και ε, τις συστάσεις. Ελπίζω από τη σημερινή συζήτηση να ε, προκύψουν προτάσεις και διορθώσεις οι οποίες θα μας δώσουν τη δυνατότητα να βελτιώσουμε και να οριστικοποιήσουμε τη μελέτη. Χρησιμοποιώ πληθυντικό διότι η μελέτη έγινε ε, από εμένα αλλά και από τον συνάδελφό μου τον κύριο Αλτσέσκι. Να δούμε λοιπόν λίγο την παρουσίαση, συντομία. Εδώ έχουμε μία περίληψη της μελέτης. Εξετάσαμε τα διεθνή πρότυπα και την πιστοποίηση, ε, την αναγνώριση των οργανισμών αυτών από τους διεθνείς εταίρους, ε, την κατάσταση ε, των οργανισμών ανθρωπίνων δικαιωμάτων στις χώρες ανατολικής συνεργασίας, την τεχνική συνεργασία, την, το πρόγραμμα αυτό συνεργασίας Γαλλίας-Πολωνίας, τα ενδιάμεσα συμπεράσματα και το σχέδιο συστάσεων. Δεν θα σας παρουσιάσω τα στοιχεία όλα αυτά, αλλά είμαι στη διάθεσή σας για να απαντήσω σε ερωτήσεις, ε, εάν φυσικά γνωρίζω την απάντηση. Περνάμε λοιπόν στο πρώτο σημείο. Τι μορφές Ιδρυμάτων Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων έχουμε στις χώρες της ε, Ανατολικής Συνεργασίας Έχουμε οργανισμούς τύπου Ombudsman μόνο στη Μολδαβία. Έχουμε τέσσερις ε, ε, κοινοβουλευτικούς εκπροσώπους που υποστηρίζονται και από ένα Ίδρυμα Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Τα θέματα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων αναπτύχθηκαν στα πλαίσια των Ηνωμένων Εθνών και βάσει των αρχών ε, του Παρισιού και φυσικά εξετάσαμε και την εντολή και τις εξουσίες αλλά και τις δεξιότητες που απαιτούνται προκειμένου να μπορούν να διεξάγουν καλά τα καθήκοντά τους. Το Συμβούλιο της Ευρώπης αρχικώς ήταν υπέρ ε, των οργανισμών ε, του τύπου του Ombudsman. Μόνο στη δεκαετία του 90 επέκτηνε την υποστήριξή του και στις Επιτροπές Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ως συλλογικά σώματα ε, σε αντιπαράθεση φυσικά με ανεξάρτητους φορείς όπως είναι ο Ombudsman. και καθορίζεται και συγκεκριμένα πρότυπα για τους οργανισμούς αυτούς που ανταποκρίνονται στις αρχές του Παρισιού. γίνεται πιστοποίηση από ένα φορέα ο οποίος ε, αναφέρεται ως ε, Διεθνής ε, Επιτροπή που περιλαμβάνει οργανισμούς από όλο τον κόσμο και έχουμε τρία επίπεδα πιστοποίησης. Το α επίπεδο σημαίνει ότι υπάρχει πλήρη συμμέρφωση με τις αρχές των Παρισίων. Δεύτε, το B, η δεύτερη κατηγορία είναι μερική συμμόρφωση και υπάρχει μια τρίτη κατηγορία στην οποία δεν υπάρχει καμία συμμόρφωση. Μόνο μια χώρα στις χώρες ανατολικής συνεργασίας, ε, η Λευκορωσία, ε, δεν έχει καμία δομή που μπορούμε να πούμε ότι τηρεί τις αρχές των Παρισίων. Τώρα, αν δούμε την κατηγορία Α των Εθνικών Ιδρυμάτων Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, ε, σε αυτή την κατηγορία εμπίπτουν άνθρωποι οι οποίοι ε, έχουν προνόμια βάσει του πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών και συγκεκριμένα δικαιώματα που υπάρχουν στην παρουσίασή μου. Όλες οι διεθνείς οργανώσεις το Συμβούλιο της Ευρώπης, τα Ηνωμένα Έθνη έχουν αναγνωρίσει τη σημασία των ε, οργανισμών ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε εθνικό επίπεδο και υπάρχουν και κάποιες δομές οι οποίες ε, έχουν πολλά κοινά στοιχεία και Ε, δεν υπάρχουν απαντήσεις για το πώς ακριβώς μπορούμε να έχουμε συνεργασία μεταξύ αυτών των οργανισμών. Και σε επίπεδο χώρας Ιδίω μέσω του αναπτυξιακού προγράμματος των Ηνωμένων Εθνών μπορούν να γίνουν κάποια πράγματα περαιτέρω. Αναπτύχθηκε το ίδιο ε, πρόγραμμα ε, από το Συμβούλιο της Ευρώπης. Δεν έχω χρόνο να σας το παρουσιάσω, αλλά βασικός στόχος του Συμβουλίου της Ευρώπης είναι να υπάρξει υποστήριξη για τους εθνικούς ε, μηχανισμούς πρόληψης που καθορίζονται βάσει του πρωτοκόλου για τη Σύμβαση κατά των βασανισμών. Τώρα, στη μελέτη αυτή παρουσιάζουμε επίσης εξετάζουμε και τα Εθνικά Ιδρύματα Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στις χώρες ανατολικής συνεργασίας. Στη μελέτη και στην παρουσίαση έχετε παρουσίαση ε, η οποία αποτελείται από τα εξή τμήματα. Υπάρχει μια γενική παρουσίαση που παρουσιάζει την εντολή, τι εξουσίες, ε, τι ανταλλαγέ και την αξιολόγηση. Η αξιολόγηση βασίζεται σε διάφορα έγγραφα από διεθνεί οργανισμούς που συνεργάζονται με τα συγκεκριμένα ιδρύματα και θα πρέπει να πω επίσης και ε, ότι βασιστήκαμε και στις εκθέσεις από τους συγκεκριμένου τους οργανισμούς. Τα πάντα εξετάζονται ξεχωριστά Τα βλέπετε και εδώ εκτεταμένα και στην παρουσίαση αλλά και στη μελέτη. Και ένας από τους τρόπους με τους οποίους ε, μπορεί να γίνει συνεργασία μεταξύ διεθνών εταίρων αλλά και σε διμερές επίπεδο σε κάποιες περιπτώσεις στις χώρες που συζητάμε είναι τεχνική συνεργασία η οποία ως στόχο έχει ε, να δημιουργήσουμε περαιτέρω δυνατότητες. Όλοι αυτοί οι οργανισμοί επικεντρώνονται ιδιαίτερα στα προγράμματά τους σε συγκεκριμένες πτυχές ε, του έργου των συγκεκριμένων ιδρυμάτων, αλλά φυσικά υπάρχουν και πάρα πολλές επικαλύψεις. Υπήρξαν δύο προγράμματα τα οποία είναι ιδιαίτερη σημασία διότι επικεντρώνονται στα συγκεκριμένα ιδρύματα και εποφελούνται τα ιδρύματα των χωρών αυτών. Έχουμε ένα πρόγραμμα ε, το οποίο είναι ένα κοινό πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Ένωσης Συμβουλίου της Ευρώπης, ένα πρόγραμμα ομολόγων, το οποίο λέγεται peer-to-peer. Το, η πρώτη φάση ήταν για το 2008-2009 και στόχος ήταν να έχουμε ένα ενεργό δίκτυο ε, δομών ανθρωπίνων δικαιωμάτων μη δικαστικών ε, προεκτάσεων και ε, υπάρχει και η δεύτερη φάση του προγράμματος για το 2010-2012 και είναι σε δύο στάδια. Υπάρχει ένα γενικό στάδιο το οποίο αφορά τη συνέχιση της υποστήριξης για τη δημιουργία δυνατοτήτων και δεξιοτήτων για τους οργανισμούς αυτούς και ένα δεύτερο στάδιο το οποίο επικεντρώνεται στην δημιουργία εθνικών προληπτικών μηχανισμών. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει τεκμηρίσει που αναφέρεται στα συγκεκριμένα δρήματα σε πολλαπλές περιπτώσεις, αλλά θα πρέπει να πω ότι σε πολλά από τα μέσα τα οποία θα μπορούν να είναι ιδιαίτερα χρήσιμα ως μέσα για συνδρομή στους εθνικούς αυτούς οργανισμούς, δεν μπορούμε να βρούμε κάποια συγκεκριμένη μνήμα. Ε, πολλές φορές αυτά τα Ιδρύματα Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναφέρονται μεταξύ πολλών ε, ε Ιδρυμάτων οι οποίοι είναι σημαντικοί για τους ε, ε διαδικασίες εκδημοκρατισμού αλλά πολλές φορές δεν υπάρχει καθόλου αναφορά σε αυτούς. Τα θέματα δημοκρατίας και ανθρωπίνων δικαιωμάτων αναφέρουν ε, κάτι για στόχο να δημιουργηθούν ιδρύματα όπου δεν υπάρχουν. Αυτά λοιπόν μπορούμε να πούμε για τα προγράμματα αυτά. Αλλά στα πλαίσια της εφαρμογής των προγραμμάτων αυτών αναπτύχθηκαν μια σειρά από προγράμματα είτε μικρότερης είτε μεγαλύτερης ε, κλίμακας. Ε, υπάρχει και η πολλογαλλική Πρωτοβουλία και ο Πολωνό διαμεσολαβητή ανθρωπίνων δικαιωμάτων θα πει κάτι γι' αυτό, Επομένω δεν χρειάζεται να σταθώ εγώ και πάρα πολύ. Να πω ότι αυτό έρχεται στη συνέχεια του προγράμματο ε, του Πύρ του Συμβουλίου τη Ευρώπη και του προγράμματος Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, το δεύτερο πρόγραμμα λοιπόν το οποίο επικεντρώνεται σε Ιδρύματα Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και εδώ έχουμε το μόνο πρόγραμμα το οποίο αφορά αποκλειστικά και μόνον ε, τα Ιδρύματα αυτά στις χώρες Ανατολικής Συνεργασίας. Να φτάσω τώρα στα συμπεράσματα παρατηρήσεις εν είδη συμπεράσματος. Καταρχώς να σας πω ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα ε, θεωρούνται ως βασικές αρχές όπως ε, διαπιστώνονται σε όλα τα ευρωπαϊκά προγράμματα και τα Ιδρύματα Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ε, νοούνται ως εταίροι Τα δύο που αναφέ, ε, προγράμματα που σας ανέφερα, ε, το peer to -peer και η υπολογαλική συνεργασία, αφορούν συγκεκριμένα τα Ιδρύματα Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ε, αλλά δεν φαίνεται να βασίζονται σε μια αναλυτική στρατηγική για πλήρη ε, εξέταση και βασίζονται σε μια ad hoc βάση και εδώ νομίζω ότι θα πρέπει να υπάρξει περαιτέρω ενίσχυση του θέματος αυτού. Ένα τελευταίο στοιχείο το οποίο θα ήθελα να αναφέρω είναι οι συστάσεις. Εδώ θα σας τα αναφέρω εν συντομία. Τα Ιδρύματα Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στις χώρες Ανατολικής Συνεργασίας έχουν σημαντικό χρόνο και εμπειρία όσον αφορά την εφαρμογή και τις εντολές τους και την ε, διεθνή συνεργασία. Η ανάλυση και τα στοιχεία που έχουμε υποδεικνύουν ότι ε, υπήρξε σημαντική πρόοδος ε, για τη δημιουργία των δυνατοτήτων αυτών των ιδρυμάτων, αλλά η συνεργασία που προσφέρεται ε, είναι ακόμα ζωτική σημασία για να δώσουμε τη δυνατότητα σε αυτά τα Ιδρύματα Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων να λάβουν πλήρω υπόψη του τι δυνατότητέ του και να συμμορφωθούν προ τι αρχέ των Παρισιών. Ε, στο ίδιο συμπέρασμα καταλήγουμε και από τις εκθέσεις που έχουμε από Ιδρύματα Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ε, στις χώρες, όπως για παράδειγμα το Αζερβαϊτζάν και τη Μολδαβία. Για να αναπτυχθεί καταλήλως αυτή η συνεργασία, να λάβουμε, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας τρεις απαιτήσει. Καταρχάς, να ε, μην τη βασίσουμε μόνο στις ανάγκες που θα έχουν αυτή τη στιγμή, αλλά και στο ρόλο που αναμένεται να διαδραματίσουν στο μέλλον για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Να λάβουμε υπόψη τη δυνατότητα απορρόφησης ε, που έχουν οι εταίροι και να διασφαλίσουμε και τη βιωσιμότητα των αποτελεσμάτων. Σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν είναι ζωτική σημασία να υπάρχει μια εταιρική σχέση ε, αυτή που προσφέρεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία θα βασίζεται σε μια πιο στρατηγική προσέγγιση ε, που θα αυξήσει την αυτονομία και την ανεξαρτησία των οργανισμών αυτών βάσει και ε, των αρχών του Παρισίου. Και φυσικά όλα αυτά ε, είναι και ε, στο σχέδιο της Υπηρεσίας Εξωτερικής ε, Δράσης για να αναπτυχθούν στρατηγικές για τα ανθρώπινα δικαιώματα στις χώρες αυτές και η στρατηγική θα πρέπει να οδηγήσει καταρχάς σε μια συνεπή και συνεκτική αναγνώριση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων μέσω συγκεκριμένων προγραμμάτων για τη συνεργασία που αφορούν τις χώρες της Ανατολικής Συνεργασίας και να θεωρούνται βασικοί παράγοντες στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, του κράτους δικαίου και της δημοκρατίας και να διασφαλίσουμε ταυτόχρονα και συνεργασία με άλλους φορείς όπως είναι το Συμβούλιο της Ευρώπης, τα Ηνωμένα Έθνη και το καθεξής. Και επίσης να ακολουθούμε την αρχή της διπλής παρακολούθησης ε, με την υποστήριξη ε, των Ιδρυμάτων αυτών και τη δημιουργία δικτύων ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Θα πρέπει να ενισχύσουμε την αυτονομία των Ιδρυμάτων Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ε, και από πλευράς οργάνωσης ε, και να διασφαλίζουμε την ανεξαρτησία τους ιδίως από την εκτελεστική αρχή. Θα πρέπει επίσης να τους εξοπλίσουμε και με συγκεκριμένες εντολές τις οποίες θα μπορούν να εφαρμόσουν εύκολα και να διατηρούν δεσμούς με την κοινωνία των πολιτών, ιδίως με τις πιο ευάλωτες ε, ε, ομάδες και τους πιο αποκλεισμένους. Και φυσικά όλα αυτά θα πρέπει να τα βασίσουμε και στην εμπειρία την οποία έχουν αποκομίσει μέχρι τούδε, λαμβάνοντας υπόψη και την αξιολόγηση των ε, ε, εγγράφων ενημέρωσης για την εξωτερική πολιτική που αναφέρονται συγκεκριμένα στην ανατολική συνεργασία και λάβουν υπόψη τους και τις συγκεκριμένες πρωτοβουλίες που είναι ήδη εν εξελίξη και τη συγκεκριμένη αξιολόγηση στρατηγικής. Θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή καταρχάς στα προγράμματα που αναπτύσσονται στα πλαίσια της ε, γαλλοπολωνικής συνεργασίας των Ombudsman και να υπάρχει και κατάλληλη χρηματοδότηση για την εφαρμογή Δεύτερον, να υπάρχει συμμετοχή των ε, Ιδρυμάτων αυτών για τα ανθρώπινα δικαιώματα των χωρών της Ανατολικής Συνεργασίας σε όλα τα ευρωπαϊκά προγράμματα, όπως για παράδειγμα το πρόγραμμα Peer-to-Peer που σας ανέφερα προηγουμένως. Παρεπιπτόντως, θα ήταν πολύ σημαντικό, διότι το πρόγραμμα αυτό ολοκληρώνεται του χρόνου, να διασφαλίσουμε ότι θα συνεχιστεί το πρόγραμμα ή θα υπάρξει κάποια παρακολούθηση ώστε να βρούμε κάποιο τρόπο να γεφυρώσουμε αυτές τις δραστηριότητες για να έχουμε βιώσιμα αποτελέσματα. Τέλος, κάτι εξίσου σημαντικό, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μπορεί να πρέπει να συμμετέχει πιο ενεργά στην ε, παρακολούθηση και την αξιολόγηση κατά την εποπτεία της εφαρμογής της στρατηγικής προσέγγισης για τα Ιδρύματα Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στις χώρες Ανατολικής Συνεργασίας. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ίσως θα έπρεπε να συμπεριλάβει αυτό το ζήτημα ως μόνιμο ζήτημα συζήτηση στη διακυβουνοβουλευτική συνεργασία. Αναφέρομαι εδώ στο Euronest πιο συγκεκριμένα και τις Επιτροπές Κοινοβουλευτικής Συνεργασίας που έχουν ιδρυθεί στα πλαίσια της Ανατολικής αυτής συνεργασίας. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ αγαπητοί κύριοι για την παρουσίασή σας. Ιδίω δε για τα συμπεράσματα που παρουσιάσατε που ε, τα βρίσκω ιδιαίτερα ενδιαφέροντα στα πλαίσια της σημερινής μας συζητήσεως. Κυρίε και κύριοι, θα ήθελα να δώσω το λόγο στους προσκεκλημένους μας των χωρών της Ανατολικής Γειτονίας. Δυστυχώς δεν έχουμε πολύ χρόνο. Πέντε λεπτά έχουμε ανά ομιλητή. Δεν είναι κοντά μας βέβαια ο διαμεσολαβητής της Ουκρανίας. Άρα σας πέφτει λίγο περισσότερος χρόνος στον καθένα ή στην καθεμία. Θα προσέξω βέβαια να σας παρακαλέσω να μην υπερβείτε τον χρόνο που σας διαθέτω για την αγόρευση σας. Πρώτα, ο κύριος Καρέν Αντρεασιάν από την Αρμενία. Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, Χαίρομαι για την ευκαιρία συνεργασίας που ε, απηχεί τις προκειμένες προσπάθειες για τις κοινέ αξίες. Σε όλες τις δημοκρατικές χώρες η ανησυχία για τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι κοινή. Ευχαριστώ και πάλι τους διαμεσολαβητές της Πολωνίας και Γαλλίας για την πρωτοβουλία για τη σφυριλάτηση συνεργασίας μεταξύ των θεσμών και χωρών μας. Ο σεβασμό για τα ανθρώπινα δικαιώματα αποτελεί προπόθεση για την ισχύ τη δημοκρατία και του κράτου δικαίου. Χωρί θεμελιώδει ελευθερίε δεν μπορεί να υπάρξει πραγματική ασφάλεια ούτε πραγματική ευημερία και ε, ε, ειρήνη σε μια χώρα. Οι πολιτικέ που ξεκίνησαν το 2009 για την ε, γειτονία βασίζονται σε κοινέ αξίε. Δημοκρατία και ανθρώπινα δικαιώματα, κράτο δικαίου Αρχέ τη ε, οικονομία τη αγοράς και αηφόρο ανάπτυξη. Ω αποτέλεσμα η προστασία των θεμελιδών ελευθεριών και ανθρωπίνων δικαιωμάτων βρίσκονται σε θέση προτεραιότητα στι σχέσει Ευρωπαϊκή Ένωση και Αρμενία και ιδίω στα πλαίσια τη συνεργασία για τη μελλοντική συμφωνία συνδέσεω των δύο πλευρών. Στην Αρμενία θεωρούμε ότι είναι ανεκτήμητη η ε, υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η υποστήριξη που δίνει στον ε, συνήγορο των ανθρώπινων δικαιωμάτων. Ο θεσμός μας παίζει σημαντικό ρόλο στο εθνικό πλαίσιο και αποτελεί σημαντικό εργαλείο για την αντιμετώπιση ε, των παραβιάσεων ανθρώπινων δικαιωμάτων. Παρακολουθούμε τις εξελίξεις σχετικά με την κατάσταση των ανθρώπινων δικαιωμάτων στη χώρα μας και είμαστε ο συνδετικό κρίκος μεταξύ του πληθυσμού και των ε, αρχών. Φροντίζομαι ώστε οι νέοι νόμοι που ψηφίζονται να υπακούν στις διεθνείς ε, επιταγές. Τον Απρίλιο του 2008 πέρασε ο νόμος μας για την προστασία των ανθρώπινων δικαιωμάτων με την δυνατότητα προς ε, υπογραφής της συνθήκης ε, των, των Ηνωμένων Εθνών για την προστασία των ανθρώπινων δικαιωμάτων και την απαγόρευση των βασανιστήριων το, ιδρύθηκε και Συμβούλιο Πρόληψης Βασανιστήριων που, στο οποίο συμμετέχουν και δικοί μας εκπρόσωποι ανεξάρτητοι εμπειρογνώμονες, ψυχολόγοι κλπ. και εκπρόσωποι της Οργανωμένης Κοινωνίας των Πολιτών με την οποία συνεργαζόμαστε και σε άλλους τομείς και πάλι εκεί με υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπάρχει και μνημόνιο συμφωνίας μεταξύ του θεσμού μας και 80 ε, μη κρατικών οργανώσεων που εργάζονται για διάφορα θέματα. Έχουμε αρχίσει ένα επικοδομητικό διάλογο και ανταλλάσσουμε εμπειρίε και προβαίνουμε σε συνεργασία για την προώθηση των ανθρώπινων δικαιωμάτων στην Αρμενία. Υπό το πρίσμα αυτό υποστηρίζουμε την ιδέα του Πολωνού συνήγορου ε, του πολίτη για να ενταχθούν τα ανθρώπινα δικαιώματα σε πολύ ευρύτερη συνεργασία. Η ανταλλαγή ε, ιδεών με τον Πολωνό ε, διαμεσολαβητή μα δίνει και την ευκαιρία να ενισχύσουμε τον θεσμό μα. Ελπίζουμε ότι η εμπειρία μα θα φανεί χρήσιμη και σε άλλου εταίρους μα και θα συνεχίσουμε την ανταλλαγή των βέλτιστων πρακτικών μα και βεβαίω την αμοιβαία υποστήριξη για το ξεπέρασμα των κοινών προκλήσεων. Θα ήθελα εν τέλει να σα συγχαρώ για την εξαιρετική αυτή διοργάνωση και να εκφράσω την ελπίδα ότι η ευρεία συμμετοχή στην ε, παρούσα εκδήλωση θα εξασφαλίσει και τη μελλοντική μας συνεργασία. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Όντως, πειθαρχήσατε όσον αφορά το χρόνο που είχατε στη διάθεσή σας. Ούτε καν πέντε, τα πέντε σας λεφτά δεν χρησιμοποίησατε, αλλά έτσι κι θα έχετε την ευκαιρία να παρεύετε και πάλι μετά από τις ερωτήσεις που θα ακούσουμε από τους ευρωβουλευτές. Ο... Τώρα η καθηγήτρια Ελμύρα Σουλιμάνοβα έχει το λόγο που είναι η συνήγορος του πολίτη από το Αζερβαϊτζάν. Ευχαριστώ πολύ κυρίες και κύριοι. Πρώτα απ' όλα θέλω να σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση που μου κάνατε προκειμένου να έρθω εδώ και θέλω να αναφερθώ ιδιαίτερα όσον αφορά τον εκδημοκρατισμό που έχουμε στη χώρα για θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων και κράτους δικαίου. Υπάρχει μια διαδικασία μεγάλων αλλαγών στη χώρα επικύρωση πάνω από 200 συμβάσεων. Επίσης η εθνική νομοθεσία τροποποιείται για να συμμορφώνεται με τις συμβάσεις αυτές. Και επίσης υπάρχουν και πολλά διεθνή σχέδια στα οποία συμμετέχουμε, αλλά και βέβαια πολλά ευρωπαϊκά. Προς ενημέρωσή σα, θέλω να σας πω ότι το δικό μας Ινστιτούτο του Συνήγορου του Πολίτη δημιουργήθηκε στο Αζερβαϊτζάν και κλέστηκε ο πρώτος συνήγορος του πολίτη το 2002. Έχουμε μια περιορισμένη εντολή. Η εντολή αυτή όμως σιγά σιγά επεκτάθηκε και συμπεριέλαβε και περισσότερες αρμοδιότητες. Το πρόγραμμα αυτό της Ανατολικής Συνεργασίας ξεκίνησε το 2009 στις 29 Σεπτεμβρίου είχαμε τη διάσκεψη της Βαρσοβίας όπου εγκρίθηκαν συγκεκριμένες προδιαγραφές και εμείς συμμετέχουμε, το Ινστιτούτο μας δηλαδή, ε, συμμετέχει από το 2011. Συμμετέχουμε λοιπόν στο πρόγραμμα αυτό αλλά και σε άλλα. Προγράμματα τα οποία κάνουμε σε συνεργασία και με το αντίστοιχο Ινστιτούτο της Γερμανίας προκειμένου να, να ενισχυθούν οι αρμοδιότητες του συνήγορου του πολίτη και να ενισχυθούν οι ελευθερίες και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Ένα κομμάτι του προγράμματος αυτού είναι σεμινάρια κατάρτισης στα οποία συζητιούνται θέματα προστασίας των πολιτών και ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Στον Κάφκασο για πρώτη φορά, στο Αζερβαϊτζάν είχαμε ένα τέτοιο πρόγραμμα και στέφθηκε από επιτυχία. Το Ινστιτούτο μας επίσης συμμετέχει, όπως είπαμε, και στο πρόγραμμα Ανατολικής Συνεργασίας από την αρχή. Η Πολωνία το συντονίζει. Στα πλαίσια του προγράμματος αυτού έλαβαν χώρα δύο σεμινάρια κατάρτιση το ένα στην Πολωνία και τον άλλο στον Πακού με συμμετοχή του προσωπικού μας. Θέματα ήταν ε, καταπολέμηση των βασανισμών, ε, ψυχολογική υποστήριξη θυμάτων ε, εγκληματικών πράξεων και άλλα θέματα που αποτελούν προκλήσεις στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, πώς να χρησιμοποιούνται νέες τεχνολογίες, τι προοπτικές υπάρχουν για παρετέρω συνεργασία κλπ. Όλα αυτά συζητήθηκαν σε λεπτομέρειες με διάφορες εναλλακτικές λύσεις που ακούστηκαν. Επιπλέον, όλα αυτά τα χρόνια εμείς διμερώς προσφέρουμε τη συνεργασία μας σε άλλους συνηγόρους του πολίτη, 12 χώρες, Πολωνία, Ρωσία, Ουκρανία, Γεωργία και την τελευταία συμφωνία την υπογράψαμε με τη Μολδαβία. Ε, συμμετέχουμε επίσης και στο Συμβούλιο της Ευρώπης, στο πρόγραμμα του Συμβουλίου της Ευρώπης, με άλλα εθνικά Ινστιτούτα επίσης και υπάρχει και ένα δίκτυο στο οποίο συμμετέχουμε για την ε, πρόληψη παραβιάσεων ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Εμείς βελτιώνουμε τις δραστηριότητές μας, αυτό αποτελεί προτεραιότητα για μας. Πρώτα απ' όλα βάζουμε την ασφάλεια την ε, ανοχή. Προγράμματα πολύ σημαντικά για όλες τις χώρες πιστεύουμε, γιατί έτσι αποφεύγουμε ε, προβλήματα συγκρούσεων ή έτσι βοηθάμε να λύνονται οι συγκρούσεις. Έχουμε ένα εκατομμύριο πρόσφυγες εμείς στο Αζερβαϊτζάν. Τα τελευταία 20 χρόνια υποφέρουν επίσης από τη διαμάχη του Ναγόνο Καραμπάχ και εξαιτία πολιτικών ε, εθνικής κάθαρσης. Υπάρχουν και άλλες προτεραιότητες που έχουμε, που είναι η αντιμετώπιση ε, θεμάτων που έχουν να κάνουν με τους βασανισμούς, ε, όπως επίσης θέλουμε να βοηθήσουμε και τα άτομα με αναπηρίες. Θέλουμε να ενισχύσουμε τις αρμοδιότητες του συνήγορου του πολίτη ως Ινστιτούτο Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων με έναν μηχανισμό ανεξάρτητο ελέγχου και εποπτείας και προστασίας ατόμων με αναπηρίες. Επίσης θέλουμε να ενισχύσουμε και τους περιφερειακούς συνηγόρους του πολίτη. Πιστεύουμε ότι όλα αυτά τα θέματα είναι θέματα τα οποία μπορούμε να συζητήσουμε σε συνεργασία με άλλους. Τέλος, αναγνωριζόμαστε σαν Εθνικό Ινστιτούτο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων από την Υποπιτροπή σας και είμαστε διαπιστευμένοι. Πρέπει να ξέρετε ότι εμείς πιστεύουμε ότι μπορούμε να βοηθήσουμε πολύ το Ευρωπαϊκό Αντίστοιχο Πρόγραμμα. Ευχαριστώ. Σας ε, ευχαριστούμε. Θα ήθελα τώρα να δώσω το λόγο στην κυρία Τατιάνα Κουντσάρια από διαμεσολαβήτρια της Γεωργίας. Πολύ ωραία το, το προφέρατε το όνομά μου κύριε Πρόεδρε. Θα προσπαθήσω να είμαι σύντομη και ας μην χρησιμοποιήσω το έξτρα λεπτό που δεν χρησιμοποίησε ο Ουκρανός. Ο διαμεσολαβητής μας της Γεωργίας δυστυχώς κολλείεται, βρίσκεται στην Ουκρανία και συζητεί θέματα με την κυρία Καρπάσοβα του μηχανισμού πρόληψης ε, βασανιστήριων. Και αυτό τον δικαθιστώ σήμερα εδώ. Δεν θα έλθω στο ιστορικό του εγχειρήματο αφού όλοι και όλες γνωρίζουμε πώς άρχισε αρχές του 2009 αλλά βέβαια τα πραγματικά εγκαίνια ας πούμε έγιναν τον Δεκέμβριο 2009 με την πρωτοβουλία του καθηγητού Ορανόφσκι και προχωρήσαμε μετά στο μνημόνιο συμφωνίας διμερούς συνεργασίας με συμμετοχή όχι δυστυχώς όλων ε, παρόντων ε, εκπροσώπων το θεσμικό μας ιστορικό αλλά και η δική μου προσωπική εμπειρία ως αναπληρώτριας διαμεσολαβήτριας δείχνει ότι η συνεργασία μεταξύ του θεσμού μας, του Γεωργιανού θεσμού δηλαδή και του Πολωνικού θεσμού πάντοτε υπήρξαν πάρα πολύ ενδιαφέρουσες και σημαντικές. Δεν λέω τίποτε για άλλες χώρες που προσωπούνται στο ίδιο εγχείρημα και γι' αυτό το λόγο θα ήθελα να τονίσω και πάλι την σημασία του εγχειρήματο που θα υπηρετήσει την ε, ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών αλλά και εμπειριών. Μέσα στα πλαίσια αυτού του project της Ανατολικής Γειτονίας η Γεωργία συμμετέσχε σε δύο συναντήσεις που και οι δύο έλαβαν χώρα το 2010 η μία ήταν ένα, ήταν ένα σεμινάριο μάλλον με συμμετοχή Πολωνών, Μολδαβών, Γάλλων και Γεωργιανών το 2010 στην Τυφλίδα και μετά ακολούθησε άλλη συνάντηση αμέσως, αμέσως μετά και που έγινε και στη Βασοβία και στην Κρακοβία πάλι με συμμετοχή ε, Γάλλων, Μολδαβών, Γεωργιανών και Πολωνών. Προσωπικά, δυστυχώς δεν μπόρεσα να συμμετάσχω στις ε, συναντήσεις αυτές, αλλά βέβαια με, η ενημέρωση που μου έδωσε το προσωπικό μου ήταν πάρα πολύ θετική. Τον Οκτώβριο του 2010 έγινε η διάσκεψη στην Τυφλίδα με εκπροσώπους με εκπροσώπους αυτών των οργανώσεων, των ε, θεσμών δηλαδή και συζητήθηκαν γενικότερα θέμα, θέματα όπως οι αρμοδιότητες ε, των διαμεσολαβητών. Ένα άλλο θέμα ήταν ο ε, Εθνικός Μηχανισμός Πρόληψης είχε προβλεφθεί και επίσκεψη σε γεωργιανό σοφροναστικό κατάστημα και διεξήχθη αυτή η επίσκεψη και μετά από την επίσκεψη αυτή οι συνάδελφοι συζήτησαν τις κύριες διαφορές των σοφρονιστικών συστημάτων στις χώρες τους. Το άλλο, ήταν, το άλλο θέμα ήταν η αποζημίωση θυμάτων ε, αδικών πράξεων η καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού και θέματα κοινωνικών ασφαλίσεων. Και στην επόμενη συνάντηση που έγινε πλέον στην Πολωνία τον Νοέμβριο του ίδιου έτους στην συνάντηση εκείνη συνεχίστηκε η συζήτηση των ίδιων θεμάτων. Αξίζει να σημειωθεί ότι η σημασία των συναντήσεων αυτών είναι μεγάλη, διότι αποτελούν το εργαλείο, την δυνατότητα να ανταλλάσσουμε εμπειρίες. Βέβαια, επισημαίνω μία έλλειψη του εγχειρήματο και ζητώ συγγνώμη εκ των προτέρων, διότι θεωρώ Α το πω αλλιώς, έχουμε, έχουμε ακόμη δύο χρόνια. Τα πρώτα δύο χρόνια έδειξαν ότι είναι αποτελεσματικό, είναι ενδιαφέρον και χρήσιμο. Όταν όμως θα σχεδιάζουμε, θα προγραμματίζουμε τις δραστηριότητες μας των επόμενων δύο ετών, θα είναι καλό να κάνουμε μια αποκοινού οργάνωση με συμμετοχή όλων όχι μόνο δηλαδή των, όπως των συναντήσεων που έγιναν μόνο στην Τυφλίδα και στην Βαρσοβία. Ευχαριστούμε βεβαίως ε, τους θεσμούς, τον γαλλικό, τον μολδαβικό, τον ουκρανικό. Έχουμε όμως πολλά κοινά στοιχεία με τους Ουκρανούς, τους Αζερμπαϊτζανούς κλπ. Ίσως λοιπόν την επόμενη φορά να μπορέσουμε να προγραμματίσουμε τις συναντήσεις μας όλοι μαζί. Α, εδώ τελειώνει ο χρόνος μου. Ε, λοιπόν, πολύ ήθελα βέβαια να μιλήσω και λίγο για το θεσμό μας, αλλά δεν μου έμεινε άλλος χρόνος. Ίσως αργότερα μπορώ να επανέλθω. Σας ευχαριστώ πολύ Ανατόλη Αμουντάνο από την ε, Μολδαβία. Είναι μεγάλη τιμή για μένα να μπορώ να σας απευθύνω χαιρετισμό και εξ ονόματός μου αλλά και όλων των συνεργατών μου ε, του διαμεσολαβητού ε, της Μολδαβίας και να σα ευχαριστήσω που μας δίνετε την ευκαιρία να συμμετάσχουμε στη σημαντική αυτή συνάντηση. Για την δημοκρατία της Μολδαβίας η συνεργασία αυτή έχει μεγάλη σημασία. Η χώρα μας διέρχεται μια διαδικασία προς την κατεύθυνση της Ευρωπαϊκής Ενοποίησης. Την τελευταία διετία μετά από την υπογραφή της σχετικής δήλωσης η Δημοκρατία της Μολδαβίας έχει επιζητήσει τον διάλογο με τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα για θέματα όπως ε, ε, ε, μετακινήσεις χωρίς προξενικές θεωρήσεις, ταξίδια δηλαδή, ελεύθερη διακίνηση, ελεύθερη διακίνηση στους εθέρες κτλ. Για αυτά χρειάζεται η αποτελεσματική συνεργασία όλων των θεσμών επί των οποίων βασίζεται το κράτος και ταυτόχρονα πρέπει οι διαμεσολαβητές, οι συνήγοροι των πολιτών, να αποτελούν βέβαια τον κατεξοχήν εγγυητή των ανθρώπινων δικαιωμάτων στις χώρες της Ανατολικής Γετωνίας. Μακροπρόθεσμος στόχος του προγράμματος συνεργασίας μεταξύ των ε, συνηγόρων πολιτών ε, των χωρών της Ανατολικής Γετωνίας απαιτεί εξέταση των εθνικών νομοθεσιών καθώς και προσαρμογή τους στις ευρωπαϊκές προδιαγραφές. Επίσης, προστασία των ανθρώπινων δικαιωμάτων, καταπολέμηση των βασανιστήριων, ομαλοποίηση της ε, κατάσταση διαβίωσης των κρατουμένων στις φυλακές και ούτω καθεξής. Δεν θα επισέλθω σε λεπτομέρειε σε ό,τι αφορά τις επιτυχίες, και ενδεχομένω και τα σφάλματά μα, αλλά μεταξύ 23 και 25 Οκτωβρίου 2009 στο Νατολίν στην Πολωνία διεξήχθη ευρωπαϊκό σεμινάριο σχετικά με, την, με τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων μέσα στα πλαίσια των χωρών της Ανατολικής Γειτονίας. Με συμμετοχή των συνηγόρων πολιτών από Μολδαβία, Πολωνία και Γαλλία και εκεί προέβησαν σε ανταλλαγή απόψεων για θέματα σεβασμού των ανθρώπινων δικαιωμάτων. Κατόπιν, στο διάστημα από 10 έως 14 Μαΐου 2010 διεξήχθησαν εργασίες στην ίδια τη Μορδαβία, μετά στην Γεωργία και στην Πολωνία και οι συνήγοροι του πολίτου προσπάθησαν να διαγράψουν τα κοινά προβλήματα και να αναζητήσουν κοινέ λύσεις προτείναμε νομοθετικές λύσεις που μπορούν να εφαρμοστούν σε χώρες της Ανατολικής Γειτονίας. Έγιναν ανταλλαγές απόψεων. Προβήκαμε σε ανταλλαγή των βέλτιστων πρακτικών στους τομείς της προστασίας των ανθρώπινων δικαιωμάτων. Οι μέχρι τώρα εμπειρίες μου ως επικεφαλής Εθνικού Θεσμού για την Προστασία των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αλλά και εκ της συμμετοχή μου στο εγχείρημα αυτό μου, επιτρέπει, μου επιτρέπουν οι εμπειρίες μου αυτές να ισχυριστώ ότι πρέπει να προγραμματίζουμε έγκαιρα τα θέματα ότι πρέπει να εφαρμόζεται μια συγκριτική μεθοδολογία να γίνονται στην πράξη ανταλλαγές καθώς και ανταλλαγές επισκέψεων μεταξύ των θεσμών μας Πρόκειται για υποδειγματική συνεργασία. Ήδη το 2011, μέσα στα πλαίσια της διεθνούς ε, διασκέψεως για την κύρωση ε, της συμβάσεως για τα δικαιώματα των ανθρώπων της, ε, με, με ειδικέ ανάγκες, με το Αζερμπαϊτζάν προχωρήσαμε σε υπογραφή συμφωνίας συνεργασίας. Θεωρώ ότι ο θεσμός του οποίου ηγούμε θα πρέπει να συνεχίσει να εκμεταλλεύεται τις ευκαιρίες που διαθέτει μέσα στα πλαίσια της ανατολικής γειτονίας και σε διμερές αλλά και σε πολυμερές επίπεδο ώστε στο μέλλον να μπορέσουμε να συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε σε ισότιμη βάση. Ευχαριστούμε πολύ. Τώρα το λόγο έχει η κυρία Ιρένα Λίποβιτς. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ που μου δίνετε το λόγο κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, αγαπητοί συνάδελφοι και αγαπητοί συνεργάτες του προγράμματος αυτού Ανατολικής Συνεργασίας, όπως επίσης ε, χαιρετίζω και την παρουσία του Γάλλου διαμεσολαβητή. Εμείς χρηματοδοτούμε τη συνεργασία των διαμεσολαβητών στην Ευρώπη και αυτό πιστεύω ότι η πρωτοβουλία αυτή έχει ήδη αποφέρει καρπούς. Με τον τρόπο αυτό, με τη στήριξη αυτή δηλαδή, μπορούμε να έχουμε θετικά αποτελέσματα. Εμείς προσπαθήσαμε να δώσουμε μια απάντηση σε όλα αυτά που μας ζητάτε. Και αυτό ακριβώς είναι το οποίο μας οδήγησε να καταλήξουμε, να χωρίσουμε την έκθεσή μας σε διαφορετικά τμήματα. Εγώ συμφωνώ με τους προλαλήσαντες που λένε ότι θα προτιμούσαν να είχε γίνει μια συνάντηση πιο νωρίς όλων των αντιπροσωπιών, αλλά παρόλα αυτά θέλω να ευχαριστήσω όλους τους συνηγόρους του πολίτη και τον Γάλλο για την ανοιχτή και ειλικρινή συζήτηση που είχαμε. Όντως έπρεπε να είναι μια ανοιχτή ανταλλαγή απόψεων στην Πολωνία, σε όλες τις διασκέψεις, σε όλες τις συζητήσεις που κάνουμε για τα προγράμματα. Προσπαθούμε να δείξουμε την πραγματικότητα. Εμείς θέλουμε να δείξουμε και τα δυνατά και τα αδύναμα σημεία της Πολωνίας στο δρόμο που ακολουθήσαμε εμείς. Οι συμμετέχοντες νομίζω ότι μάθανε πολλά ενδιαφέροντα πράγματα και το προσωπικό μου με ευχαρίστησε για τη δυνατότητα που είχαν να συναντηθούν με τους συνηγόρους του πολίτη άλλων χωρών γιατί έτσι είχαν μια ειλικρινή ανταλλαγή απόψεων και εμπειριών. Πολύ καλή δηλαδή αυτή η συνεργασία, η ανατολική συνεργασία. Μιλάω εξάλλου νομίζω και εκ μέρους του κύριου Μποντής από τη Γαλλία όταν λέω ότι δεν θα θέλαμε το πρόγραμμα αυτό να περιοριστεί σε αυτές τις χώρες. Πιστεύω ότι εμείς μπορέσαμε και δημιουργήσαμε κάτι βιώσιμο και ήδη εντοπίζουμε τα θετικά από τη συνεργασία αυτή. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελεί γόνιμο έδαφος για τέτοιου είδους συνεργασίες. Και εμείς είμαστε ευγνώμονες που σήμερα το απόγευμα βρισκόμαστε εδώ και με, με περηφάνεια μπορούμε να σας δείξουμε τα επιτεύγματά μας. Πολύ θα θέλαμε την αναγνώριση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη συνεργασία μας αυτή. Να μας πει δηλαδή η Ευρωπαϊκή Ένωση ότι ανταποκρίνεται στους στρατηγικούς στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νομίζω ότι ισχύει αυτό στις, ε, στα τέλη Σεπτεμβρίου στη διάσκεψη της Βαρσοβίας που είχαμε για την Ανατολική Συνεργασία αναφέρθηκαν τα ανθρώπινα δικαιώματα στη δήλωση. Αυτό δείχνει και ποια είναι η θέση μας και ότι εμείς πιστεύουμε στα ανθρώπινα δικαιώματα. Από εδώ και πέρα κοιτάμε προς τα μπρος, προς το μέλλον του προγράμματος αυτού. Θέλουμε να συνεχίσουμε με τον πολιετή προγραμματισμό και εξού και εξετάζουμε τις δραστηριότητε μας για το 2012. Πάντως, από αυτά που ακούσατε και από τους προλαλήσαντες, καταλαβαίνετε ότι για θέματα όπως είναι η Σύμβαση για την Πρόσβαση Ατόμων με Αναπηρίες, οι θέματα που έχουν να κάνουν με εθνικές μειονότητες και τα δικαιώματά τους ή για θέματα που έχουν να κάνουν ε, με τις εκλογές, εκλογικά δικαιώματα δηλαδή και μη διάκριση βάση ε, κλπ. Όλα αυτά είναι θέματα τα οποία είναι στην ε, ημερήσια διάταξή μας και είναι θέματα τα οποία καλύφθηκαν από τη διάσκεψη της Πολωνίας. Θα θέλαμε να πούμε περισσότερο σε λεπτομέρειες και να μιλήσουμε για παράδειγμα για ε, διατάξεις σχετικά με τα παιδιά τα οποία είναι θύματα κάποιας εγκληματικής πράξης. Θέλουμε δηλαδή να φροντίσουμε τα παιδιά αυτά ε, μία μόνο φορά να πρέπει να μεταφέρουν την υπόθεσή τους στις αρχές, να μην χρειάζεται να περνάνε ξανά και ξανά από ανακρίσεις. Θέλουμε επίσης να κάνουμε περισσότερα πράγματα για να συμμετέχουν οι μη κυβερνητικέ οργανώσεις στο έργο μας. Θέλω πάντως να ευχαριστήσω όλους όσοι έβαλαν τόσο πολλές προσπάθειες στις δραστηριότητές μας. Είναι βαθιά μου πεποίθηση ότι μπορούμε να είμαστε περήφανοι για το έργο μας Ακριβώς γιατί δόθηκε πολύ μεγάλη σημασία στον Εθνικό Μηχανισμό πρόληψη. Εμεί δεν θέλουμε εδώ να καλύψουμε τα δύσκολα πράγματα, να τα βάλουμε κάτω από το χαλί, όχι. Αλλά πιστεύουμε ότι η συζήτηση πρέπει να είναι ανοιχτή για να καταφέρουμε με δημιουργικό τρόπο να δώσουμε λύσεις στα προβλήματα τα σημερινά και τα μελλοντικά. Ευχαριστούμε την καθηγήτρια. Να δώσουμε τώρα το λόγο στον κύριο Ντομινίκ Μποτέ. <coughs> Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε και ευχαριστώ την Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων που οργάνωσε ε, τη συνάντηση αυτή. Χαίρομαι πολύ επίσης που μπορώ εδώ να ευχαριστήσω και για την πρωτοβουλία της Πολωνίας, για την ε, ανατολική αυτή συνεργασία η οποία ξεκίνησε το 2009 με την προκάτοχο με τον προκάτοχο, τον κύριο Κοβανόφσκι, προκάτοχο της κυρίας Λίτοβιτς και με το δικό μου ε, προκάτοχο, τον Σαπόλ Ντελβουά, που ήταν ε, συνήγορος του πολίτη της Γαλλικής Δημοκρατίας. Και χαίρομαι που βλέπω εδώ τους συναδέρφους από τις έξι χώρες που συμμετέχουν στην συνεργασία αυτή και χαίρομαι που βλέπω ότι συνεχίζεται η δράση μας. Εδώ θέλω να ενημερώσω και τους συναδέρφους εδώ και τους ε, ευρωβουλευτές και τους εκπροσώπους της Κομισιόν για μια θεσμική μεταρρύθμιση που έλαβε χώρα στη Γαλλία φέτος. Δεν είμαι πια ε, συνήγορος του πολίτη της γαλλικής δημοκρατίας. Είμαι δηλαδή, αλλά ε, βάσει της μεταρρύθμισης αλλάζει το όνομα και τώρα είμαι ε, συνήγορος των δικαιωμάτων. Και δεν είναι μόνο γλωσσική αλλαγή, είναι και νομική, με πολλές συνέπειες. Θετικές, πιστεύω, για τους πολίτες. Πρώτον, ο συνήγορος των δικαιωμάτων πριν ονομαζόταν στη Γαλλία διαμεσολαβητής ε, φέρνει και μια συνταγματική αλλαγή. Με ένα παραπάνω νομικό βάρος από ό,τι είχε ε, η προηγούμενη θέση. Άρα λοιπόν πρόκειται τώρα για μια συνταγματική αρχή και για μια αρχή της οποίας η ανεξαρτησία διασφαλίζεται καλύτερα. Και διασφαλίζεται καλύτερα μέσω μιας διαδικασίας ορισμού όπου συμμετέχει η εκτελεστική εξουσία και το κοινοβούλιο. Πριν ο διαμεσολαβητή τη Γαλλική Δημοκρατία οριζόταν από τον ε, πρόεδρο τη Γαλλική Δημοκρατία. Σήμερα ο συνήγορο των δικαιωμάτων προτείνεται από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, αλλά στη συνέχεια περνά από ακρόαση στην ε, Γαλλική Εθνοσυνέλευση, η οποία μπορεί να αντιταθεί στον ορισμό, αν θέλει. Άρα λοιπόν συμμετέχει εδώ και εκτελεστική εξουσία, αλλά και ε, η Βουλή. Κάτι το οποίο διασφαλίζει την ανεξαρτησία. Έπειτα, έχουμε περισσότερα μέσα. Ο συνήγορος των δικαιωμάτων έχει ε, περισσότερες δυνατότητες δράσης στη δικαιοσύνη, έχει περισσότερες δυνατότητες να ζητήσει γνωμοδότηση από άλλα θεσμικά όργανα της Γαλλικής Δημοκρατίας. Μπορεί να ζητήσει από άτομα νομικά και φυσικά να έρθουν σε ακρόαση, μπορεί να προχωρήσει ε, και να κάνει κατασχέσεις ή μπορεί να προχωρήσει και σε διάφορες δραστηριότητε που τον βοηθάνε στο έργο του. Έχει επίσης ένα ανοιχτό πεδίο μπροστά του. Πριν από τη μεταρρύθμιση, ο πολίτης έπρεπε να περάσει από έναν βουλευτή, ευρωβουλευτή, από έναν γερουσιαστή, προκειμένου να έχει πρόσβαση στον διαμεσολαβητή της Γαλλικής Δημοκρατίας. Ενώ σήμερα κάθε άτομο μπορεί από μόνο του, χωρίς κανένα περιορισμό, είτε είναι γαλλικής υπηκότητας, είτε όχι, οποιοδήποτε βρίσκεται σε γαλλικό έδαφος μπορεί να ζητήσει κάτι από τον συνήγορο των δικαιωμάτων. Ένας ανήλικος για παράδειγμα μπορεί να το κάνει αυτό. Και η αίτηση άρα έρχεται απευθείας και είναι και δωρεάν. Ένα άλλο βασικό στοιχείο είναι ότι ο συνήγορος των δικαιωμάτων στη Γαλλία συγκεντρώνει τέσσερις θεσμούς οι οποίοι υπήρχαν πριν είναι ο διαμεσολαβητής της Γαλλικής Δημοκρατίας, γνωστό, το αντίστοιχο τον Ombudsman, που υπάρχει εδώ και 40 χρόνια στη Γαλλία, αλλά προστίθενται σε αυτό και τρεις άλλες ε, περιπτώσεις που βρίσκονται στην περίμετρο των αρμοδιατήτων του συνήγορου των δικαιωμάτων. Είναι ο διαμεσολαβητής, όπως είπαμε, της Γαλλικής Δημοκρατίας. Είναι επίσης ο συνήγορος των παιδιών, που υπάρχει πάνω από 10 χρόνια τώρα. Υπάρχει η Επιτροπή Δεοντολογίας για την Ασφάλεια, που επίσης υπάρχει εδώ και πάνω από 10 χρόνια και που φροντίζει για την τήρηση της διοντολογίας από όλε τις υπηρεσίες ασφάλειας. Την αστυνομία, τη χωροφυλακή, τη δημοτική αστυνομία, ιδιωτικούς οργανισμούς ασφάλειας κλπ. Και τέλος, Υπάρχει μια άλλη αρχή που ονομαζόταν στη Γαλλία Άλντε, που ήταν ε, η ανώτατη αρχή κατά των διακρίσεων και προώθησης της ισότητας. Ήταν δηλαδή ένα όργανο το οποίο είχε σαν καθήκον να καταπολεμά τις 18 διακρίσεις που έχουν εντοπιστεί, διακρίσεις που οφείλονται είτε στην προέλευση του ατόμου, είτε στο φίλο του, είτε σε κάποια αναπηρία που έχει, στον ε, ε, σεξουαλικό προσανατολισμό του κλπ. Αυτά τα τέσσερα όργανα λοιπόν τώρα γίνονται, μπαίνουν μαζί και είναι υπό μία αρχή συνταγματική που είναι ο συνήγορος των δικαιωμάτων. Διαθέτουν ομάδες που έχουν συγκεντρωθεί με περισσότερα νομικά μέσα στη διάθεσή τους, κάτι το οποίο πιστεύω θα μας βοηθήσει να επεξεργαστούμε ακόμα καλύτερα τις 100.000 περίπου προσφυγές που μας στάνουν κάθε χρόνο. Και θα ολοκληρώσω με το εξή. Έχουμε τρία μέσα δράσης στους τέσσερις τομείς που ανέφερα. Τα τρία μέσα που έχουμε είναι ε, να διακανονίζονται ιδιωτικέ υποθέσεις. Στη συνέχεια έχουμε την πρόθεση των βέλτιστων πρακτικών για την ισότητα και τρίτον την δυνατότητα να προτείνουμε μεταρρυθμίσεις στο Κοινοβούλιο και στην κυβέρνηση. Οπότε έτσι και οι συναδελφοί μου και οι ευρωβουλευτές ενημερώθηκαν για τις εξελίξεις αυτές στη Γαλλία. Εννοείται ότι θα συνεχίσουμε με τον ίδιο τρόπο τη συνεργασία μας τα πλαίσια της ε, ανατολικής συνεργασίας, της οποίας την πρωτοβουλία είχε η Πολωνία, και συγχρόνω να σας πω ότι συμφωνώ απόλυτα με την πρόταση της κυρίας Λίποβιτς. Τη στηρίζω, δηλαδή να διευρύνουμε και σε άλλες χώρες την πρωτοβουλία αυτή στα πλαίσια της πολιτικής γετνίασης. Πιστεύω λοιπόν ότι θα ήταν ενδιαφέρον και στα πλαίσια που ζούμε τώρα από την αρχή του 2011 να σκεφτούμε πώς μπορεί να διευρυνθεί αυτή η πολιτική γυτνίασης ώστε να συμπεριλαμβάνει την διάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και να επεκταθεί ε, στη Μεσόγειο και από την νότια πλευρά της Μεσογείου επίσης. Να ξέρετε ότι είμαστε στην διάθεσή σας, χωρίς αυτό να σημαίνει βέβαια ότι θα βάλουμε λιγότερες προσπάθειες στην ανατολική συνεργασία, καθόλου. Ελπίζω πάντως ότι το 2012, εφόσον η Ευρωπαϊκή Ένωση μας δώσει τα μέσα, να οργανώσουμε ένα συμπόσιο, μερικές ημέρες δηλαδή, σε μία από τις χώρες εταίρους, στην Πολωνία, στο Παρίσι, όπου κρίνουμε ότι θα είναι το καλύτερο. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Μπούντι. νομίζω ότι από την πείρα σας ως εθνικός βουλευτής, όλα όσα έχετε κάνει στο Συμβούλιο της Ευρώπης, είναι στοιχεία τα οποία θα μας επιτρέψουν να διαχειριστούμε όλο αυτό το θέμα των δικαιωμάτων και των αρμοδιοτήτων στο οποίο αναφερθήκατε. Θα ήθελα τώρα να δώσω το λόγο στον εκπρόσωπο του EAS για πέντε λεπτά. Δεν ξέρω ποιος θα λάβει το λόγο. Ο κύριος Γιαννόφσκι, παρακαλώ. Thank you very much Ευχαριστώ πολύ. Καταρχάς για την πρόσκληση και κατά δεύτερον διότι μου δίνετε το λόγο. Άκουσα ιδιαίτερα προσεκτικά όλους τους ε, εκπροσώπους των διαμεσολαβητών και των ανθρωπινών δικαιωμάτων και θα ήθελα να τους ευχαριστήσω για την ε, συμμετοχή τους θα ήθελα να πω ένα-δύο πράγματα για το τι ακριβώς γίνεται για τον εκδημοκρατισμό ε, και τα θέματα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων εν γέννη. Η Ανατολική Συνεργασία εργάζεται σε δύο ε, πτυχές, ε, τη διμερή και την πολυμερή πτυχή. Αναφερθήκατε στα στοιχεία αυτά στις ομιλίες σας, αλλά θα ήθελα να τονίσω το θέμα της διμερούς πτυχής ε, εργαζόμαστε προς όφελος της βαθύτερης και βιώσιμης δημοκρατίας, ιδίως στις Επιτροπές Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και η κάθε χώρα με την Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναπτύσσει ε, τα διάφορα θέματα. Οι υποεπιτροπές αυτές ε, προς το παρόν ε, είναι επί τη βάση νομικώς δεσμευτικών διμερών μέσων ε, τα οποία έχουν ε, θεσπιστεί με κάθε χώρα. Η περιμερή πτυχή είναι νέα μετά από την εμπειρία του 2009 και εδώ προσπαθούμε να ενισχύσουμε αδυναμίες και τους αδύναμους κρίκους που έχουμε σε κάθε διμερές επίπεδο. Επί παραδείγματι, από το 2009 και μετά έχουμε ένα πολυμερές πλαίσιο σε πολλούς τομείς, όπως για παράδειγμα τη δημοκρατία, την καλή διακυβέρνηση και τη σταθερότητα. Στο πλαίσιο αυτό θα ήθελα να σας υπενθυμίσω την τελευταία συνεδρίαση που είχαμε σε πολυμερή επίπεδο, την αποκαλούμε πλατφόρμα 1, είναι η πλατφόρμα για τη δημοκρατία, τη σταθερότητα και τα ανθρώπινα δικαιώματα και εκεί παρουσιάστηκε το κοινό γαλλοπολωνικό πρόγραμμα και αποφασίστηκε να γίνουν περαιτέρω εργασίες γι' αυτό στο πολυμερές πλαίσιο. Αυτή τη στιγμή λοιπόν εκπονούμε το νέο πρόγραμμα εργασίας, το οποίο θα καλύψει την επόμενη διετία αυτών των ε, δημοσιονομικών προοπτικών ε, και θα παρουσιάσουμε και ένα πρόγραμμα εργασίας το οποίο θα περιλαμβάνει και κάποια στοιχεία τα οποία σας ενδιαφέρουν ιδιαίτερα. Αυτά λοιπόν ενημερωτικά για τα στοιχεία που έχουμε εμείς από πολευράς μας. Τώρα, στους τομείς ε, που επεσήμαναν οι συνάδελφοι. και που καλύπτουμε στο διμερές πλαίσιο έχουμε όλα τα θέματα επιμόρφωσης και κατάρτισης, ε, τα προγράμματα αδελφοποίησης και αυτό που αποκαλούμε το συνολικό πρόγραμμα δημιουργίας θεσμών. Αυτό είναι κάτι το οποίο ε, αναπτύξαμε για τις χώρες σας και σε κάποιες περιπτώσεις, όχι σε όλες, αλλά για παράδειγμα στην περίπτωση της Γεωργίας καλύπτει και το ε, συνήγορο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και κάποια από τα χρήματα τα οποία ανατίθενται διμερώς ε, στη Γεωργία για παράδειγμα θα δοθούν και για την ενίσχυση του συνογόρου των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα τώρα να ξεκινήσει η συζήτηση. Να δώσω και το λόγο στα μέλη της Επιτροπής μας. Η κυρία Λοχμπίλερ έχει ζητήσει το λόγο καταρχάς. Ευχαριστώ λοιπόν. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω και για τα όσα ακούσαμε από πλευρά σας. Είναι πολύ ενδιαφέρον να ακούμε τι γίνεται σε εθνικό επίπεδο και θα ήθελα να κάνω δύο σχόλια. Όταν σας άκουγα, ε, θυμήθηκα ε, τότε που εργαζόμουν εγώ στην Εργα... Γερμανία εκ μέρους κοινωνίας των πολιτών. Στις αρχές του 2000 ε, δημιουργήσαμε ένα ιδιωτικό ίδρυμα για τα ανθρώπινα δικαιώματα, γιατί η κυβέρνηση στη Γερμανία θεωρούσε ότι δεν υπήρχε ανάγκη. Και κατανόησα πόσο δύσκολο ήταν να υπάρχει ένα ανεξάρτητο όργανο, διότι όλοι όσοι ασχολούνται με την αστυνομία και ε, ε, τα θέματα δημοσίας τάξεως ε, ασκούν ε, ιδιαίτερη πίεση. Και αυτό δεν το ανέφερε κανένας από εσά ότι μπορεί να είστε και συνεχώς υποπίεση. Διότι όταν εκδίδεται μία έκθεση για τα εθνικά αποτελέσματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων και μπορείτε να επεξεργαστείτε την έκθεση αυτή και να τη διαβιβάσετε σε κάποιο διεθνή περιφερειακό φορέα, ε, σίγουρα αντιμετωπίζετε δυσκολίες και επομένω, ε, είναι μεγάλο ο αγώνας όχι μόνο για να τηρούνται οι αρχές του Παρισιού αλλά και για να πείσετε τον πληθυσμό και τους ασχολούνται με τα ανθρώπινα δικαιώματα στις χώρε. σα. Γι' αυτό και θα πρέπει να υπάρχει ευελιξία και να είστε ανοιχτόμυαλοι για να μπορείτε να αντιμετωπίσετε και τα προβλήματά σας εσωτερικώς. Γι' αυτό που είπε ο συνάδελφος από τη Μολδαβία, ε, με βρίσκει σύμφωνη. Ε, ισχύει δηλαδή ιδιαίτερα όταν πρέπει να αντιμετωπίσετε θέματα βασανισμών ή ε, κρατήσεις σε σοφρονιστικά καταστήματα. Ε, ανέφερε και κάποιος άλλος ότι είναι πολύ σημαντικό να δουλεύει κάποιος ανεξάρτητα και έχω μία ερώτηση και συγχωρέστε με για την αγνοία μου. Εγώ νόμιζα ότι στη Γαλλία υπάρχει Υπουργείο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων είναι ακόμα ενισχύ. Εάν όντω είναι ακόμα ενισχύ, θα ήθελα να ξέρω πώς ο συνήγορος του πολίτη ε, συνεργάζεται με το Υπουργείο. Επίσης θα ήθελα να σας ε, πω ε, για μια συζήτηση που είχαμε με το συνήγορο του πολίτη στη Νέα Ζηλανδία. Ε, υπήρχε μια εκπρόσωπο τη νέα Ζηλανδία από ένα δίκτυο ε, Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων που δημιουργείται στα πλαίσια των Ηνωμένων Εθνών. Συζητήθηκαν τα όσα κάνουν ε, αυτοί μαζί ε, μας. Ε, υπήρχαν και παλιότεροι και ε, νεότεροι οργανισμοί και επισήμαναν πόσο σημαντικό είναι να υπάρχει συνεργασία σε περιφερειακό επίπεδο. Και εδώ στις Βρυξέλλες, για παράδειγμα, δεν υπάρχει, ακόμα και με κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν υπάρχει μια μόνιμη αντιπροσωπεία που να ε, μοιράζεται την εμπειρία που έχουν ε, με τους εθνικούς οργανισμούς ή με τον συνήγορο του πολίτη. Ε, καλό θα ήταν να υπάρχει λοιπόν μια ανταλλαγή εμπειριών και όταν γίνεται λοιπόν άνοιγμα και με θεσμούς εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης να μοιράζεστε εμπειρίες και να στραφώ τώρα και στην Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης θέλουμε και υποστήριξη ώστε να υπάρχει τουλάχιστον μία μόνιμη δομή εργασίας για να παρακολουθούμε τα όσα συζητά η Ευρωπαϊκή Ένωση και που θα ήταν χρήσιμα και για σας. Και μια ερώτηση προς τον κύριο Τσέτσια που έκανε τη μελέτη. Θα μπορούσαμε ίσως να χρησιμοποιήσουμε και την εμπειρογνωμοσύνη που έχετε εσείς. και να τους ακούμε όταν η Ευρωπαϊκή Ένωση ετοιμάζει τις στρατηγικές αναχώρα. Θα ήταν χρήσιμο και να έχουμε τη δική του συνεισφορά. Και δεν ξέρω αν εμείς θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε τη δική σας εμπειρογνωμοσύνη, όλοι έχετε διάφορες γνώσεις ανάλογα με τα γραφεία σας και καλό θα ήταν να υπάρχει στενή επαφή και να μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τις γνώσεις σας για το τάδι το δίνα θέμα όταν ε, ε, ζητούμε μελέτες ή εξετάζουμε ε, υποψήφιους Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Ζέγκ. Σας ευχαριστώ πολύ για τη δυνατότητα που μου δίνετε να συζητήσουμε το θέμα αυτό και το γεγονός ότι μου δίνετε το λόγο για να μιλήσω για ένα πολύ σημαντικό θέμα. Όταν εξέτασα το θέμα αυτό στην ημερήσια διάταξη της συνεδρίασής μας, δεν είχα φανταστεί ότι η συζήτηση θα μας είχε αποδείξει ότι μιλάμε για ένα πολύ σημαντικό τομέα για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η πρωτοβουλία που συζητάμε είναι πολύ σημαντικό να υπενθυμίσουμε ότι είναι μόλις δύο ετών, αλλά είναι πολύ χρήσιμη και πολύ επίκαιρη και ως Πολωνός χαίρομαι ιδιαίτερα που το ε, Υπουργείο μας ε, ήταν ε, αυτό το οποίο σκέφτηκε τη συνεργασία αυτή. Θα ήθελα να σας εκφράσω τις ανησυχίες μου εδώ. Γνωρίζαμε ότι δεν θα είναι παρόν εκπρόσωπος της Λευκορωσία, διότι δεν υπάρχει κάποιο οργανισμός αυτής της μορφής στη Λευκορωσία, αλλά φαντάστηκα ότι θα υπήρχε τουλάχιστον κάποιος από την Ουκρανία, για να μπορέσουμε να συζητήσουμε πολλά μαζί του. Ίσως η απουσία να οφείλεται και σε διαδικαστικούς λόγους, μπορεί να υπήρχαν προβλήματα χρηματοδότησης ή να είναι για άλλη μια φορά απόδειξη του γεγονότος ότι οι αλλαγές ε, στην Ουκρανία είναι πάρα πολύ βραδίες, ιδιαίτερα όσον αφορά το σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων των πολιτών. Υπάρχουν πολύ σοβαρά προβλήματα και πολύ σοβαρά κενά στο σεβασμό των ε, θεμελιωδών αρχών. Θα ήθελα να μας δοθεί μία εξήγηση για την απουσία. Ήταν για οργανωτικούς και μόνον λόγων ή οι συνάδελφοι από την Ουκρανία αποφάσισαν συνειδητά να απόσχουν της σημερινή συνάντηση. Φαντάζομαι ότι αυτή η απόφαση τη σημερινη συναντηση φανταζομαι οτι αυτη η αποφαση εληφθη σε υψηλό επίπεδο. Όταν αναφερόμαστε στην ε, λειτουργία των Ινστιτούτων αυτών και το ρόλο των διαμεσολαβητών, όταν αναφερόμαστε στο σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων, των ε, θεμελιωδών πολιτικών δικαιωμάτων, αναφερόμαστε σε ζητήματα στρατηγική σημασία για την Ευρωπαϊκή Ένωση και ο σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων αποτελεί θεμέλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό που μα ενδιαφέρει όμως ε, επίσης είναι ο σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων και σε άλλες χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιδίω στι χώρες εταίρους μα. Και ιδίω σε χώρες που θα γίνουν εταίροι τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Όπως υπενθύμησε και η Πρόεδρος, και εγώ θεωρώ ότι η υπηρεσία εξωτερικής δράσης θα πρέπει να διαδραματίσει ουσιαστικό ρόλο. Έχουμε προσδοκίες και γι' αυτό και κάνουμε και το συγκεκριμένο αίτημα προς την υπηρεσία εξωτερικής δράσης. Σήμερα εδώ είναι παρούσες πολλές χώρες όπου υπάρχει ε, αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπάρχει σκέλος ε, της υπηρεσία εξωτερικής δράσης και είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει και διπλωματική παρουσία που θα ασχολείται με θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων και θα μπορούν να συνδράμουν και τους θεσμούς και τους οργανισμούς που δραστηριοποιούνται σε θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν να υπάρξει και διπλωματική υποστήριξη. Ε, η Γεωργία, επί παραδείγματι. Η Γεωργία είναι σαφώς ε, σημαντική χώρα, αλλά δεν είναι και η μόνη χώρα που συμμετέχει στην Ανατολική Συνεργασία. Θα πρέπει φυσικά να υπάρξει υποστήριξη και για τις άλλες χώρες. Θα ήθελα να πω επίσης ότι ε, είναι μια διαδικασία η οποία ξεκίνησε εδώ και πολύ λίγο καιρό και καλό θα ήταν να μην ε, ολοκληρωθεί στο τέλος της Πολωνικής Προεδρίας. Θεωρώ ότι είναι πολύ επίκαιρη και πολύ καλά στοχευμένη η όλη πρωτοβουλία και ε, είναι προ όφελο ε, των βασικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα πρέπει λοιπόν και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να σκεφτεί πώ μπορεί να βοηθήσει τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία. Ευχαριστούμε πολύ. Άλλο κανείς θέλει μήπως να πάρει το λόγο τώρα. Δεν βλέπω. Οπότε θα δώσω το λόγο στην κυρία Λίποβιτς, η οποία θέλει να απαντήσει. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ την κυρία Λόχμπιλα και τον κύριο Ζέμκε για τα καλά τους λόγια και ευχαριστώ πολύ και τους εκπροσώπους της Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης. Ίσως μπορώ να πω κάτι για τη Λευκορωσία. Φυσικά και θα θέλαμε η Λευκορωσία να συμμετέχει στην Ανατολική Συνεργασία. Ξέρουμε όμως ποια είναι τα προβλήματα. Μάλιστα έχω μια συγκεκριμένη πρόταση. Ε, ίσως είναι περισσότερο ευσεβής παρά πρόταση γιατί δεν έχουμε τους οικονομικούς πόρους γι' αυτό. Αλλά αυτό που θα είχα να προτείνω είναι αν βρίσκαμε τη χρηματοδότηση εμείς είμαστε έτοιμοι να συμπεριλάβουμε νέους φοιτητές ε, με υποτροφίες που θέλουν στο μέλλον να ασχοληθούν με τα ανθρώπινα δικαιώματα και να έρθουν στο δικό μας γραφείο του Πολωνού, δηλαδή συνήγορου του πολίτη, και να δουλέψουν εκεί ως καταρτιζόμενοι. Δεδομένου ότι και γλωσσικά και γεωγραφικά είμαστε κοντά, αυτό είναι κάτι το οποίο θα μπορούσε να είναι πολύ χρήσιμο. Είμαστε ανοιχτοί στην ιδέα του να ανοίξει η συνεργασία αυτή και σε άλλες χώρες. Αλλά συγκεκριμένα για τη Λευκορωσία, ειλικρινά, θα μπορούσε να έχει πολύ μεγάλη σημασία για το μέλλον. Διότι υπάρχουν εκεί νέοι που θέλουν να δουλέψουν για τα ανθρώπινα δικαιώματα εκεί και εμείς αν μπορούμε, ευχαρίστως να τους βοηθήσουμε. Έρχομαι τώρα στην Ουκρανία. Εδώ Είχαμε τόσο ενδιαφέρουσε ανταλλαγές με τους Ουκρανούς και ειλικρινά λυπάμαι πολύ που δεν έχουμε την Ουκρανή συνήγορο του πολίτη μαζί μας. Εμείς προσπαθούμε με τις επαφές που έχουμε να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Δεν θέλουμε να κρύβουμε κάτω από το χαλί τις δυσκολίες δεν προσπαθούμε να κρύψουμε τίποτα. Ευχαριστώ επίσης τον κύριο Μποντής για το γεγονός ότι στο γραφείο ε, της Πολωνίας υποδεχτήκαμε νέους που φιλοξενήσαμε από την Τινησία, για παράδειγμα, οι οποίοι συμμετείχαν στις αλλαγές εκεί και εγώ είμαι πολύ ανοιχτή σε τέτοιου είδου συνεργασία. Οπότε κατά κάποιο τρόπο έχει ήδη συμβεί το να δεχόμαστε νέους από άλλες χώρες. Έπειτα για το θέμα της περιφερειακής συνεργασίας που αναφέρθηκε από κάποιον εδώ, εμείς συνεργαζόμαστε με τους συνηγόρους που βλέπετε εδώ μπροστά σας, όχι μόνο όμως στα πλαίσια της συνεργασίας, της ανατολικής συνεργασίας, αλλά και στα πλαίσια των Ηνωμένων Εθνών. Έχουμε συνεργαστεί και υπό την αιγύδα των Ηνωμένων Εθνών για θέματα όπως είναι επισκέψεις σε φυλακές και πιστεύω ότι είναι μια μεγάλη ευκαιρία ειλικρινά οι συνάδελφοι από την Ανατολική Συνεργασία και αυτοί ε, θέλουν να ανοίξουν οι φυλακές ώστε να μπορούμε να τις επιθεωρήσουμε. Πρόεδρος, ευχαριστώ πολύ. Ο καθηγητής Κέντζα τώρα. Θέλετε και εσείς το λόγο μετά τα όσα ακούσατε. Παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. αφού, <clears throat> αφού δεν υπήρξαν ερωτήσεις. Αυτό που επιθυμώ να δηλώσω είναι ότι εποφελήθηκα από τις παρεμβάσεις και βέβαια και από τα πληροφοριακά στοιχεία που διαθέτουμε ήδη και από ορισμένα συμπληρωματικά. Με την ευκαιρία δε που ευρίσκονται εδώ οι διάφοροι εκπρόσωποι των εθνικών οργάνων. Θα ήθελα να παρακαλέσω τα γραφεία των θεσμικών αυτών οργάνων να μας παράσχουν όλες τις πληροφορίες που θεωρούν ότι θα είναι χρήσιμες για την συμπλήρωση της μελέτης. Θα είναι χρήσιμο να έχουμε τις πληροφορίες από τα ίδια τα θεσμικά αυτά όργανα και όχι μονάχα αυτές που μπορούμε να αντλήσουμε από σχετικά υλικά. Θα σημάνει αυτό μια ποιοτική διαφορά. Και θα ήθελα να παρακαλέσω τα θεσμικά αυτά όργανα να μας τις πληροφορίες. Έχουμε ήδη στείλει την σχετική αλληλογραφία και πολύ ευχαρίστως να αναζωογονήσω τις επαφές αυτές και να σας παράσχω όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για την διαβίβαση των πληροφοριών σχετικά με την εργασία σας. Πιθανώς θα είναι και η σημαντικότερη συμβολή που μπορούμε να έχουμε τις επόμενες εβδομάδες έτσι ώστε να ε, ολοκληρώσουμε την εργασία συντάξεως του εγγράφου. Σα ευχαριστώ, λέει ο Προεδρεύων. Κυρίε και κύριοι, δεν νομίζω να υπάρχουν άλλε ερωτήσεις από τα μέλη. Α, σχετικά με τα συμπεράσματα, κύριε Μποντή, Ίσως μπορούμε για τον τελευταίο γύρο να αρχίσουμε από εσάς. Ας δώσω ορισμένες απαντήσεις. Βεβαίως για τον ε, καθηγητή κύριο Κέτζια θα του διαβιβάσουμε όλα τα απαραίτητα έγγραφα. Ένα καινούριο θέμα είναι αυτό της συνεργασίας πολιτικής γειτονίας προς Νότον. Η κυρία Λίποβιτς είπε πριν ότι έχει λάβει, έχει δεχτεί μάλλον Αιγυπτίους, Τινησίους και είναι αληθές ότι βλέπουμε τους ομολόγους μας από την αντίπερα ακτή της Μεσογείου που έρχονται εδώ διμερώς να μας δουν. Οι διάφοροι συνηγοροί του πολίτη, δι, διάφορους μάλλον συνηγορούς του πολίτη εδώ, αλλά νομίζω ότι είναι χρήσιμο να διαφροθεί στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ίσως της Υπηρεσίας Εξωτερικών Δράσεων, μία συνεργασία βασισμένη στο ίδιο πρότυπο που υπάρχει ήδη για την ε, συνεργασία προς Ανατολάς. Γιατί βλέπουμε από την Αίγυπτο, την, την και κλπ. Άνθρωποι οποίοι θέλουν να προχωρήσουν τα θέματα ανθρώπινων δικαιωμάτων, αλλά βέβαια βρίσκονται αντιμέτωποι με δυνάμεις οι οποίες επιθυμούν μια οπισθοδρόμηση και νομίζω ότι έχουμε μια ιστορική ευθύνη. Και αυτή τη στιγμή δυστυχώς την αγνοούμε. Ιδού λοιπόν, ως παλαιό Ευρωβουλευτή σας τα λέω αυτά και ως νυν συνήγορο του πολίτου. Σας λέω ότι δυστυχώς με την εξέλιξη αυτή. Υπάρχει αυτή τη στιγμή ανοιχτή μια ευκαιρία, αλλά δεν θα μείνει ανοιχτή για πάντα. Μιλώ για τους ανθρώπους οι οποίοι από την άλλη πλευρά της Μεσογείου θέλουν να δημιουργήσουν ε, ε, όργανα τα οποία θα υπηρετήσουν τα ανθρώπινα δικαιώματα. Για τι ερωτήσει σα, κύριε Πρόεδρε, πράγματι υπήρξε ε, γραμματεία δικαιωμάτων ανθρώπου στη Γαλλία για έναν αριθμό ετών. Αυτή συγχωνεύτηκε τώρα στο Υπουργείο Εξωτερικών. Νομίζω, ωστόσο, ότι καλύτερα εξασφαλίζεται η προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων από μια ανεξάρτητη αρχή παρά από ένα μέλος της κυβερνήσεως που είτε το θέλουμε είτε όχι δεσμεύεται από ένα καθήκον αλληλεγγύης προς τον ε, συνάδελφό του Υπουργό των Εσωτερικών ή της Δικαιοσύνης ή των Κοινωνικών Υποθέσεων και δεν έχει εν τέλει την ελευθερία του λόγου όπως θα μπορούσε να την έχει ένα ανεξάρτητο όργανο με έναν μόνιμο ε, επικεφαλής και ε, που εν πάση περιπτώσει δεν θα μπορεί να εκδιωθεί από την θέση του. Υπήρξαν πιέσεις, ρωτήσατε. Θα σας δώσω την ίδια απάντηση που μου έδιναν παλαιά όταν ήμουν δημοσιογράφο δημοσιογράφος τηλεόραση. Ναι, υπήρξαν πιέσει. Το ζήτημα είναι όμως, μπορεί κανείς να αντισταθεί στις πιέσει, Εφόσον ανθίσταται κανείς στις πιέσει, τότε βέβαια πιέσει όλο και εξασθενούν και εν τέλει εξαφανίζονται. Θα πρέπει λοιπόν να λειτουργήσει κανείς στη βάση των φυσικών αρχών των ε, θυρών που όσο και περισσότερο όσο περισσότερο πιέζουν, τόσο περισσότερο κλείνουν. Μάλιστα, σας ευχαριστώ. Κύριε Μποντή, για τα συμπαράσματα που συναγάγατε και θα παρακαλέσω την κυρία Μπίλερ τώρα, πρόεδρό μας, να εξηγήσει για ποιο λόγο απουσιάζει ο Ουκρανός ε, εκπρόσωπος που νομίζω ότι οι λόγοι απουσίας του είναι μάλλον τεχνικοί. Καλά. Τήθηκε το θέμα της απουσίας της κυρίας Καρπάτσοβα από την Ουκρανία η οποία μου έγραψε για να μου πει ότι δεν μπορεί παρά μονάχα μετά τις 19 Οκτωβρίου. Δεν συζητήσαμε αν ίσως υπάρχει κάποιο θέμα, αλλά θα συστήσω η αντιπροσωπεία μας για τις σχέσεις με την Ουκρανική Βουλή, εγώ θα έλθω σε επαφή μαζί τους και θα τους παρακαλέσω την επόμενη φορά που θα επισκεφθούν την Ουκρανία να έλθουν σε επαφή μαζί της. Το, η επιστολή της ήταν απλώς για να δηλώσει το κόλλημα αυτό. Μάλιστα, σας ευχαριστώ. Υπάρχει τώρα τίποτε άλλο που θα ήθελα να δηλώσουν οι ε, προσκεκλημένη μας. Τελευταία σας ευκαιρία. Επανέρχομαι σε δύο θέματα. Ένα της Γεωργιανής συναδέλφου για την μεγαλύτερη δηλαδή αποδοτικότητα της συνεργασίας αυτής. Συνήθως θα πάμε στις δυτικές ευρωπαϊκές χώρες για να διεξαγάγουμε τις επαφές και να δούμε ποια πράγματα είναι χρήσιμα για μας, αλλά για τους επόμενους γύρους θα είμαστε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι εάν έλθουν οι ομόλογοι μας από τις δυτικές ευρωπαϊκές χώρες να εξετάσουν πιο συγκεκριμένα θέματα που, προέρχονται, που προκύπτουν από το δικό μας περιβάλλον, από τις δικές μας δημοκρατίες, ώστε αυτά να αποτελέσουν εισρωές από πιο έμπειρες χώρες σχετικά με το τι αντιμετωπίζουμε στις δικές μας χώρες τώρα. Και για το δεύτερο σχόλιο, πώς μπορούμε δηλαδή εμείς να αποβούμε γενικότερα χρήσιμοι ω εθνικοί οργανισμοί προστασίας των ανθρώπινων δικαιωμάτων στο διάλογο με τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και βέβαια με τις αρχές μας. Εδώ αντί να αντιδρούμε προτιμούμε να αναλάβουμε δράση και νομίζω ότι είμαστε οι πιο ευρωπαϊκοί θεσμοί στις χώρες μας με την κατανόηση και με την δική μας νοοτροπία μπορούμε να αποτελέσουμε διαμεσολαβητές μεταξύ ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων και των δικών μας εθνικών αρχών και βεβαίως ουδήποτε βουλευτού ή άλλου προσώπου από την Δυτική Ευρώπη που θα επιθυμούσε να εργαστεί μέσω ημών πολύ ευχαρίστως. Να σας προσφέρουμε δηλαδή και την τεχνογνωσία μας αλλά και τους πόρους που διαθέτουμε. Σας ευχαριστώ και πάλι για την ευκαιρία που μας δώσατε να προσέλθουμε και να συζητήσουμε μαζί Ευχαριστώ πολύ, κύριε Αντιδασιάν. Και άλλος κανείς. Really Πολύ σύντομα, ε, συνεχίζοντας αυτό που είπε ο Αρμένιος ε, συναδελφός μου, όχι μόνο μπορούμε να δείξουμε στους Ευρωπαίους ομολόγους μας τι κάνουμε ή ποιοι είμαστε. Μπορούμε, μάλιστα, να διδάξουμε κιόλας σε ορισμένες συγκεκριμένες υποθέσεις τους Ευρωπαίους συναδελφούς. Είμαστε ε, νεαροί θεσμοί βεβαίως εδώ. Από την άλλη μεριά αντιλαμβάνομαι από ορισμένε επισκέψεις που κάναμε σε ευρωπαϊκές χώρες ότι για παράδειγμα οι εθνικοί μηχανισμοί πρόληψης του γεωργιανού συνηγόρου είναι πολύ ισχυρότεροι από από ό,τι σε ορισμένους ευρωπαϊκούς ε, ε, οργανισμούς και εκεί πραγματικά νιώσα υπερήφανη για, για, τον, για, μας τους ίδιους. Μπορούμε λοιπόν βεβαίως και να διδαχθούμε από τους Ευρωπαίους συναδέλφους μας, αλλά ταυτόχρονα μπορούμε και να τους διδάξουμε. Ορισμένα πράγματα. Ευχαριστούμε, κυρία Κουντσάρια. Η κυρία Σούλεμάνοβα τώρα, παρακαλώ. Ευχαριστώ. Θέλω εγώ να αναφέρω ότι έχουμε συμμετοχή σε όλο και περισσότερα δίκτυα, διεθνή δίκτυα, στο νέο μηχανισμό, για παράδειγμα, για την περιοδική αναθεώρηση. Είναι κάτι πολύ χρήσιμο, γιατί έτσι μπορούμε να αναλύσουμε όλες τις προσφυγές που μας έρχονται, να ανακαλύψουμε τι παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων γίνονται, τι ελλείψεις υπάρχουν και όσο γίνεται πιο γρήγορα να υποβάλουμε και συμπληρωματική έκθεση. Το επόμενο έχει να κάνει με την προστασία των δικαιωμάτων ε, του παιδιού. Εκεί πετύχαμε πολύ γιατί διαπιστώσαμε ότι υπάρχουν πολλές και διαφορετικές προτάσεις που πηγαίνουν στο Υπουργείο και σε άλλα σώματα. Χρειάστηκε λοιπόν συνεργασία με ε, κυβερνητικούς, ε, κυβερνητικά σώματα. Μια άλλη μεγάλη μας επιτυχία ήταν η συγχρηματοδότηση. Χρησιμοποιώντας ε, λοιπόν τις δυνατότητες που είχαμε, ε, δουλέψαμε και για τα πολιτιστικά δικαιώματα, για την κοινωνία των πολιτών, Και έτσι, κάθε φορά με τη συνεργασία αυτή μπορούμε να έχουμε έκθεση και από την άλλη πλευρά Άρα έρχονται και εναλλακτικέ εκθέσεις για κάθε υπόθεση που εμείς αναλαμβάνουμε. Έτσι συλλέγουμε όλο και περισσότερη εμπειρία. Αλλά συνεργασία μας χρειάζεται ακόμα με όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε. Άλλος. Παρακαλώ κι εσείς. Σας ευχαριστώ πολύ. Όσον αφορά την οργάνωση συνεδριάσεων, στα πλαίσια της ανατολικής συνεργασίας. Εγώ προτείνω στους συναδέρφους να συζητάμε προηγουμένως ποια είναι τα θέματα τα οποία θα μπορούσαν να μας ενδιαφέρουν και πάνω σε τέτοια θέματα να ανταλλάσσουμε εμπειρίες. Για παράδειγμα, έχω ήδη ετοιμάσει εν ώψη της σημερινής συζήτησης κάποια θέματα τα οποία θα μπορούσαν να είναι ενδιαφέροντα ώστε να έχουμε ανταλλαγή απόψεων. Θα μπορούσα εγώ να σας τα παρουσιάσω από πλευρά της Μολδαβίας και να ακούσουμε μετά και οι άλλοι συνάδελφοι από την Ανατολική Συνεργασία τι εμπειρίες έχουν να μοιραστούν μαζί μας. Μπορούμε επίσης να συντονίσουμε και τις διευθύνσεις μας. Αυτό είναι κάτι που μπορεί πιστεύω να γίνει και άτυπα. Συνεπώς, σε επίσημο επίπεδο μπορούμε να συντονιστούμε και να διορθώσουμε καλύτερα τις ανταλλαγές αυτές πληροφοριών. Μπορούμε να επιλέγουμε δηλαδή κάθε φορά μερικά θέματα τα οποία και να μοιραζόμαστε και να ανταλλάσσουμε μεταξύ μας. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Κέντζα για την έκθεσή του και για τα συμπεράσματα που μας παρουσίασε. Τα συμπεράσματα αυτά είναι ενδιαφέροντα και για μας. Θέλω να επανέλθω λίγο στο θέμα της πίεσης. Πίεση που υπάρχει μεταξύ συνήγορου του πολίτη και Υπουργείο Εσωτερικών, Αστυνομία κλπ. Στα πλαίσια της συνεργασίας μας προσπαθούμε να δείξουμε ότι αυτό που είναι σημαντικό είναι να οργανώνουμε συνεδριάσεις κάθε έξι μήνες, για παράδειγμα στην Πολωνία, με τον επικεφαλής της Εθνικής Αστυνομίας και με το Υπουργείο Εσωτερικών αλλά και με εκπροσώπους και άλλων οργάνων ενδεχομένω. Κατά τις ε, συναντήσεις αυτές εμείς παρουσιάζουμε τα πιο σημαντικά προβλήματα που αντιμετωπίζουμε τους τελευταίους έξι μήνες. Σύμφωνα με τις προσφυγές δηλαδή που μας φτάνουν. Αν η συνάντηση αυτή δεν οδηγήσει σε αποτελέσματα, τότε οργανώνουμε μια δημόσια διαβούλευση. Και εφόσον η δημόσια διαβούλευση δεν αποφέρει καρπούς, τότε κάνουμε εμεί προσφυγή στο Συνταγματικό Δικαστήριο, άρα και εμεί πιέζουμε το Υπουργείο Εσωτερικών ή την αστυνομία προκειμένου να αλλάξουν συμπεριφορά. Θέλω ακόμα να ευχαριστήσω εδώ και τον ε, συνήγορο δικαιωμάτων για τη συνεδρίαση που θα λάβει η χώρα στο Παρίσι. Και τέλος θέλω να αναφερθώ στη σημασία που έχουν οι μη κυβερνητικέ οργανώσεις. Η κριτική που έρχεται από τις οργανώσεις αυτές είναι πολύτιμη για μας διότι μας κάνει να μην επαφιόμαστε στις δάφνες μας, αλλά να συνεχίζουμε τη δουλειά μας. Και πάλι ευχαριστώ πολύ που οργανώσετε αυτή τη συνεδρίαση. Παρακαλώ, κύριο Γκέριν. Σε ευχαριστώ. Δυστυχώ δεν ήμουν εδώ όλη τη διάρκεια τη συνεδρίαση, γιατί ήμουν σε άλλη συνεδρίαση με Αφρικανού εκπροσώπου. Από αυτά που άκουσα όμω για του συνήγορου του πολίτη στι διάφορε χώρε. Ευρωπαϊκής Ένωσης και ανατολικά της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι πολύ ε, ευχάριστα. Αλλά εγώ θέλω να ρωτήσω το εξή. Υπάρχουν δικαιώματα τα οποία δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν. Πριν από μερικά χρόνια, εξηγώ ότι εννοώ, υπήρξε ένα σκάνδαλο σε σχέση με την μεταφορά και παράνομη κράτηση ε, φυλακισμένων που τους μετέφεραν πάνω από την Ευρώπη για να τους πάνε τελικά στο Γουαντάναμο. Το Συμβούλιο της Ευρώπης με πολύ θάρρος, τόλμη και ξεκάθαρο πνεύμα χάρη σε έναν ελβετό εισηγητή διευκρίνησε κάπως την κατάσταση. Διαβάζοντας εγώ την έκθεση αυτή καταλαβαίνω ότι έχουμε να κάνουμε με την εφαρμογή από διάφορες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και χωρών μη μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε σχέση με την υποχρέωσή τους να σέβονται τα ανθρώπινα δικαιώματα. Πιστεύω ότι είναι τροπή. Λοιπόν, οι συνήγοροι του πολίτη που βρίσκονται εδώ τα ξέραν αυτά, ήταν εν γνώση τους. Και εφόσον υπάρχουν τέτοιες περιπτώσεις σε βάρος των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, παραβίας ανθρωπίνων δικαιωμάτων, τα λένε ή τελικά οι διάφοροι οργανισμοί αυτοί που πρέπει να παρακολουθούν την τήρηση ή μη των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ε, ερμηνεύουν διαφορετικά τα πράγματα. Έχουμε την Επιτροπή Monitoring του Συμβουλίου της Ευρώπης για τις υποχρεώσεις των κρατών μελών. Εδώ διαφορετικά βλέπουν οι οργανισμοί αυτοί, ή άλλοι του, της ΟΑΣΕ, βλέπουν διαφορετικά τη σύμβαση της ε, Βενετίας. Αν ναι, τότε έχουμε πρόβλημα. Γιατί όλες οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως και όλες οι χώρες του Συμβουλίου της Ευρώπης, θα έπρεπε με τον ίδιο τρόπο να τηρούν τη σύμβαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Οπότε δεν με ικανοποίησαν όλα αυτά που άκουσα πλήρως. Ευχαριστώ. Η Μπαρμπαρα Κύριε Γκέρεντς, Θα ήθελα να σας απαντήσω, γιατί νομίζω ότι κατά την προετοιμασία δεν ζητήσαμε από τα Ινστιτούτια Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων να απαντήσουν στο συγκεκριμένο ζήτημα. Να σας ενημερώσω λοιπόν, νομίζω ότι στην τελευταία συνεδρίαση πριν από τις καλοκαιρινές διακοπές είχαμε πάλι το ΔΙΚ Μάρτι στο Στρασβούργο, αν δεν κάνω λάθος, και εξήγησε πολύ σύντομα ότι πολλέ από τις συστάσεις τους δεν τις ακολούθησαν ούτε τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, ούτε οι μέλη, ούτε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Και εδώ νομίζω ότι δικαίω η Επιτροπή ΛΥΜΠΕ αποφάσισε να κάνει μια έκθεση παρακολούθησης, διότι αφενός έχουμε την έλλειψη παρακολούθηση τη έκθεση ΦΑΒΑ που είχαμε στην προηγούμενη θητεία και στην Επιτροπή μα εμεί θα έχουμε μια γνωμοδότηση βάσει του άρθρου 50 για να μπορέσουμε να παρουσιάσουμε τα αιτήματά μας και να τα δώσουμε στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων βάσει και της διαδικασίας. Εντάξει, μπορεί να μην αποτέλεσε το στόχο της συνεδρίας αυτό. Αλλά ε, δεν μπορούμε να κρίνουμε τον υπόλοιπο κόσμο χωρίς να είμαστε άψογοι Πρέπει να είμαστε απολύτως άμεμπτοι όταν πάμε να δώσουμε μαθήματα στον υπόλοιπο κόσμο. Για μένα εξακολουθεί να αποτελεί έσχος, ακόμα χειρότερα. Απαραβιάσει ανθρωπίνων δικαιωμάτων με συνενοχή των κεντρικών αρχών που υποτίθεται, και δεν μιλώ για τους συνηγόρους του πολίτη, αλλά των κυβερνήσεών μας, που υποτίθεται ότι προστατεύουν και οι οποίες παρέμειναν σιωπηλέ σε όλες τις επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εάν δεν φωτιστεί η κατάσταση αυτή, νομίζω ότι... Διακόπτε μικρόφωνο ο κ. Κιόρενς. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Κέντζα. Τέθηκε το ερώτημα της γενικότερης αξιολόγησης των οργανισμών αυτών και το ανέφερα και στην εισαγωγή μου υπάρχει αυτή η ταξινόμηση ε, γ της κατάστασης του κάθε οργανισμού. Αν θέλετε επιπλέον πληροφορίες, να σας πω ότι η κατάσταση έχει ως εξής αυτή τη στιγμή. Πρόκειται για μια διαδικασία πιστοποίησης βάσει της Επιτροπής Διεθνούς Συντονισμού που γίνεται από την Υποεπιτροπή Πιστοποίησης και κάθε οργανισμός ανθρωπίνων δικαιωμάτων που έχει κάνει αίτηση για πιστοποίηση για πρώτη φορά, μετά από πέντε χρόνια πρέπει να επανεξετάζεται, γίνεται μια αξιολόγηση ε, για την ανανέωση της πιστοποίησης. Και προς το παρόν, οι χώρες ε, της Ανατολικής Συνεργασίας εντάσσονται ως εξής. Τέσσερις χώρες βρίσκονται στην κατηγορία Α, υπάρχει ένα πρόβλημα ε, με το Ινστιτούτο του Αζερβαϊτζάν γιατί η υποεπιτροπή ε, πιστοποίησης πρότεινε νομίζω το περασμένο φθινόπωρο να υποβαθμιστεί στην κατηγορία Β αλλά ο Αζέρος ε, συνήγορος του πολίτη είχε αντιρρήσεις και αυτή τη στιγμή είναι υπό εξέταση το ζήτημα νομίζω ότι θα ολοκληρωθεί σύντομα και το Ινστιτούτο της Μολδαβίας βρίσκεται στην κατηγορία Β. Αυτά έχουμε προς το παρόν. Οι άλλες τρεις χώρες, η Ουκρανία, η Αρμενία και η Γεωργία βρίσκονται στην κατηγορία Α. Ευχαριστώ. Η κυρία Σουλεϊμάνοβα, ε, Είναι πολύ ενδιαφέρουσα η ερώτηση. Εμείς είμαστε οργανισμοί οι οποίοι είμαστε αναγνωρισμένοι από πολλούς ε, διεθνούς οργανισμούς. Υπάρχει το εξή πολύ ενδιαφέρον. Λάβαμε τρεις φορείς ε, ερωτήσεις, κάθε φορά απαντήσαμε και κάθε φορά μας ξαναέθεσαν ερώτηση και πάντα λάβαμε την απάντηση ότι δεν είναι ικανοποιημένοι. Ήμουνα σε μια συνεδρίαση του ΣΚΑ και του ζήτησα να μου στείλουν κατεπηγόντως οποιονδήποτε ειδικό εμπειρογνώμονα έχουν και η απάντηση ήταν θα μας αποστείλουν ένα μέλος του ICC από τη Γαλλία εντός κάποιων ημερών. Είμαστε πολύ ανοιχτοί, είναι διάφανη διαδικασία, μπορείτε να αναλύσετε τα αποτελέσματά μας. Ε, και κάποιες φορές βρέθηκα ενώπιον των 50 χωρών, των εκπροσώπων των χωρών και τους ζήτησα ποια είναι η άποψή σας, γιατί αποφασίσατε να μας υποβαθμίσετε. Δεν έλαβα καμία απάντηση και ελπίζω σύντομα μετά από την αναθεώρηση θα λάβουμε και τα αποτελέσματα, διότι το βλέπουμε σε κάποιους διεθνείς οργανισμούς η πολιτική ε, βούληση, το πολιτικό της συμφέρον όχι μόνο παρισφρεί στα ανθρώπινα δικαιώματα αλλά παρεμβαίνει κιόλα. Το είπα λοιπόν, μπορείτε να έρθετε να μας ερευνήσετε. Ήρθαν και άλλοι δύο-τρεις εμπειρογνώμονες, δεν υπήρχε κανένα πρόβλημα, καμία παραβίαση βασικών αρχών. Ευχαριστώ πολύ. Υπάρχει μία ακόμα αίτηση από την κυρία Λικόβιτς. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Ευρωβουλευτή για την παρέμβασή του, αλλά δεν ε, εξετάσαμε εμείς το θέμα αυτό. Έγιναν καταγγελίες και για την Πολωνία και ασχολείται η Πολωνική Εισαγγελία με το θέμα αυτό. Όσον αφορά τώρα τα πρακτικά των διαδικασιών. Εγώ όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία θα μπορέσω να διαβάσω τα πρακτικά. Δεν είχα πρόσβαση ε, στο παρελθόν, αλλά μόλις μου δοθεί το νομικό δικαίωμα να τα εξετάσω θα κάνω και τον έλεγχο. Θα ήθελα όμως να διαμαρτυρηθώ εδώ. Δεν θέλουμε εμείς να διδάξουμε τίποτα σε κανέναν. Η ανατολική συνεργασία δεν προβλέπει διδαχές εμείς είμαστε απλώς περήφανοι διότι έχουμε καταλήξει σε κάποιες ευρωπαϊκές λύσεις που είναι χρήσιμες, αλλά προβλέπουμε να γίνει ανταλλαγή απόψεων. Δεν θα θέλαμε να χρησιμοποιείτε λοιπόν τέτοια, ε, τέτοιο λεξιλόγιο, δεν προσπαθούμε να διδάξουμε τίποτα σε κανέναν. Η παρατήρησή σας μου επιτρέπει να άρω μια παρεξήγηση. Εγώ μιλάω για μας, για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, δεν μιλάω για σας. Έχω κάθε σεβασμό για το έργο σας η ανησυχία μου είναι να συνεισφέρουμε ώστε να μην υπάρχουν διεξοδοί ούτε λήψει όσον αφορά την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Εσείς έχετε ένα ιδιαίτερα ευγενές έργο, το αναλαμβάνετε με ιδιαίτερη αξιοπρέπεια, αντιλαμβάνομαι τις δυσκολίες. Για όλους μας όμως προέχει να μην υπάρχουν τρόποι να ξεφύγει κανείς όταν πρόκειται για το σεβασμό ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Πρόεδρος, ευχαριστούμε πολύ. Κυρίε και κύριοι, ε, αντιλαμβάνομαι ότι υπάρχουν πολλά ακόμα θέματα που θα μπορούσαμε να συζητήσουμε. Πρέπει όμως να ολοκληρώσουμε αυτή τη ε, συζήτηση και να σας ευχαριστήσω όλους που ήρθατε και συμμετείχατε στην τόσο ενδιαφέρουσα αυτή συζήτηση. Σας ευχαριστώ επίσης που παρουσιάζετε και τους πρώτους καρπούς της συνεργασίας αυτής. Όπως είπε ο καθηγητής Κέντσα, υπάρχουν επιτυχίες και υπάρχει και εμπειρία που έχουμε συλλέξει και είναι πολύ θετική για τη συνεργασία μεταξύ μας στο μέλλον. Η συνεργασία αυτή ελπίζω να συνεχιστεί. Τόσα ακούσαμε εδώ ήταν πολύ ενδιαφέροντα. Πρόκειται για μια ανταλλαγή, ανταλλαγή εμπεριών. Έχουμε να μάθουμε με ένα από τους δε. Πράγματι, οι χώρες που πέρασαν από μεταβατικές περιόδους ε, χρειάστηκε να λύσουν προβλήματα που τέθηκαν σε αυτές. Οπότε, την εμπειρία σας αυτή θέλουμε να τη μοιραστούμε μαζί σας. Ευχαριστώ επίσης και όσους συμμετείχαν στην πρωτοβουλία αυτή, δηλαδή ε, την Πολωνία και τη Γαλλία και κάθε επιτυχία ε, στη συνέχεια του έργου σας. Ευχαριστώ πολύ για την Αρμενία, το Αζερμπαϊτζάν, τη Γεωργία και τη Μολδαβία για την παρουσία τους εδώ σήμερα. Κύριε Κένσια, σας ευχαριστώ και σας πολύ για την δουλειά που μας παρουσιάσατε και για τα συμπεράσματα τα οποία θα μας βοηθήσουν εμάς στο έργο μας στη συνέχεια. Τελειώνουμε αυτό το σημείο στην ημερήσια διάταξη και περνάμε στο επόμενο σημείο της ημερήσιας διάταξης. Λέει Πρόεδρος. Στην ημερήσια διάταξη έχουμε τώρα ανταλλαγή απόψεων για τις εξελίξεις στην Ιεμένη. Και είμαστε πολύ τυχεροί που μπορούμε τηλεφωνικά να συνδεθούμε με κάποιον που δραστηριοποιείται στα ανθρώπινα δικαιώματα στην Ιεμένη. Είμαστε σε τηλεφωνική επαφή λοιπόν μαζί του και έχουμε εδώ και εκπροσώπους από την Υπηρεσία την Ευρωπαϊκή Εξωτερικής Δράσης. Οπότε εσείς μπορείτε να μείνετε άμα θέλετε, αλλά ησύχω γιατί καταλαβαίνετε ότι τεχνικά είναι δύσκολη η επικοινωνία ή να βγείτε από την αίθουσα εφόσον θέλετε να αναχωρήσετε. Πρόκειται για την κυρία Μπάσα. Κυρία Μπάσα, μας ακούτε? E- hi, good,